So, ladies and gentlemen. Κυρίες και κύριοι αγαπητοί συνάδελφοι, καλώς ήρθατε όλες και όλοι. 9 και 3 λεπτά είναι η ώρα, οπότε μπορούμε να ξεκινήσουμε. Everybody got an uh, agenda. Έχετε όλη τη μέρη σχεδιάταξη για σήμερα. Υπάρχουν προτάσεις τροποποίησης. Όχι από ό,τι φαίνεται, επομένω εγκρίνεται. Σημείο 2. Έγκριση των πρακτικών. Έχετε τα σχέδια των πρακτικών στους φακέλους σας. Αν δεν υπάρχει αντίρρηση στη διάρκεια της ε, συνεδρίασης, θεωρούνται εγκεκριμένα. Σημείο 3. Έχετε στους φακέλους σας και τις αποφάσεις ε, της συνεδρίασης της 11ης Οκτωβρίου, της συνεδρίασης των συντονιστών και αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις ούτε και για αυτή τη συνάντηση θεωρούμε ότι εγκρίνονται τα πρακτικά της συνεδρίασης των συντονιστών και περνάμε στο σημείο 4 ανακοινώσεις του Προέδρου. Ως ήθιστε μεταδίδεται στο διαδίκτυο η σημερινή μας συνεδρίαση Να είμαστε λοιπόν κόσμοι και να μιλάμε και σχετικά αργά. Θα ήθελα επίσης να προσκαλέσω, να συγγνώμη, ευχαριστήσω τους ε, προσκεκλημένους από Λισαβόνα, Ελσίνκη, τα Ορμίνα που είναι εδώ και να τους καλωσορίσω. Επίσης θα σας πω ότι 31 Οκτωβρίου και 1 Νοεμβρίου έλαβε χώρα η τρίτη συνάντηση της κοινή ε, μεικτής κοινοβουλευτική Επιτροπής Καριφόρουμ Ευρωπαϊκή Ένωση, στο Τριντάθ και τον Πάγκο. Είναι κάτι το οποίο είχαμε ε, πιέσει. Η συμφωνία με το Κάριφόρουμ έχει τεθεί σε ισχύ εδώ και λίγα χρόνια. Προχωρούμε σιγά σιγά. Υπάρχουν βέβαια κάποια ζητήματα τα οποία χρήζουν συζήτηση. Ε, επηρεάζουν, αλλά όχι και πολύ, αλλά τέλο πάντων επηρεάζουν τι οικονομικέ εξελίξει. Υπάρχει το θέμα επίση τη συμμετοχή κοινωνία των πολιτών και το καθεξή, αλλά τις εκθέσεις, την έκθεση μάλλον θα τη συζητήσουμε στην επόμενη μας συνεδρίαση. Σημείο 5. Μια σύντομη παρουσίαση της επίσκεψής μας την προηγούμενη εβδομάδα Ζηλανδία και Αυστραλία. Αλλαγές και νέα κυβέρνηση, ενδιαφέρουσες εξελίξεις. Δεν ξέρω ακριβώ και για τον νέο Υπουργό Εμπορίου σε τι κατάσταση βρισκόταν, δεν τα είχε ακόμη τα πράγματα ξεκαθαρίσει. Υπάρχει το ζήτημα στην πισπικότητα, στη Γερουσία και τέλος πάντων ήταν ταραγμένα τα νερά και στη Βουλή και στη Γερουσία. Παρ' όλα αυτά, promote our resolution. You we είχαμε εγκρίνω όπως ξέρετε και αυτό το ψήσιμο την προηγούμενη εβδομάδα στο τεφατέο σχέδιο εντολή για την Αυστραλία Νέα Ζηλανδία. Και μιλήσαμε και με τους επιβαλείς πραγματευτές και τις ομάδες, τους βασικούς ουλευτές και εκπροσωπήθηκαν επίσης πολλοί άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς και από την κοινωνία των πολιτών. ήταν σαφέστατο ότι τους ενδιαφέρει όλους να υπάρξει στενότερη συνεργασία. Και ε, τέθησαν βέβαια και κάποια ζητήματα ό,τι αφορά κάποιους δασμούς, γεωργικούς ή το θέμα το 10% για την Αυστραλία για τους ελληνικούς δασμούς ε, και για τα αυτοκίνητα και το 33% των ε, φόρων που επιβάλλονται σε κάποια οχήματα. Δηλαδή, το αυτό το ζήτημα των διαπραγματεύσεων. Αλλά είμαι ότι μπορούμε να συμβιβαστούμε. Συζητήσαμε επίση ε, με τα συνδικάτα στην Αυστραλία. Υπάρχει το θέμα της, ε, του σεβασμού των εργασιακών δικαιωμάτων. Στην Ζηλανδία Εδώ από τα πρότυπα του Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας δεν έχουν επικυρωθεί. Ζητήθηκε λοιπόν το θέμα της επιβολής η περιβαλλοντική, μάλλον η προστασία των επενδύσεων είναι ένα θέμα που συζητήθηκε επίση. Δεν είναι ικανοποιημένη στην Νέα Ζηλανδία και την Αυστραλία με το παλιό σύστημα το ISDS. Άρα αυτό είναι ένα καλό δείγμα ότι υπάρχει νέα όθηση σε ό,τι αφορά την προστασία των επενδύσεων. Και αυτό που κάπως με εξέπληξε ήταν το τρίτο σημείο που σχολίασαν τα συνδικάτα. για κάποια ζητήματα που αφορούσαν ε, μετανάστες ε, και εργαζόμενους από τρίτες χώρες. Σε κάποιες συμφωνίες. Η επίσκεψή μας, ιδίως γιατί υπήρχε κάποια καθυστέρηση σε αυτή την επίσκεψη τη Επιτρόπου Μάλστρομ στι χώρε αυτέ. Άρα, εμεί δώσαμε ένα καλό μήνυμα. Πιστεύω ότι είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε διαπραγματεύσει. Για να έχουμε μια δίκαιη και καλή εμπορική συμφωνία. Δεν ξέρω αν κάποιοι θέλουν να προσθέσουν κάτι από όσους ήταν μαζί. Κάρολα, ίσως. Σε ευχαριστώ. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω για μια ακόμη φορά τη Γραμματεία για την πολύ καλή οργάνωση της ε, αποστολής αυτής τη αντιπροσωπείας και εγώ θεώρησα ότι ήταν πολύ καλή αυτή η επίσκεψη, πολύ επίκαιρη για την Αυστραλία και την Ισλανδία. Ε, ήταν φορτωμένο το πρόγραμμα, σχεδόν τρέχαμε από το ένα μέρος στο άλλο για να το συναντήσουμε όλους. Ε, ήταν πολύ ενδιαφέρον, παρατηρήσαμε επίσης ε, ότι άξιζε ε, η μετακίνησή μας εκεί. Μιλήσαμε με τα συνδικάτα, όπως είπες, αλλά και με υπουργού και νομίζω ότι ήταν πολύ σημαντικό που είχαμε ήδη εγκρίνει εκ των προτέρων το ψήφισμα που ανέφερες και εσύ, γιατί ήταν ένα σημείο συζήτηση και μπορούσαμε έτσι να ε, αναφέρουμε κάποια θέματα. Αυτό το οποίο παρατήρησα είναι ότι Φαίνεται ότι για τις διαπραγματεύσεις αυτές αυτές υπάρχει ενθουσιασμός. Όλοι θέλουν να υπάρχει αυτή η συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θεωρούν ότι θα έχει προσθέμενη αξία κάτι τέτοιο. Και από πολλές πλευρές επίσης έγινε αναφορά ε, στην ανάγκη να είναι ρεαλιστικές οι διαπραγματεύσεις αυτές. Υπάρχουν ε, κάποιοι βέβαια ευαίσθητοι τομείς, λίγοι όμως, Τώρα, σε ό,τι αφορά τη διαπραγματευτική εντολή, το ότι μόνο Φεβρουάριο ή Μάρτιο θα εγκριθεί και θα συνεχίσουν μετά οι διαπραγματεύσει, αυτό δεν ήταν και τόσο θετικό. Υπήρξε κάποια απογοήτευση, γιατί θα ήθελα να ξεκινήσουν ίσω από φέτο ε, οι διαπραγματεύσει για να υπάρχει μια γρήγορη εξέλιξη. Εμείς βέβαια τους είπαμε ότι δεν μπορούν να γίνουν διαπραγματεύσεις μέσα σε ένα-δυο μήνες και ήδη ο στόχος του 2019 είναι αρκετά φιλόδοξος. Επιμείναμε όμως ότι το θέμα είναι η ποιότητα, όχι ταχύτητα. Και παρόλα αυτά πιστεύουμε ότι θα έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα όταν ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις. Πολύ καλό ταξίδι, ευχαριστώ. Εγώ πραγματικά ε, πήρα πολλά μαζί μου, γνώρισα πολλούς ενδιαφέροντες ανθρώπους, ε, έκανα πολύ ενδιαφέρουσες συζητήσεις. Ευχαριστώ για μια ακόμη φορά. Ευχαριστώ. No cóż, e, e, e, trzeba powiedzieć szczerze, że był bardzo budujący. Ευχαριστώ. Αυτό που μπορώ να πω ήταν ότι πραγματικά ε, και ήταν ε, πάρα πολύ καλή οργάνωση αλλά και γιατί κάναμε συναντήσεις ε, στην Αυστραλία και ε, στη Νέα Ζηλανδία και είδαμε πραγματικά ένα ευρύ φάσμα εκπροσώπων διαφόρων θεσμών που ενδιαφέρονται άμεσα για τις συμφωνίες αυτές. Όχι δηλαδή μόνο εκπροσώπους της κυβέρνησης ε, και της Βουλής, αλλά και εργοδότες, εργαζομένους, ε, συνδικάτα ε, και μειονότητες επίσης που έχουν τα δικά τους προβλήματα στη Νέα Ζηλανδία. Μπορεί στην Αυστραλία να μην είναι τόσο μάλλον να είναι λιγότερο οξυμένο το πρόβλημα από τις Αυστραλία. που υπάρχουν και εκεί προβλήματα και συζητήσαμε να δούμε και τι ευκαιρίες μπορούν να αναδυθούν με την υπογραφή μια συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκή ε, Ένωση και Νέα Ζηλανδία. Για μένα πραγματικά ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η επίσκεψη. Άκουσα τις απόψεις των μειονοτήτων με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στην Ζηλανδία που φαίνεται ότι έχουν και πολλές οικονομικές ελπίδες και προσδοκίες από την ε, οικονομίας ό,τι αφορά τους διάφορους τομείς και κλάδους της οικονομίας. Έπειτα, σε σχέση με την Αυστραλία, βλέπουμε κάποια ε, κοινωνικές εξελίξεις ή τέλος πάντων η κοινωνία έχει απαιτήσει και προσδοκίες. Ποιες τώρα είναι οι προοπτικές είπε και ο πρόεδρος, είπε και η προλαλήσασα, ότι ναι, πράγματι ε, θα μπορούσαμε να επιταχύνουμε κάπως τα πράγματα και να υπογράψουμε νωρίτερα, αλλά δεν, ε, δεν μπορούμε να βιαστούμε τόσο πολύ. Είναι δύο κράτη αυτά βέβαια τα οποία έχουν πολύ στενούς δεσμούς, πολιτιστικούς, θρησκευτικού κτλ. Μας ενώνουν πολλά ε, σε ό,τι αφορά την παγκόσμια θεώρηση, την εμπορική θεώρηση του πράγματο κτλ. Και μπορούμε, πιστεύω, να προχωρήσουμε γρήγορα, γιατί αυτά που μας ενώνουν είναι πολύ περισσότερο από αυτά που μας χωρίζουν. Οι συνομιλίε με τον Καναδά, για να σας δώσω ένα άλλο παράδειγμα, επίσης ε, ε, ήταν αντίστοιχου χαρακτήρα, γιατί και οι Καναδοί μοιάζουν πολύ με εμά σε πολλά τώρα. Υπάρχουν κάποια εμπόδια ίσως ε, που πρέπει να ξεπεράσουμε, αλλά νομίζω ότι μπορούμε πολύ γρήγορα να ολοκληρώσουμε τις διαπραγματεύσεις. Η σκέψη μας λοιπόν ε, ήταν πάρα πολύ χρήσιμη και νομίζω ότι δημιούργησε ένα καλό κλίμα τελικά σε διάφορα επίπεδα. Ευχαριστώ. And uh, now I will give the floor to David. Και τώρα θα δώσω το λόγο στον David. <laughs> Thank you, Mr. Chairman. Congratulations getting my full name Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και συγχαρητήρια που είπατε το όνομά μου ολόκληρο. Ήταν πράγματι πολύ ενδιαφέρουσα η συνάντηση. Εγώ παρέμεινα ε, όταν η υπόλοιπη αντιπροσωπεία πήγε στην Αυστραλία. Δεν σας ακολούθησε στην Αυστραλία. Ήταν όμως πολύ ενδιαφέρουσα η συνάντηση που είχαμε με τον Μακλέη, τον Υπουργό ε, μετά την αναχώρησή σας. Και ήμασταν η πρώτη αντιπροσωπή από το εξωτερικό που συναντήθηκε με τη νέα κυβέρνηση της Νέας Ζηλανδίας και ιδιαίτερα τον Υπουργό Εμπορίου και Εξωτερικών. Συναντήθηκα επίσης με εκπροσώπους αγροτών, με κτηνοτρόφους του γαλακτικού τομέα, άκουσε τα προβλήματά τους. Ορισμένοι από αυτούς ε, ανησυχούν μάλλον για την πιθανότητα να επισέλθουν προστατευτικά μέτρα ή ακόμα και κυρώσεις. Το Γενικό Προμηθευτικό καθεστώ. Επίση ήταν ένα ζήτημα που μας αποσχόλησε και το συζητήσαμε. Και το γεγονό ότι δεν υπάρχει ένα κεφάλαιο για τις επενδύσεις τελικά ε, φαίνεται να το καλοδέχτηκαν. Να, να είτε. Υπάρχει επίσης ένα ζήτημα σε σχέση με την συμπληρωματικότητα για αυτούς είναι σημαντικό. Και εξαιτία του γεγονότο, μια και βρίσκονται στο νότιο ημισφαίριο, η περίοδο ε, για τι ε, σοδιές, η περίοδο για, για το άρπαγμα, για όλα αυτά, για την παραγωγή των προϊόντων του είναι διαφορετική από αυτή που έχουμε στην Ευρώπη ενάντια στις συμφωνίες υπήρχε μια κάποια αντίσταση από κάποιους παραγωγούς, αλλά γενικά μιλώντας, οι περισσότεροι κλάδοι την έχουν υποδεχτεί θετικά. Και θα έλεγα ότι η επίσκεψη μας εκεί και οι συζητήσεις που είχαμε εκεί ήταν χρήσιμες. Πράγματι, έτσι πιστεύω και εγώ ότι ήταν ε, αποτελεσματική και χρήσιμη η επίσκεψή μας και στη Νέα και στην Αυστραλία. Είναι απαραίτητο για την Ευρωπαϊκή Ένωση να προσπαθήσει να ενισχύσει τον σεβασμό των κανόνων στο διεθνές εμπόριο, ιδιαίτερα σε μια εποχή που παραδοσιακοί μας εταίροι, άλλες χώρες έχουν ε, κινηθεί προς την κατεύθυνση του δικαίου του ισχυρού. Θα ήθελα πάλι να ευχαριστήσω τη Γραμματεία για την οργάνωση της ε, επίσκεψης και βεβαίως δεν πρέπει να ξεχνά κανεί ότι τέτοιου τύπου επισκέψει είναι περίπλοκε, γιατί υπάρχουν πολλέ συναντήσει που η μία ακολουθεί την άλλη και πρέπει όλε να γίνονται ε, στην ώρα του. Ωραία. Αυτή ήταν η πρώτη ενημέρωση για την επισκέψή μα. Έχουμε 20 λεπτά τώρα στη διάθεσή μα, δηλαδή δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε μια πλήρη συζήτηση, απλώ μια ενημέρωση θα θέλαμε να ακούσουμε από την πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ίσω να του. Ε, ε, θέσουμε και κάποιες ερωτήσεις. Θα επανέλθουμε στο θέμα, γιατί αυτό που θα κάνουμε σήμερα είναι κάπως καινούριο. Είναι κάτι το οποίο το ζητούσαμε εδώ και καιρό. Γιατί πάντοτε επιθυμούμε να παρακολουθούμε την πρόοδο των διαπραγματεύσεων και να ε, εκφράζουμε τις απόψεις μας στην Επιτροπή που τις διεξάγει αυτές τις διαπραγματεύσεις, δεδομένου ότι και στο τέλος οποιαδήποτε συμφωνία πρέπει να εγκριθεί από το Κοινοβούλιο. Καλύτερα όμως είναι ε, αυτές οι συζητήσεις να γίνονται κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων και να σκεφτόμαστε, να, μάλλον να, να, το να εξετάζουμε πώς τελικά εφαρμόζονται οι εμπορικές συμφωνίες μας βοηθά να διαμορφώνουμε τις απόψεις μας και για την διαπραγμάτευση τέτοιων συμφωνιών. Σήμερα λοιπόν θα ακούσουμε την παρουσίαση της Επιτροπής όπου... η οποία προετοίμασε μια αξιολόγηση του πώς έχουν εφαρμοστεί οι διάφορες συμφωνίες ελευθέρου εμπορίου Είναι η πρώτη φορά λοιπόν που έρχεται η Επιτροπή να μας κάνει μια τέτοιου τύπου παρουσίαση. Πρώτη φορά σήμερα λοιπόν θα συζητήσουμε αυτό το θέμα. Θα υποβάλουμε κάποια ερωτήματα. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα το ξανασυζητήσουμε. Και θα δώσω το λόγο στον κύριο Κάρτερ, αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή τη Γενικής Διεύθυνσης Εμπορίου, DigiTrade. Καλημέρα Ευχαριστώ κύριε Λάγκε για την εισαγωγή, για το καλωσόρισμα. Με βοηθάτε επίσης γιατί θέσατε το πλαίσιο ε, μέσα στο οποίο η Επιτροπή ήρθε να σας παρουσιάσει αυτό το νέο είδος έκθεσης, μια έκθεση που εξετάζει την εφαρμογή των διαφόρων συνθήκων ελευθερού εμπορίου. Όπως είπατε, η Επιτροπή διαπραγματεύεται νέες ε, συμφωνίες ελευθερών εμπορίου, αλλά τα παράλληλα φροντίζει και την εφαρμογή των υφιστάμενων, τα αμυντικά μέτρα ε, και ίσως αυτό το έργο της Επιτροπής, η εφαρμογή των υφιστάμενων συνθήκων δηλαδή, να μην σε αυτό να μην δίνεται το, η απαιτούμενη προσοχή. Ε, προετοιμάσαμε λοιπόν αυτή την έκθεση είναι ε, απαραίτητο να σας δίνουμε αυτές τις πληροφορίες και για λόγους διαφάνειας, αλλά επίσης και για να ε, εντοπίσουμε τα προβλήματα που υπάρχουν ε, στοιχεία που μας απογοητεύουν, που μας προβληματίζουν είτε από τη δική μας την πλευρά είτε από την πλευρά των εμπορικών μας εταίρων. Και γενικότερα για να έχει κανείς μια, εικόνα του, των εξελίξεων στον τομέα του διεθνούς εμπορίου και της βιώσιμης ανάπτυξης. Όλα αυτά τα στοιχεία λοιπόν μπορεί να τα βρει κανείς σε αυτή τη νέα έκθεση. Τώρα, ε, ε, έχω το εξή πρόβλημα. Ε, Δυστυχώ δεν μπορώ να σα την παρουσιάσω γιατί δεν έχει εγκρόμα εγκριθεί από τη, το, το Κολόγιο των Επιτρόπων, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επομένω, θα σας παρουσιάσω αυτό που θα πρόκειται να εγκριθεί και σας διαβεβαιώνω ότι θα σας την αποστείλουμε ε, κατά τη διάρκεια της ημέρας, γιατί η έγκρισή της θα γίνει σήμερα. Και πάλι σας ζητώ συγγνώμη για αυτό. Θα ήταν πολύ καλύτερα να την είχα στα χέρια μου. Έχει δύο στόχους η έκθεση. Όπως σας είπα, είναι ένα σημαντικό εργαλείο για την βελτίωση της διαφάνειας και έναντι ε, ημών και έναντι των κρατών μελών και οποιοδήποτε άλλο ενδιαφερόμενο μέρους. Γιατί ώστε όλοι αυτοί οι ενδιαφερόμενοι να γνωρίζουν τι κάνουμε στον τομέα του διεθνούς εμπορίου. Το δεύτερο στοιχείο που είναι πολύ σημαντικό είναι ότι θα είναι ετήσια αυτή η έκθεση. Φέτος είναι η πρώτη χρονιά, αλλά σκοπεύουμε να παράγουμε τέτοιε εκθέσει κάθε χρόνο θα αξιοποιήσουμε και την υποδοχή που θα επιφυλάξετε εσείς στην έκθεση αυτή και οι άλλοι εταίροι μας για το πώς θα τη δούνε για να την βελτιώσουμε τις επόμενες χρονιές. Και νομίζω ότι θα μπορούμε να αξιοποιούμε και φέτος και κάθε χρόνο τη δημοσίευση, τη στιγμή της έγκρισης αυτής της έκθεσης και τη δημοσίευσή της για να συζητούμε τα θέματα αυτά. Μέχρι σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, παρουσίαζε εκθέσεις υλοποίησης για τρία, τρεις ε, συμφωνίες ελευθερού εμπορίου, την Κορέα, την Κεντρική Αμερική ε, και, στην Κεντρική Αμερική, μάλλον στην Κολομβία και το Περού. Για αυτές τις τρεις ε, συμφωνίες υπήρχε η νομική υποχρέωση να το πράττουμε αυτό. Σήμερα η έκθεση που σας παρουσιάζω ε, εξετάζει την υλοποίηση 22 εμπορικών συμφωνιών επιπλέον. Άρα 22 συν 3, 25. το ερώτημα είναι, ε, έχουμε καλύψει όλε. Όχι. Ε, συνολικά ε, είναι πάνω κάτω 40 οι συμφωνίε ελευθέρου εμπορίου που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι 15 που λείπουν είναι αυτές που δεν είχαμε τη δυνατότητα να εξιολογήσουμε σε αυτό το χρονικό στάδιο, γιατί πρόκειται για χώρες ίσως πολύ μικρές, όπως η Ονδόρα, το Μαυροβούνιο, το Κωσυφοπαίδιο, ε, για τις οποίες δεν έχουμε ακόμα, για την υλοποίηση αυτών των συμφωνίων δεν έχουμε ακόμα αρκετά στοιχεία, πάντως θα τις καλύψουμε την επόμενη χρονιά. Υπάρχει ένα έγγραφο εργασία του προσωπικού τη Επιτροπή που είναι πάνω από 140 σελίδε, που είναι πολύ αναλυτικό. Αν θέλετε οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία θα τη βρείτε εκεί. Για κάθε μια λοιπόν από τις 25 συμφωνίες ελευθερών πορείου υπάρχουν αναλυτικά στοιχεία και ε, για πρώτη φορά εξάγουμε και κάποια γενική φύσεων συμπεράσματα που ισχύουν για όλες τις συμφωνίες. Το πρώτο που μας απασχολεί είναι πώς τελικά εφαρμόζονται οι προβλέψεις για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Το δεύτερο είναι μια εκ των υστέρων αξιολόγηση της κάθε μιας ε, συμφωνίας. Και επίση υπάρχει και μια, μια ενότητα της έκθεσης η οποία αναφέρεται στις δραστηριότητες και στο εσωτερικό της Επιτροπής και έναντι τρίτων ε, που έχουμε αναλάβει για την σύναψη νέων τέτοιων συμφωνιών. Τέσσερις ομάδες, σε τέσσερις ομάδες θα μπορούσαμε να ομαδοποιήσουμε ε, τις ε, συμφωνίες αυτές. Η πρώτη ομάδα θα ήταν το Μεξικό, η Χιλή, οι χώρες της Μεσογείου, η Τουρκία. Ήταν η πρώτη γενιά, οι οποίες ήταν περιορισμένου είχαν ένα περιορισμένο εύρος εφαρμογή. Η δεύτερη γενιά είναι οι λεγόμενες ε, συνολικές deep and comprehensive. Ε, αυτές ε, τέτοιου τύπου συμφωνία έχουμε για παράδειγμα με τη Γεωργία. Μια τρίτη ομάδα είναι οι συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης, EPA, και η τέταρτη ομάδα είναι οι πιο πρόσφατες, οι συμφωνίες ελευθέρων εμπορίου νέας γενιάς όπως λέμε, με την Κορέα, με την Κολομβία, με το Περού και στο μέλλον με το Βιετνά, με την Ιαπωνία, οι οποίες αναμένουμε, ελπίζουμε ότι θα εγκριθούν. αυτές οι τελευταίες προφανώς ε, δεν καλύπτονται στην φετινή έκθεση, θα καλυφθούν στην έκθεση της επόμενης χρονιάς. Το θετικό στην έκθεση αυτή είναι ότι επίσης υπάρχει και μια επεξήγηση όλων των διαφορών μεταξύ των εμπορικών συμφωνιών και αξιολογούμε κάθε μια από τις συμφωνίες με βάση πέντε δείκτες. Πρώτα απ' όλα τις ροές, τις εμπορικές με τις χώρες αυτές, πώς χρησιμοποιήθηκαν οι ποσοστώσεις τους δασμούς, τι συνέβη με τα υπόλοιπα προτιμησιακά καθεστώτα, δηλαδή το, όταν ε, συμφωνείται μια μείωση ενός δασμού, πώς, ποιο, είναι ο αριθμός των επιχειρήσεων στην Ευρώπη που τελικά υποφελούνται από αυτή τη συμφωνία. Μετά κοιτάμε τον βαθμό των επενδύσεων και τέλος το, το βαθμό της δραστηριότητας των διαφόρων οργάνων που έχουν δημιουργηθεί για την υλοποίηση των συμφωνιών αυτών. Από όλα αυτά τα ε, στοιχεία εξάγουμε δεξί συμπεράσματα. Το μόνο σίγουρο είναι ότι οι συμφωνίες ελευθέρου εμπορίου αυξάνουν τις εξαγωγές μας και ενισχύουν τις εμπορικές συναλλαγές. Να σας δώσω ένα παράδειγμα είχαμε μια αύξηση των εξαγωγών από την Ευρωπαϊκή ε, Ένωση προς το Μεξικό 416%, 470% προς το Μεξικό, 625% ε, προς την Σερβία και 60% προς την Κορέα. Αυτό αφορά μια πολύ μεγάλο εύρος προϊόντων ε, ιδιαίτερα τα αγροτικά προϊόντα, φαίνεται ότι ε, προ... ε, για αυτά τα προϊόντα προκύπτουν και τα σημαντικότερα ωφέλη. Ιδιαίτερα από τις νέες, ε, νέες γενιάς συμφωνίες. Αν δούμε το ζήτημα των ποσοστώσεων των δασμών, ένα άλλο ευαίσθητο θέμα διαπιστώνουμε, ποσοστού μάλλον τη μείωση των δεσμών, διαπιστώνουμε ότι σε πολλέ περιπτώσει δεν γίνεται πλήρε αξιοποίηση αυτή τη δυνατότητα ούτε από τι ευρωπαϊκέ επιχειρήσει ούτε από του εταίρου μα. Και δεν, ε, δεν αξιοποιούμε πλήρω αυτέ τι μειώσει των δασμών. Εδώ τα πράγματα είναι πιο άσχημα γιατί το ποσοστό της μη αξιοποίηση είναι υψηλότερο για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις από ό,τι για τις επιχειρήσεις των εταίρων μα. Τέλος, όσον αφορά την ε, ε, εφαρμογή των στόχων βιώσιμη ανάπτυξη, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι έχει ξεκινήσει ικανοποιητικό διάλογος με τους εταίρους ε, όσον αφορά πολύ περίπλοκα εργασιακά και περιβαλλοντικά ε, ζητήματα τα οποία μας ενδιαφέρουν ιδιαίτερα στις ε, νέες πιο σύγχρονες FTAs συμφωνίες. Ε, και είναι καλό που είμαι σήμερα εδώ γιατί πιστεύω ότι είναι καλό να συνεργαζόμαστε, να δουλεύουμε μαζί σας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο έτσι ώστε να απλουστεύουμε τις, τις δραστηριότητες εκεί που μπορούμε, να ε, άρουμε τις, ε, τα προσκόμματα όπου είναι δυνατόν και βεβαίως να μπαίνουμε σε βάθος σε ορισμένα σημεία και ζητήματα τα οποία πρέπει να συζητούμε εντελεχώς και μαζί σας και με άλλους ενδιαφερόμενους. Νομίζω ότι αυτά θα ήθελα να να σας πω σήμερα. Γνωρίζουμε βεβαίως ότι ε, η κυρία Σαϊφή ε, ε, προετοιμάζει μια έκθεση ίδιας πρωτοβουλίας όσον αφορά την κοινή εμπορική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εν ευθέτω χρόνο θα ασχοληθούμε και με αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρος, εγώ σας ευχαριστώ. Όπως είπα και στην αρχή, δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο στη διάθεσή μας και επομένως δεν θα γίνει συζήτηση πραγματικά σε βάθος. Πιο πολύ ε, θα τεθούν ερωτήματα. Έχουν ζητήσει τέσσερι συνάδελφοι το λόγο. Ενάμιση λεπτό ο καθένας παρακαλώ. Πέντε, πέντε έχουν ζητήσει το λόγο. Ενάμιση λεπτάκι ο καθένας, Μαρία. Euh, euh, Σας ευχαριστούμε πολύ για τις διάφορες πληροφορίες. Βεβαίως με ε, μεγάλη ανυπομονησία θα περιμένω την ίδια την έκθεση έτσι ώστε να μπορέσω να την ε, διαβάσω ε, για να καταλάβω κάθε λεπτομέρεια. Όσον αφορά τους δείκτες βλέπουμε ότι οι δείκτες είναι απολύτως ποσοτικοί δεν πρόκειται για ποιοτικού δείκτε. Είναι ε, εντύπωση δικιά μου σε σχέση με αυτά που είπατε ή ε, στους δείκτε που θα περιλαμβάνονται στην έκθεση θα βρούμε και ποιοτικού δείκτε όσον αφορά το εμπόριο. Δεύτερη ερώτηση και μας απασχολεί το ερώτημα αυτό γιατί έχει ξεκινήσει προβληματισμός για τη γεωργία γενικά. Λέτε ότι ε, το εμπόριο ωφέλησε πολύ τη γεωργία. Υπάρχουν κάποιοι δείκτες ε, όσον αφορά το, το είδος της γεωργίας που ωφελήθηκε περισσότερο γιατί εάν θέλουμε μόνο την ε, εντατική ενεργοποιημένη, ε, ε, καθαρά προσανατολισμένη στη μεγάλη παραγωγή γεωργία, αυτό δεν μας ενδιαφέρει γιατί τότε το διακύβευμα δεν είναι το σωστό ε, και αντιθέτως θα έχει αποτελέσματα που δεν τα θέλουμε. Μας ενδιαφέρουν περισσότερο η διαφοροποίηση της γεωργίας, η βοήθεια στους μικρούς γεωργούς, η πρόθεση γεωργικών πρακτικών λιγότερο επιζήμιων για την υγεία κτλ. Ευχαριστώ πολύ ο κύριος Φίσας. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να συγχαρώ την Κομισιόν για αυτήν την πρωτοβουλία η οποία θεωρώ ότι είναι ιδιαίτερως χρήσιμη. Ε, δύο συγκεκριμένα. Στην Συμφωνία Ελευθέρου Εμπορίου με το Περού και την Κολομβία προστέθηκε και ε, το Εκουαδόρ. Θα ήθελα να ξέρω εάν εάν ε, μαζί με το Περού και την Κολομβία ε, έχει προσθεθεί πραγματικά ε, και αυτή η χώρα των Άνδεων, στις υπόλοιπες μάλλον χώρες των Άνδεων ή είναι κάτι διαφορετικό. Επίσης, και εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό το θέμα της γεωργίας. Νομίζω ότι πάντα έχουμε με την Επιτροπή Γεωργίας έτσι σημεία σύγκρουσης και εδώ νομίζω ότι πραγματικά θα έχουμε ε, σημείο τριβής. Ε, ίσως καλό θα ήταν να έχουμε μια κοινή συνεδρίαση με την Επιτροπή Γεωργίας έτσι ώστε να μας δώσετε τα συγκεκριμένα στοιχεία για τη Γεωργία γιατί ε, συνήθως η Επιτροπή Γεωργίας βλέπει λίγο με μισό μάτι αυτές τις συμφωνίες ελευθέρου εμπορίου. Κάμπε Μπάνεμαν. Um, Πολύ σύντομα κύριε Πρόεδρε σε σχέση με τις πιο σύγχρονες ε, ε, μορφές ε, Καναδά, Νότια Κορέα, Περού, Κολομβία. Υπάρχει αυτό το θέμα των MFN αυτό θα μπορούσε να έχει κάποια σχέση με το Brexit. Ε, θα ήθελα να μας πείτε δύο λόγια γι' αυτό. Ε, υπάρχει δεσμευτική συμφωνία σε σχέση, ε, σε σχέση με μελλοντικές συνολικές συμφωνίες που θα έχουν αυτήν την ρήτρα σχετικά με τη μεταχείριση του μάλλον ευνοούμενου κράτους, MFN treatment. Ε, ποια είναι η άποψή σας γι' αυτό και πόσο δεσμευτική μπορεί να είναι μια τέτοια ρήτρα. Thanks Κύριε Ντάλη, ευχαριστώ πολύ και εγώ θα ήθελα να έχω στην, στα χέρια μου την έκθεση αυτή έτσι ώστε να είναι και πιο σωστές ίσως και σε βάθος οι ερωτήσεις που θα υποβάλαμε. Πολύ ενδιαφέρον θα ήταν να δούμε πληροφορίες σχετικά με την ε, επίπτωση στις εμπορικές ε, ροές. Ε, θέλουμε να δούμε και στο Ηνωμένο Βασίλειο τι θα εγκαταλείψουμε εάν εγκαταλείψουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω ότι λαμβάνοντας υπόψη το, την δεδομένη στιγμή είναι καλό να έχουμε τέτοια στοιχεία. Επίσης σε σχέση με αυτό που είπε και η Μαρία, ποιοτικοί ε, ε δείκτες ε, ε, που να υπόκεινται και στο κεφάλαιο των, ε, της βιώσιμης ανάπτυξης υπάρχουν τέτοιοι δείκτες. θα ήθελα να μας πείτε μερικά πράγματα. Δεν είναι διαδικαστικά μόνο αυτά, είναι ουσίας. Ευχαριστώ πολύ ο κύριος Αλαφράγκα. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε δεν θα μου πάρει ένα μισή λεπτό και εγώ θα ήθελα να πω ότι με ενδιαφέρει πάρα πολύ να διαβάσω ε, αυτή την έκθεση. Θέλουμε μεγαλύτερη διαφάνεια και κυρίως αποτελεσματικότητα των εμπορικών εργαλείων, όχι μόνο για, τα 40, για τις 40 συμφωνίες, αλλά ε, και για άλλα στοιχεία τα οποία είναι πολύ σημαντικά όπως είπε και η Κομισιόν. Εγώ θα ήθελα να ξέρω εάν η ανάλυση των ισχυουσών συμφωνιών περιέχει κεφάλαιο ε, σχετικά με την επίλυση ε, συγκρούσεων και διαφωνιών ε, και κυρίως θα ήθελα να έχω μια ιδέα για τις ρήτρες διασφάλισης που περιλαμβάνονται σε αυτές τις συμφωνίες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Πράγματι είναι δύσκολο χωρίς την έκθεση να συζητούμε για αυτήν την έκθεση. Γι' αυτό λοιπόν ε, μία ερώτηση έχω. Κατά πόσον στην έκθεση περιλαμβάνετε κάτι. Γιατί είπατε για το έστι και τα σχετικά ε, κεφάλαια ότι θα υπάρχει ε, στην έκθεση ένα σχετικό κομμάτι και γίνονται πολλές συζητήσεις από αυτού. Υπάρχει μια προσπάθεια συναγωγής συμπερασμάτων, ποια θα είναι επιπτώσει για το μέλλον δηλαδή για την Κορέα συγκεκριμένα και τη σχετική συμφωνία. Ιδίω ό,τι αφορά την ε, εφαρμογή των εργασιακών δικαιωμάτων. Εκεί υπάρχουν ε, κάποιες συμφωνίες ή απλά γίνεται μία περιγραφή ότι έγιναν ε, συζητήσεις. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Έχετε πέντε λεπτά στη διάθεσή σας. Γιώστ, παρακαλώ, για να απαντήσετε. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, και ζητώ συγγνώμη που δεν υπάρχει ακόμη έκθεση. Θα έχουμε φαντάζομαι τη δυνατότητα να το ξανασύσουμε σας το εγγυώμαι, λέει ο κύριος Λάγκη. Και έτσι θα έχω και πιο πολύ χρόνο να προετοιμαστώ, λέει ο πρόσωπο τη Κομισιόν. Την κυρία Ρενά, ακούστε, οι δείκτες είναι πράγματι ποσοτικοί προς το παρόν, έχετε δίκιο επ' αυτού. Σε ό,τι αφορά τη Γεωργία, δεν νομίζω ότι πηγαίνουμε στο βάθος που θα θέλατε εσείς. Μέχρι στιγμής ε, έχουμε μάκρο οικονομικά ε, στοιχεία για τα γεωρικά πρώτα. Ίσως στο μέλλον θα μπορούσαμε να πάμε λίγο πιο μακριά. Για το κεφάλαιο βιώσιμης ανάπτυξης, η ανάλυση εδώ είναι πολύ πιο ποιοτική. Δεν έχουμε δηλαδή νούμερα. Εκτός από τις συναντήσεις, ε, πόσες συναντήσεις είχαμε, δεν υπάρχουν άλλα νούμερα. Η έκθεση εκεί έχει πολύ πιο ποιοτικό ε, χαρακτήρα, εστιάζει σε ποιοτικά ζητήματα. Το επόμενο ζήτημα για το Εκουαδόρ δεν καλύπτεται ε, στην έκθεση διότι το 2016 προέκυψε και δεν το έχουμε για το Περού και την Κολομβία πράγματι 2006 τέλος πάντων η διάσταση του Brexit είναι σαφές από την έκθεση και την προσέγγιση που ακολουθείται ότι αυτές οι συμφωνίες έφεραν συναλλαγών για την Ένωση θα ισχύουν και το 27 θα έχει φύγει το Ηνωμένο Βασίλειο. Θα πρέπει να δει το Ηνωμένο Βασίλειο τι απώλειες μπορεί να προκύψουν γιατί δεν θα εφαρμόζονται πλέον για το Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτό είναι σαφές. Η επίλυση διαφορών αν καλύπτεται, ναι καλύπτεται. Στο κεφάλαιο όπου γίνεται λόγος για τη δημιουργία θεσμών. Οι παλαιότερες πρώτης γενιάς σύμφωνοι δεν έχουν αυτή τις, αυτές τις ρήτρε, άρα εκεί που δεν αφορά, στις συμφωνίες που δεν αφορά δεν υπάρχει, όπως για την Τουρκία ή για κάποιες άλλες χώρες. Και είναι και πραγματικά ε, αδύνατα σημεία θα έλεγα των συμφωνιών αυτών για ε, έλλειψη τέτοιων ρητρών για το TST και την Κορέα. Αυτά θα τα δούμε σε μια ξεχωριστή έκθεση, γιατί για την Κορέα έχουμε ξεχωριστή έκθεση, όπου κάνουμε μια ποιοτική αξιολόγηση και προσπαθούμε να προχωρήσουμε λίγο πιο πέρα. Δεν αρκεί να σας δώσουμε τον αριθμό των συναντήσεων. Και όπως καταλαβαίνετε δεν είναι αυτή η έκθεση το τέλος. Θα συζητήσουμε στη συνέχεια την εφαρμογή και τις κυρώσεις. Θα συνεχίσουμε φυσικά. Αυτή η έκθεση απλά αναφέρει κάποια πραγματικά περιστατικά, δίνει την εικόνα της κατάστασης, αλλά σίγουρα θα έχουμε ε, μια συζήτηση πιο πολιτική και σίγουρα και πιο πολύπλοκη. Ευχαριστώ, Γιώστη. ο Πρόεδρος. Νομίζω ότι πραγματικά κάναμε ένα πολύ μεγάλο βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Κύριε Πρόεδρε, κύριο Σκάμπερ Μπάνερμαν, δεν απάντησε ο κύριος στην ερώτησή μου για την ρήτρα που αφορά το πιο ευνοημένο κράτος, ε, το MFN, αυτό το παρακάμψατε. Δεν ξέρω να σας απαντήσω, λέει ο κύριος ε, Κόρτ. Ναι, είναι τεχνικό πράγμα. Ναι, θα επανέλθω αν ε, μου επιτρέπει. Ναι, είναι σημαντικό για τις μελλοντικές Ναι, ναι, και για τη Βρετανία. Uh, ο Πρόεδρος, θέλω να σας ευχαριστήσω εκ νέου. Γιώστ, όπως είπα, κάναμε ένα σημαντικό με προς σωστή κατεύθυνση και προσβλέπουμε τώρα στην υλοποίηση των συμφωνιών αυτών. Θα παρακολουθούμε τα σχετικά θέματα και θα συζητήσουμε στο μέλλον, ε, δηλαδή σε μια μελλοντική μας συνδρία, στην έκθεσή σας σε βάθος. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα πηγαίνουμε σε μια συμφωνία που είναι παλαιά με βάση τα κριτήρια του Γιώστο. Ανοίξει την κατηγορία 1. Συμφωνία με το Μεξικό. πρέπει να μπει στην κατηγορία 4. Νέες συμφωνίες. Εφόσον συζητούμε τον εξυγχρονισμό τη εμπορική συμφωνία με το Μεξικό. Δεν θα κάνω κάποια εισαγωγή γιατί δεν έχουμε και πολύ χρόνο στη διάθεσή μας. Απλά θα καλωσορίσω μια αντιπροσωπεία από το Μεξικό. Τον πρέσβη του Μεξικού, την αυτοξοχότητα Σεγκόβια και τον επικεφαλής διαπραγματευτή τον κύριο Γουέρα, που είναι εδώ. Και συνοδεύονται και από άλλα μέλη της, της Μεξικανικής Αντιπροσωπείας. Θα ήθελα να μας πείτε λοιπόν τι γίνεται, πώς προχωρούν οι εργασίες της, ε, του εξυγχρονισμού. Βέβαια, καταρχάς θα ακούσουμε το δικό μας επικεφαλής διαπραγματευτή, πολύ γνωστό από την Κομισιόν. Μάρο, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ. Αλλά θα πρέπει να σας διορθώσω φοβού. Ευτυχώς για μένα δεν είμαι ο επικεφάλης διαπραγματευτής. Ένα συνάδελφό μου έχει την τιμή. Όπως αυτή τη στιγμή μάλιστα ταξιδεύει. Αλλά παρακολουθώ του σύνεγγυ αυτές τις διαπραγματεύσεις και με τα χαρά να σα ενημερώσω. Επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο, θα συντομεύσω την παρουσίασή μου. Και θα σας υπενθυμίσω απλώς ότι είναι κάπως περίεργη αυτή η διαπραγμάτευση που έχουμε για τον εξυγχρονισμό μιας φυστάμενης συμφωνίας. Άρα πολλά είναι ήδη εκεί, παραδείγματο χάρη ε, οι δασμοί. Αυτό έχει οριστεί εδώ και καιρό και είχαμε πολύ καλά αποτελέσματα και για την Ένωση και για το Μεξικό. Υπάρχουν κάποιοι βασικοί κανόνες για τα πραγματικά δικαιώματα, SPS, ε, επενδύσεις, ε, αλλά είναι βασικά, στοιχειώδη, ε, τα πιο πολλά, ιδίω σε ό,τι αφορά τι υπηρεσίε. Άρα, τι θα πει εξυγχρονισμό, ουσιαστικά να ολοκληρωθεί αυτή η συμφωνία, παραδείγματο χάρη, διαπραγματεύσει ε, για του γεωργικού δασμού. Σχεδόν έχουμε ολοκληρώσει για την πρόσβαση υπηρεσίε και εκεί έχουμε σχεδόν ολοκληρώσει και θέλουμε να ε, προσαρμόσουμε κάποια στοιχεία όπως ας πούμε τη συμφωνία με το Καναδά, που επειδή αυτές οι δύο οικονομίες προσωμιάζουν, μπορούμε να έχουμε κάποια προσέγγιση. Πολλές βελτιώσεις λοιπόν, αλλά έχουμε ακόμη διαπραγματεύσεις μπροστά μας. Ο στόχο, ο κοινό στόχο με το Μεξικό είναι οι διαπραγματεύσει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το τέλο του τρέχοντο έτου. Στόχο δύσκολο να επιτευχθεί, αλλά προσπαθούμε να τον επιτύχουμε ακόμη. οι σχέσεις Μάστρου ε, Γκουαχάρντο είναι πολύ καλές και επιβεβαιώθηκε και από τις δύο πλευρές ότι αυτός είναι ο στόχος. Πάντως είμαστε σε μια δύσκολη φάση αυτή τη στιγμή στις διαπραγματεύσεις. Πολύ δουλειά αναμένεται και πρόοδος επίσης πρέπει να επιτευχθεί. Το δικό μας λόγκαν είναι ότι η ουσία έχει την ουσία και όχι ο χρόνος, όχι το timing. Αυτό είναι σημαντικό για όλες τις διαπραγματεύσεις. Για τη συγκεκριμένη διαπραγμάτευση όμω ακόμη πιο πολύ. Γιατί έχουμε συμφωνία με το Μεξικό. Και αν δεν μπορούμε τελικά να τη βελτιώσουμε, δεν έχει και νόημα. Άρα η ουσία είναι πρωτή τη σημασία και παραμένει. Παρότι καλό θα ήταν και για το Μεξικό και για την Ευρωπαϊκή Ένωση να μπορούσαμε να έχουμε ολοκληρώσει τον επόμενο μήνα ή τι επόμενε λίγε εβδομάδε. Γιατί έχουμε δυσκολίε. Το Μεξικό δεν φαίνεται να μπορεί να προχωρήσει τα πράγματα σε ομοσπονδιακό επίπεδο. Γιατί ε, κολλάμε τα πράγματα στις πολιτείες, στο επίπεδο των πολιτιών. Πρέπει να έχουμε κάποια πρόσβαση σε υποομοσπονδιακές προμήθειες και θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε το θέμα αυτό να το λύσουμε. Πρέπει να ενισχύσουμε του κανόνε για τι επιδοτήσει και τι κρατικέ επιχειρήσει. Έχουμε αναπτύξει καλού κανόνε σε πρόσφατε συμφωνίε και με χώρε όπω το Βιετνάμ. Που έχει πιο πολλέ κρατικέ επιχειρήσει από άλλε χώρε. Γιατί λοιπόν να μην το πετύχουμε και με το Μεξικό. Φιλοδοξία δεν είναι επαρκή στο κεφάλαιο αυτό. Με το Μεξικό θα έχουμε μια δεύτερη προσφορά για το κεφάλι των υπηρεσιών. Γεωγραφικές ενδείξεις. Δεν έχουμε διαφορετικούς στόχους. Το Μεξικό έχει από τις λίγες γεωγραφικές ενδείξεις που είναι προστατευμένες στο αλλά η συζητήσεις ε, δεν έχουν την τροπή που θέλουμε. Ξέρετε πόσο ευαίσθητο είναι το θέμα των κεντροφικών ενδείξεων για μας. Εμείς είμαστε διατεθειμένοι να είμαστε ρεαλιστές. Ε, αν υπάρχει πρόβλημα επιτόπου όμως, ειλικρινά, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε δεν νομίζουμε ότι μπορούν να αντιμετωπίσουν πιο εύκολα αν δεν βρεθεί συμβιβασμό. Ένα άλλο κλασικό πρόβλημα είναι η προστασία των επενδύσεων. Εμεί θέλουμε τη μεταρρυθμισμένη προσέγγιση και για το σύστημα το δικαστικό. Δεν θα επανέλθω στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο με ένα σύστημα ISDS διαφορετικό. Μπέρντ, η μόνη διαφορά είναι ότι θα έχουμε ίσως κάποια στιγμή ένα πολυμερές δικαστήριο επίλυσης. και δεν έχουν πιστεί ακόμη οι Μεξικανοί φίλοι μας και δεν είναι και μόνοι, το ξέρουμε αυτό. Είναι στο στρατόπεδο των επιφυλακτικών ως προς το θέμα αυτό. Και αυτό μας δυσκολεύει. Δύο τελευταία. Δύο τομείς όπου δεν υπάρχει καμία απόκληση απόψεων μεταξύ μόνο και του Μεξικού ως προς την κατεύθυνση. Υπάρχουν όμως διαφορές ως προς το πώς θα πάμε εκεί. Καταπολέμηση διαφθορά σε εμπόριο. Εκεί έχουμε προβλήματα με την προσεξτήστη. Όμως ετάστε αυτό σε μια συμφωνία. Διαβουλεύσουμε με τις κοινωνία των πολιτών όχι μόνο το εμπορικό σκέλος ή το TST. Έχουμε τους συναδέλφους ΕΕ, από την ΕΕ, την Εξωτερική Υπηρεσία, για το γενικό κομμάτι. Έχουμε μια καλύτερη πρόβλεψη για διαβουλεύσεις με την κοινωνία των πολιτών για το σύνολο της συμφωνίας και όχι το TST μόνο. Η διαπραγμάτευση είναι ξεχωριστή όμως, γι' αυτό δεν το βλέπετε. Της ουσίας δεν έχουμε κάποια διαφορά για την προσέγγιση, αλλά δυσκολευόμαστε στο θέμα της επιβολής. Uh, Θέλαμε να δούμε τι θα πρόκειται από τη συζήτηση σε επίπεδο του Συμβουλίου αν χρειάζεται αλλαγή προσέγγισης για την υποτίστη. Δεν έχει ολοκληρωθεί αυτή η συζήτηση. Έχει υπευραδυνθεί κάπως. Ή τέλος πάντων είναι, δεν είναι τόσο γρήγορα, τα, η εξέλιξη δεν είναι τόσο γρήγορα όσο θα θέλαμε. Ε, Εμεί έχουμε την εντολή μας και θέλουμε και τη ρήτρα αναθεώρησης για να μπορούμε να ξανασυζητήσουμε το Μεξικό εφόσον αλλάξει προσέγγιση η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί την τη της διαφθοράς. Αυτό είναι κάτι καινούριο. Για ε, πρώτη φορά έχουμε ένα τέτοιο κεφάλαιο. Λεπτομέρειες ξέρετε και αν έχετε ερωτήσει θα προσπαθήσω να σας απαντήσω. Θα πω ένα σημαντικό. Δύο είναι οι βασικές αρχές. Πρώτον, επιβεβαίως πολυμερούς δέσμευσης. Αυτό δεν είναι καινούριο. Αυτή την προσέγγιση ακολουθούμε πάντα στο τα πρότυπα είτε αφορούν αξίες, είτε αφορούν προϊόντα, είτε αφορούν εργασιακά δικαιώματα, είτε την κατασκευή ενός οχήματος. Έχουμε τη συγκεκριμένη αυτή πολιτική. Το νέο όμως στοιχείο είναι προσπάθεια να έχουμε διμερείς κανόνες για την αποτροπή, την πρόληψη. Δυστυχώς και αυτό είναι κάτι καινούριο στο δεύτερο προσκήνιο. Δεν μπορούμε να προσκεφθούμε ότι θα λειτουργήσει. Γνωρίζουμε όμως από την άλλη ότι ο κολλασμός της διαφθοράς είτε θα είναι συστηματικός, γιατί τέλος θα λειτουργήσει, γιατί πρέπει να εξαλειφθούν τα αίτια. Σταματήσω εδώ, Μπέρντ. Και κατακλείδη θα πω ότι το Μεξικό είναι σημαντικό, επειδή είναι το Μεξικό, και επειδή το εμπόριο με το Μεξικό τα πηγαίνει πολύ καλά και από τα συμφωνία. Αλλά και συστημικό έχει μεγάλη σημασία. Γιατί ζούμε σε, ένα, σε μια εποχή όπου η δική μα προσέγγιση στι εμπορικέ συμφωνίε με βάση τις αξίες και τις αρχές, τι κοινέ είναι σε κίνδυνο. Έχουμε τα εμπορικά ισοζύγια, τι ανισορροπίε, και πρέπει να ε, συνεργαστούμε με τους ώστε να επανεπιβεβαιωθεί ότι το ανοιχτό δίκαιο εμπόριο με βάση κοινού κανόνες είναι η μόνη οδός. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστούμε πράγματι. Αυτό το τελευταίο, τελευταία παρατήρηση σα την επαναλαμβάνω και συμφωνώ πλήρω. Το λόγο στον εισηγητή μα τον κύριο Μόιζα. Θα ξεκινήσω από το τελευταίο που ανέφερε ο Μάουρο και τον οποίο ευχαριστώ για την παρουσία του εδώ. Η προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τις εμπορικές συμφωνίες έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια και με τη σημαντική συνεισφορά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτό σημαίνει ότι σήμερα πλέον η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να καλύψει το κενό που δημιουργείται στην παγκόσμια οικονομία που αφήνουν άλλοι και να προσπαθήσει να ε, προασπίσει τα συμφέροντά της, ε, όμως κάνοντας το αυτό προωθώντας τις αξίες της. Και σε αυτό το πνεύμα πιστεύω ότι είναι σημαντικό να ολοκληρώσουμε τη συμφωνία με το Μεξικό στο δυνατόν συντομότερα, δηλαδή μέχρι το τέλος της χρονιάς. Ε, είναι ένας τρόπος επίσης να δείξουμε σε μια φιλική χώρα ότι την υποστηρίζουμε σε μια περίοδο αστάθειας αβεβαιότητας και όπως είπε και ο Μάουρο θα ε, έχει και ε, ουσιαστικά πλεονεκτήματα η νέα συμφωνία θα πρέπει να είναι συμβατή με την νέα προσέγγιση την οποία προσπαθούμε να ακολουθούμε και στη βάση της οποίας έχουμε προσπαθήσει να νομιμοποιήσουμε τις πολιτικές επιλογές που έχουμε κάνει στην εμπορική μας πολιτική. Γι' αυτό έχει σημασία και το timing αυτής της συζήτησης ε, που έρχεται σε μια στιγμή που ε, είναι κρίσιμη για την πορεία της διαπραγμάτευσης. Ε, και έρχομαι λοιπόν στα θέματα που ο Μάουρο ανέφερε ως ανοιχτά η σχέση της συμφωνίας αυτής με την πιθανότητα να ξανανοίξει η διαπραγμάτευση της ναύτα. Δεν θα ήταν καλύτερο να αναμένουμε να δούμε το αποτέλεσμα αυτής της α, συζήτησης. Για τα αγαθά η ε, ε, διαπραγμάτευση είναι πολύ σημαντική γιατί στεγόμαστε στα ευαίσθητα για μας προϊόντα, δηλαδή τα αγροτικά και τα αλλιευτικά. Για τις υπηρεσίες ε, καταλαβαίνω από την παρουσίαση του Μάουρο ότι υπάρχουν διαφορές στην προσέγγιση και στις διώξεις της κάθε πλευράς. Η ερώτησή μου είναι ποια είναι η σχέση αυτών των επιδιώξεων με, με τους στόχους που θέσαμε στην ΤΙΣΑ. Στην ΤΙΣΑ είχαμε προσπαθήσει και όπως και στην ΑΦΤΑ να έχουμε ε, την προσέγγιση του MSN, του μάλλον ευνοούμενου κράτους. Ε, ίσως αυτό βέβαια ξανανοίξει στο πλαίσιο της για την ΑΦΤΑ. Όσον αφορά την απελευθέρωση, ε, το ζήτημα αυτό είναι σημαντικό για μας, το ανέφερε και ο Μάουρο από την πλευρά του ICS. Και ένα άλλο σημαντικό ζήτημα είναι η πρόσβαση στις αγορές, στις διάφορες αγορές του Μεξικού. Τώρα, όσον αφορά το ρυθμιστικό πλαίσιο, φαντάζομαι και ελπίζω ότι δεν θα πέσουμε στην παγίδα να ακολουθήσουμε αυτή την κυκλική προσέγγιση που ακολουθείται στην Αμερική, ότι μπορεί κανεί να κάνει οτιδήποτε επιθυμεί αρκεί να μην παραβιάσει τη συμφωνία. Ε, έχουμε τι πολιτικέ μας όσον αφορά αυτό. Ε, ένα άλλο ζήτημα που θα μα απασχολήσει και που είναι πολύ σημαντικό είναι η πρόσβαση που θα έχουμε στι δημόσιε προμήθειε. Κάτι ακόμα είναι η ροή των δεδομένων και ποια ρύθμιση θα ε, δεχτούμε τελικά σε αυτή. Όσον αφορά την επίλυση διαφορών, γνωρίζετε ότι είχαμε μια προσέγγιση την οποία φάνηκε από την διαπραγμάτευση με την ΤΙΣΑ αλλά και με άλλες χώρες ότι θα πρέπει να πάμε προς μια κατεύθυνση κυρώσεων Αυτό δεν είναι προφανώ μια υποχρέωση, το γεγονό ότι το υποθετήσαμε σε άλλε συμφωνίε, αλλά δείχνει ένα σήμα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι πρέπει να το εξετάσει ω μέθοδο. Τώρα, δεδομένου του πώς λειτουργεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, υπάρχει μια συγκεκριμένη διατύπωση, η οποία τελικά προκύπτει από την ε, συμφωνία των διαφόρων πολιτικών ομάδων σε ένα ψήφισμα. Ε, το Μεξικό το έχει ήδη δει αυτό και το έχει αποδεχτεί. Έρχομαι στα συμπεράσματα, γιατί μου δώσατε πέντε λεπτά, έχω μιλήσει τέσσερα. Συμπερασματικά. Πώς μπορούμε να λύσουμε το ζήτημα του TSD. Η Συμφωνία των Παρισίων έχει, είναι ένα καλό παράδειγμα. Κάθε μέρος της συμφωνίας δεσμεύεται να την υλοποιήσει. Και γνωρίζουμε ότι το Μεξικό τη σκοπεύει να ε, είναι μια από τι χώρε οι οποίε ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για την καταπολέμηση τη κλιματική αλλαγή. Επομένω, είμαστε σίγουροι ότι θα προσπαθήσει να ελπίσει τη Συμφωνία του Παρισίων παρά το γεγονό ότι το κείμενο του σχετικό βρίσκεται ακόμα σε αγγείλε. Ε, θα ήταν σκόπιμο, πιστεύω, να, ιδιαίτερα ξεκινώντας από εταίρους μας οι οποίοι ήδη το σέβονται αυτό, να βάζουμε τις αναφορές στη Συμφωνία των Παρισίων σιγά σιγά στις εμπορικές μας συμφωνίες. Επίσης, οι αναφορές στις συμφωνίες του ILO. Προβλέπεται και προτείνεται να προβλέπεται ότι ο Διεθνής Οργανισμός Εργασίας θα έχει τη δυνατότητα να ερευνά και να να καταλήξει μια έκθεση για τα πραγματικά περιστατικά όταν δεν υπάρχει κάποιο πρότυπο το οποίο να έχει πληρωθεί από την χώρα. Και αυτό είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Ίσως λοιπόν αυτές, αυτές οι δύο μέθοδοι που σας παρουσίασα να είναι ένας τρόπος να πάμε προς τη σωστή κατεύθυνση παρά το γεγονό ότι δεν κλείνουν όλη τη συζήτηση που έχουμε για το TSD. Ωραία. Κάνουμε κάποιες ε, γενικές ε, παρατηρήσεις. Δύο λεπτά. Πρώτος ηγητής, κύριος Φίσας. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Χαίρομαι γιατί βλέπω ότι υπάρχει πραγματική ε, ικανότητα, δυνατότητα να ολοκληρωθεί η συμφωνία φέτος. Νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχουμε ιστορικά, ε, ιστορικούς δεσμούς ε, με το Μεξικό και αξίζει τον κόπο να καταβληθεί η ε, προσπάθεια. Νομίζω ότι η συνεργασία με τον συνάδελφο εισηγητή κύριο Μόησα ήταν πάντα πολύ καλή νομίζω και σε σχέση και με αυτά που είπε η Κομισιόνα βλέπω ότι με ικανοποίηση αυτή την αναφορά της αύξησης των εμπορικών ροών μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Μεξικού Μεξικό που ε, ε, ξεπερνάει το 400%. Αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Αλλά έχω και κάποιες ε, ερωτήσεις το θέμα που ανέφερε και ο εισηγητής κ. Μόιζα όσον αφορά τις δημόσιες, τους δημόσιους διαγωνισμούς Γνωρίζω το Μέξικο καλά. Ε, εν πάση περιπτώσει όμως, εάν το Μεξικό ε, μπορεί ε, να έρθει σε επαφή με όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν είμαστε ακόμα, δεν έχουμε ακόμα μορφή ομοσπονδιακή, θα πρέπει αντίστοιχα να υπάρχει και η δυνατότητα εμπορικών αντιστοίχων σχέσεων με όλα τα κρατήδια του, του θα ήθελα να ξέρω δε την επιχειρηματολογία σχετικά με το θέμα αυτό της ε, μεξικανικής ε, πλευράς. Επίσης, μία διευκρίνηση όσον αφορά την ενέργεια και τους, ε, τις πρώτες ύλες. Ποια είναι τα επιχειρήματα, πού βρισκόμαστε εδώ και επίση όσον αφορά τους κανόνες ε, για την προέλευση, ξέρω ότι είναι πολύ τεχνικό το ζήτημα, ωστόσο είναι και πάρα πολύ σημαντικό, είναι, πολύ, ε, είναι θεμελιώδου σημασίας να μπορούμε να καθορίσουμε ε, την προέλευση των προϊόντων, σε ποιου τομεί θα ισχύσει αυτό, με ποιο τρόπο. Σας ευχαριστώ πολύ. Άλντε δεν είναι εδώ ο, ο και αντικαθίσταται. Ευχαριστώ πολύ. Η ομάδα Άλντε απολύτως προσυπογράφει την ε, ε όσο γίνεται πιο σύντομα ε, επικαιροποίηση της Συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Μεξικό ε, γιατί θεωρεί ότι προς ώρας δεν χρησιμοποιούμε όλο το δυναμικό ε, το οποίο μπορεί να ε, περιλαμβάνει η σχέση αυτή. Ε, υπάρχουν ακόμα δασμολογικές, δασμολογικά εμπόδια τα οποία θα πρέπει να αμβληθούν. Επίσης στην εξυγχρονισμένη μορφή της συμφωνίας θα πρέπει να περιλαμβάνει για την προστασία των δεδομένων. Αυτό είναι καλό και για το Μεξικό αλλά και γενικότερα για τον καθορισμό ορίων για τα δεδομένα. Το κάναμε με την Ιαπωνία, δεν είναι δυνατόν να μπορούμε να το κάνουμε με το Μεξικό. Ευελπιστούμε ότι ε, μέχρι τα τέλη του μήνα θα έχουμε αρκετή πρόοδο έτσι ώστε να ορκωθεί η συμφωνία. Ευχαριστώ πολύ Μαρία Ρενά. Ευχαριστώ. Μία ερώτηση τεχνικής μάλλον φύσεως που αφορά το θέμα ε, της, ε, του μείγματος μετά από την απόφαση της ε, Σιγκαπούρης ξέρουμε ότι υπάρχει ένα τμήμα το οποίο θα είναι non-mixed και άλλο ένα τμήμα το οποίο θα είναι στο κοινό mixed όπως ας πούμε είναι οι επενδύσεις ε, στη βελτίωση της συμφωνίας με το Μεξικό πώς την βλέπετε ε, στα πλαίσια αυτής της νέας συμφωνίας στα τμήμα μεικτό ή μη μεικτό πώ πώς πιστεύετε ότι θα μπορείτε να διαχειριστείτε καλύτερα δεύτερο ε, όσον αφορά τη βιώσιμη ανάπτυξη. Είπατε ότι η λύση θα μπορούσε, αν κατάλαβα καλά, να είναι η ρήτρα αναθεώρησης και επομένως ε, να μπορέσετε έτσι να συνεχίσετε όσον αφορά το θέμα αυτό. Η θέση ε, της ομάδας μου τουλάχιστον ήταν σαφής. Το κεφάλαιο τη βιώσιμης ανάπτυξης ε, ε, με το θέμα των κυρώσεων που δεν θα πρέπει να αφορά μονάχα ε, τη βιώσιμη ανάπτυξη αλλά θα πρέπει να ισχύει με τον ίδιο ακριβώ τρόπο επί του συνόλου της συμφωνίας η θέση λέω, της ομάδας μου ήταν σαφής. Αναφέρατε το θέμα των κυρώσεων αλλά θα ήθελα να, το να, μας, να μας το αναφέρετε σε σχέση με το ερώτημα το οποίο υποβάλλω εγώ γιατί υπάρχει εν πάση περιπτώσει μια συμφωνία, μια βάση συζήτησης με το Μεξικό. Σας ευχαριστώ πολύ και η Καρολίνα τελευταία. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το ερώτημά μου είναι ότι χθε έγινε για το ψηφιακό εμπόριο μία ακρόαση και εκεί ε, μας είπαν ότι στη συμφωνία με το Μεξικό ε, προβλέπεται κεφάλαιο σχετικό. Ε, θα μπορούσατε να μας πείτε πράγματι ισχύει αυτό, υπάρχουν έγγραφα τα οποία θα μπορούσαμε να ε, συμπεριλάβουμε και να ενημερωθούμε για αυτά. Μάουρο, έχεις 5-6 ε, λεπτά. Α, συγγνώμη. Please, you have to waste your hand, Mr. Salafranca. Δεν σας είδα, να σκόντε τα χέρια σας, κύριε Σαλαφράγκα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ήθελα να συμφωνήσω ότι αυτή, να υπενθυμίσω ότι πρόκειται για μια συμφωνία σύνδεσης εκτός από την ε, ελεύθερη ε, ελεύθερο εμπόριο. Εγώ είμαι συγητή στην Ανεμόδια Επιτροπή για το θέμα αυτό και θα ήθελα να υπενθυμίσω αυτό που μας είπε ο κύριος Φίσας ε, το οποίο μάλιστα το είχε ε, αναφέρει ο προηγούμενος ε, ομιλητής της Κομισιόν. 416% έχουν αυξηθεί οι ανταλλαγές με το Μεξικό επί της βάσης της προηγούμενης συμφωνίας, αλλά επιπλέον υπάρχει και μία σημαντική τροποποίηση της φύσης των προϊόντων που έχει εξάγει το Μεξικό από το 25% των, ε, προϊόντων πρώτης, ε, πρώτων υλών έχουμε φτάσει σε 75% προϊόντων με προστιθέμενη αξία. Επομένως, ε, θα ήθελα να μας πει η Κομισιόν δύο λόγια σχετικά με τον στόχο εκπλήρωσης μέχρι το τέλος του χρόνου. Έχουμε δει δύο μάλιστα δηλώσεις του Συμβουλίου και από την Κομισιόν. Ένα, μία δήλωση από τον πρόεδρο της Κομισιόν και καταλαβαίνω βεβαίως όταν ήρθε να μα δώσει τα αποτελέσματα του Συμβουλίου. Ε, καταλαβαίνω ότι δεν θέλουμε να θυσιάσουμε κατά κάποιο τρόπο το περιεχόμενο τη συμφωνία, αλλά εδώ πρέπει να δούμε εάν έχουμε τη δυνατότητα να επιτύχουμε βελτίωση των συνθήκων και θα πρέπει να δούμε και να μετρήσουμε τον πόη μα, να δούμε αν μπορούμε να ε, έχουμε τι φιλοδοξίε μια συγκεκριμένη πολιτικής, εμπορικής πολιτικής. Το Μεξικό ε, όσον αφορά την ενέργεια και τις τηλεπικοινωνίες έχει κάνει πάρα πολύ μεγάλε μεταρρυθμίσεις ε, ε, και δεν θα πρέπει εμείς να μείνουμε στην ουρά ε, περιμένοντας να δραχθούμε της ευκαιρίας ε, αυτής της τροποποιημένης κατάστασης και επομένως όπως είπε και η Επίτροπος Μάλστρομ πιστεύουμε ότι η Κομισιόν θα πρέπει να δράσει με τρόπο ώστε να προκύψει αυτή η συμπροματική συμφωνία. Εγώ κύριε Πρόεδρε συμφωνώ με τη γραμμή του εισηγητού και έχω και εγώ μια ερώτηση όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα Εάν ξέρουμε ότι έχει ξεκινήσει η διαδικασία αναθεώρησης της ναύτα, θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να περιμένει να ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτή πριν προχωρήσει. Ε, εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να δει τα δικά της συμφέροντα. Ευχαριστώ πολύ ο κύριος Φερόν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε συντονιστής, ε, παρεμβαίνω ως συντονιστής ε, της Ευρώπης των Εθνών να υπενθυμίσω λίγο όσον αφορά τη μορφή κάτι. Από το 2006 η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, ξεκίνησε τη διαδικασία σειράς, ε, υπογραφής σειράς συμφωνιών ελεύθερου εμπορίου που συνέβαλαν εις την άρση κάποιων ε, περιορισμών δασμολογικών και εμπορικών. Το λέω γιατί από την αρχή της ε, θητείας ε, βλέπουμε πολλές συμφωνίες. Η συμφωνία ΣΕΤΑ, ε, συμφωνία με την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία. Βλέπουμε επίσης τις δυσκολίες που έχει η Μερκοσούρ να υλοποιηθεί και τώρα μας υποβάλλεται αυτή η νέα συμφωνία με έναν οικονομικό παράγοντα πολύ σημαντικό όπως είναι το Μεξικό. Πριν υποβάλω την ερώτησή μου λοιπόν, θα ήθελα να πω ότι θεωρώ ότι η παρουσίαση που μας έγινε ε, μας βάζει λίγο κάποιες σκέψεις αμφιβολίας σχετικά με το κατά πόσο είμαστε έτοιμοι για τη συμφωνία με το Μεξικό. Το έγγραφο το οποίο, στο οποίο γίνεται σαφής αναφορά ε, στην ε, ε Συμφωνία θέλω να ξέρω εάν πρόκειται για μια συμφωνία η οποία στην ουσία έχει ε, παρακάμψει το πρόβλημα με τις Ηνωμένες Πολιτείες ή όχι. Η ερώτησή μου τώρα είναι πάρα πολύ απλή. Σήμερα η Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Μεξικό μήπως θα αποτελέσει την ε, νέα βάση επί της οποίας θα πατήσει η βελτίωση της ε, συμφωνίας ε, ε, των Ηνωμένων Πολιτειών και θα οδηγήσει δυστυχώς σε μια νέα συμφωνία ελεύθερων ανταλλαγών. Πολύ σύντομα κύριε Πρόεδρε. Εμείς ως ECR βλέπουμε πολύ θετικά αυτή την συμφωνία. Αλλά έχω και κάποια ερωτήματα. Αναρωτιόμαστε εάν οι διαπραγματεύσεις με την ναύτα ε, με οποιοδήποτε τρόπο επηρεάζουν αυτήν την, ε, το Μεξικό στη διάρκεια αυτής της δικιάς μας συμφωνίας. Δεύτερον, μπορείτε να μας πείτε περισσότερα ε, σχετικά με τα εμπόδια τα οποία τίθενται όσον αφορά τις δημόσιες προμήθειες, δημόσιους διαγωνισμούς. Ευχαριστώ. You're really not generous today, are you? Um, all right, in which case... Μάλιστα. Ζητώ συγγνώμη που δεν μπορώ να σας δώσω λεπτομέρειες. Θα τα πω όσο πιο γρήγορα μπορώ. Είμαστε όλοι στη διάθεσή σας. Μπορούμε να επανέλθουμε ή αν θέλετε στείλτε μας στους συνεργάτες σας για να πάρουν λεπτομέρειες. Εφόσον οι απαντήσουν δεν σας ικανοποιήσουν εκ των προτέρων σας ζητώ συγγνώμη που δεν θα τα καλύψω όλα και ξεκινώ γιατί η συμφωνία, γιατί τώρα ναύτα, συμφωνία σύνδεσης. Μας υπενθύμισε και ο κύριος ε, Σάλαφρακ ότι πρόκειται για μια συμφωνία σύνδεσης, ε, τη λέμε συνολική συμφωνία. Πάνω από 10 χρόνια έχει τεθεί σε ισχύ και λειτουργεί πάρα πολύ καλά. Της λείπουν κάποια πράγματα, είναι η πρώτη, ε, η δεύτερη τέλος πάντων από τις πρώτες γενιάς συμφωνίες. Και κάτι που δεν έχει είναι το TST ας πούμε, το κεφάλαιο που και μόνο αυτό ε, είναι λόγος για να υπάρξει αυτή η τροποποίηση, ο εξεχρονισμός. Πρόκειται για μια συμφωνία σύνδεσης. Και να τη δούμε συνολικά. Μην δείτε τα άλλα τμήματα. Μίλησα για την κοινότητα των πολιτών, ένα μόνο από τα πολλά άλλα ενδιαφέροντα. σχέση με τη Συμφωνία των Παρισίων, αν θα πρέπει να είναι αυτή μια ρήτρα. Εμείς θα ήμασταν υπέρ. Οι συνάδελφοι από την θα ΕΕ ασχολούνται. Σε αυτή τη συζήτηση έχουν λόγο τα κράτη-μέλη απευθείας. Δεν ξέρω τι θα γίνει, αλλά θα είναι καλό να συμβεί. Να αυτά. Αν θα πρέπει να περιμένουμε. Αν περιμένουμε για κάθε διαπραγμάτευση που συμμετέχουν οι εταίροι μας και το αντίστροφο θα περιμένουμε μέχρι τη Δευτέρα παρουσία. Το ίδιο πρόβλημα το είχαμε και το ξεπεράσαμε περίπτωση αυτή θα δούμε αν πρέπει να περιμένουμε, να δούμε δηλαδή πόσο δύσκολα μπορούν τα πράγματα για το Μεξικό, τι θα γίνει με την ναύτα. Δεν μπορώ όμως να προδικάσω. Εμείς δεν θέλουμε να περιμένουμε, δεν είναι αυτή η πρόθεσή μας και δεν έχουμε από το Μεξικό και κάποια ένδειξη ότι και αυτοί περιμένουν ή θα περιμένουν. Κάποιες φορές η ζωή γίνεται πιο δύσκολη από ό,τι μπορεί να περιμένει κανείς. Δεν σας λέω τι θα γίνει ή τι δεν θα γίνει, γιατί δεν μπορώ να το ξέρω. Σας λέω ότι δεν είναι πρόθεσή μας να συμβεί. Αν συμβεί θα είναι παρά τη θέλησή μας. Υπηρεσίες σε σχέση με σίτα, ναύτα και τα λοιπά. Ο στόχος μας είναι κατά τάξη μεγέθους ό,τι έγινε με σύτα και η Ιαπωνία. Θα υπάρχουν κάποιες διαφορές στις λεπτομέρειες να σας δώσω ένα παράδειγμα. Θαλάσσιες μεταφορές δύσκολα με, την, ε, με τον Καναδά, πιο δύσκολα με την Ιαπωνία, πολύ λιγότερο με το Μεξικό. Υπάρχουν άλλοι τομείς όπως είναι οι μετακινήσεις ανθρώπων. Με τον Καναδά έχουμε δυσκολίες. Ε, ε, με την Ιαπωνία όχι τόσες και με το Μεξικό θα έχουμε δυσκολίες και υπάρχουν κάποιες λεπτομέρειες που μας περιορίζουν αλλά υπάρχει επίπεδο φιλοδοξίας ε, αντίστοιχο με συνταγή Για το δικαίωμα αριθμισή. Έχουμε την προσέγγισή μας και έναν απόσπαστο τμήμα της προσέγγισής μας. Και δεν θέλουμε να μετακινηθούμε. Εγώ την ευρωπαϊκή θέση σας λέω. Δεν συμφωνεί σε όλο το μυξό, γιατί αν συμφωνούσα θα είχαμε ολοκληρώσει. Ελπίζω να μπορέσουμε να τους πείσουμε ότι δεν έχουν να φοβούνται τίποτα από την προσέγγιση αυτή και το αντίθετο είναι προ το συμφέρον του Μεξικού. Δημόσια συμβάσει. Πολύ σημαντικό να έχουμε πρόσβαση στο υπο-ομόσπονδο επίπεδο. Το τι θα γίνει θα το δούμε. Υπάρχουν νομικοί περιορισμοί ε, και το Μεξικό προσπαθεί να τους, ε, να παρακάμψει. Το έχουμε κάνει μάλιστα στους δικές χώρες όπως ο Καναδάς. Μια από τις πιο δύσκολες ομοσπονδιακές χώρες που θα αντιμετωπίσουμε λόγω παράδοσης είναι πολύπλοκο με το Μεξικό, δεν μας εκπλήσει που αυτό δείχνει να είναι δύσκολο και μας παίρνει χρόνο. Ροές δεδομένου. Θα το παρακάμψω για τον πολύ απλό λόγο. Την κατάσταση τη γνωρίζετε. Υπάρχει συζήτηση στην Κομισιόν, δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη. Οπότε εγώ δεν είμαι σε θέση να σας πω το οτιδήποτε που να βγάζει νόημα σήμερα. και κυρώσεις. Έχουν ε, ακουστεί δυνατές φωνές, ξεκάθαρες φωνές από το Κοινοβούλιο για τις κυρώσεις. Δεν θέλω να μπω σε συζήτηση για το τι σημαίνει κυρώσεις κτλ. Έχει τελειώσει αυτή η συζήτηση. Εμείς είμαστε υπόλογοι στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Και συγγνώμη που τώρα, αλλά θέλουμε μια σαφή ένδειξη και οδηγία για να αλλάξουν προσέγγιση. Ότι υπάρχει θέμα υπάρχει. Είναι σαφές. Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να προδικάσουμε. Τίποτα στις τρέχουσες διαπραγματεύσεις μέχρι να τις ολοκληρώσουμε. Και θα αδράξουμε τη σωστή στιγμή γιατί και πάλι έχει δει και ο κύριος Αλαφράκο ότι αυτή είναι η σωστή στιγμή. Μπορούμε, θα δείξει. Πιστεύω ότι μπορούμε, αλλά δεν είμαι σίγουρος. Αν μπορούμε να το κάνουμε τώρα, θα είναι μια συμφωνία που θα συμπεριλαμβάνει περί πολύ σημαντικά πράγματα. Συμβάσει ε, διεθνού οργάνωση εργασία. Στο μεξικανικό σύστημα υπάρχει ε, ελπίδα τώρα ότι θα υπογραφεί τελευταία σύμβαση. Θα μας ενημερώσει ομόλοι. Αλλά είναι ένα θέμα ενώπιον του Κογκρέσου του Μεξικού και είναι εθνική κυριαρχία ζήτημα. Ξέρουμε ότι και κάποια κράτη-μέλη δεν είχαν εφαρμόσει και δεν είχαν ε, επικυρώσει όλες τις συμβάσεις. Εμείς δεν θα συνεχίσουμε, δεν θα σταματήσουμε, συγγνώμη, να προσπαθούμε να πείσουμε το Μεξικό με τα επιχειρήματά μας. Ότι αυτό είναι το σωστό. Ούτε πριν, ούτε κατά, ούτε μετά δεν θα σταματήσουμε να πιέζουμε το Μεξικό. Είναι σημαντικό κομμάτι της πολιτικής μας. Και δεν θα αφιστούμε να προσπαθούμε να τους πείσουμε ότι πρέπει να την εφαρμόσουν και να την επικυρώσουν βέβαια πρώτα αυτή την σύμβαση. Ενέργεια πρωτεσίλες. αρκετά ανοιχτή αγορά ε, της ενέργειας στο Μεξικό και στην Ένωση. Θα προσπαθήσουμε αυτό να μπει στο σχετικό κεφάλαιο. Έχουμε πρόοδο, αλλά έχουμε κάποιες δυσκολίες, περιορισμοί σε εξαγωγές λόγω της πολιτικής του Μεξικού. Θέλουμε να του εξαλείψουμε αυτούς τους περιορισμού αυτό είναι ένα δύσκολο σημείο. Αλλά στο κεφάλαιο αυτό γενικά υπάρχει συνένεση. Κανόνας προέλευση. Τα περισσότερα κεφάλαια τα έχουμε κλείσει. Και είμαστε κοντά στο να κλείσουμε και τα υπόλοιπα. Ένδυση, κλωσεφαντουργία, μεταποίηση και αυτοκίνητα οχήματα. Αυτή είναι η τομή που μένουν ανοιχτή και είναι κατανοητό για το μείγμα. Μετά τη γνωμοδότηση του δικαστηρίου ήταν σαφές το τι θα γίνει με τις εφιστάμενες συμφωνίες. Δεν θα τις... Ε, yes, it has to be reconcluded and ratified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 Όταν ξεκίνησαν οι πραγματεύσει για τον εξοικονομισμό τη συμφωνία μα, είχαμε πέντε επίσημου γύρου, εντάσθηκαν οι διαπραγματεύσει από φέτο ε, και πρακτικά κάθε μήνα συνεδριάζαμε είτε επίσημα είτε διοργανικά και αυτό δείχνει ε, πόσο δεσμευμένα είναι τα δύο μέρη για να προσπαθήσουμε να ολοκληρώσουμε φέτος τις διαπραγματεύσεις. Βέβαια για αυτό το σκοπό έχουμε την επόμενη εβδομάδα συνεδρίωση ορισμένων ομάδων στις Βρυξέλλες και έχουμε και τον έκτο γύρο διαπραγματεύσεων στις, ε, την εβδομάδα της 27ης Νοεμβρίου στην πόλη του Μεξικού και μια ε, πρόσθετη 18 Δεκεμβρίου συνεδρία συνεδρίαση Βρυξέλλες, σε υπουργικό επίπεδο αυτή τη φορά. Έχουμε ολοκληρώσει δύο μόνο ε, κύκλους, δύο τραπέζια ε, και ήταν νομίζω θετικά, ενθαρρυντικά τα δείγματα. χάρη για την καταπολέμηση της διαφθοράς. Η πρόταση της Ένωσης ε, πριν ε, από ένα μήνα, στον πέμπτο γύρο διαπραγματεύσεων, ε, διαβιβάστηκε στην πλευρά. Είδαμε τη ε, χρηματοοικονομική αναφορά, διαφάνεια στον ιδιωτικό τομέα, ξέπλυμα χρήματο. Πρέπει να έχουμε υπόψη ότι η εστίαση στα θέματα τη καταπολέμηση τη διάβρωση των εμπορικών πυλώνα πρέπει μόνο στι επενδύσει και το εμπόριο να περιοριστεί. Σε άλλα θέματα έχουμε σημαντική πρόοδο, όπω εμπόριο με βιώσιμη ανάπτυξη. Μέχρι ε, τις πρόσφατες διαπραγματεύσεις όπως είναι η συμφωνία με τον Ειρηνικό κτλ. Το Μεξικό μέχρι τότε δεν είχε διαπραγματευτεί κεφάλι για περιβαλλοντικές ούτε εργασιακές πτυχές στις διεθνείς εμπορικές του συμφωνίες και επομένως είναι μια από τις πρώτες εμπειρίες μας για συγκεκριμένα αυτά θέματα που αφορούν την βιώσιμη ανάπτυξη και το εμπόριο. Μεξικό και Ευρωπαϊκή Ένωση είχαμε επικοδομητικό διάλογο μέχρι τώρα και έχουμε βρει σημεία σύγκληση που υπερβαίνουν τους γενικούς συμβιβασμούς και ένα γενικό πλαίσιο συνεργασίας, αλλά εξετάζουμε πλέον και ειδικέ διατάξεις συγκεκριμένες για τη διατήρηση και τη βιώσιμη χρήση της βιοπικιλότητας. Βιώσιμη διαχείριση δατοκαλλιέργειας ε, και θαλάσσιων αποθεμάτων, κλιματική αλλαγή, ε, φωδιαστική αλυσίδα κτλ. Ένα από τα πιο πολύπλοκα ζητήματα τη διαπραγμάτευσης είναι ο μηχανισμός επίλυση ε, διαφορών. Υπάρχει μια διαφορά στην εστίαση. Εμείς θεωρούμε ότι πράγματι ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, εστιάσει κάποια θέματα, θεωρεί σημαντικά. Θα δούμε ε, τα καινοτόμα στοιχεία, αν μπορούμε να αντιοθετήσουμε. Μπορεί να έχουμε αμφιβολίες για ένα σύστημα που δεν θεωρούμε ότι έχει δοκιμαστεί ως αποτελεσματικό. Υπάρχουν κάποια που μπορούμε, που μπορούμε να τα διασώσουμε για να καταλήξουμε σε συμφωνία. Τώρα κάποια θέματα που συζητούνται δεν θέλω να εστιάσω γιατί τα είπε και ο προλαλή σα. Έχουμε τις γραφικές σε ένα πρόβλημα εδώ. είναι ένα σημαντικό για εμάς ε, ζήτημα, κανόνες προέλευση, το γενομική κανόνες και αυτό είναι σημαντικό. Αλλά η βασική ανησυχία του Μεξικού είναι πρόσβαση στην αγορά αγαθών. Πολλά είναι ακόμη. Αυτά πρέπει να γίνουν για να βρούμε τις ισορροπίες που θέλουμε και να ευοδοθεί τελικά αυτή η συμφωνία σύνδεσης μεταξύ Ευρωξένου και Μεξικού. Ευχαριστώ. Gracias. Um, Σας ευχαριστώ. Μπορούμε να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση για το θέμα αυτό, για τον εξοχρονισμό της Συμφωνίας Εμπορίου με το Μεξικό. Σας ευχαριστώ όλους. ήταν το θέμα πολύ ενδιαφέρον, αλλά τώρα θα περάσουμε στο σημείο 8 της ημερής της διάταξης της ψηφοφορίας. Ξεκινώντας από το ψήφισμα για την 11η Υπουργική Σύνοδο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, θα ήθελα πριν ξεκινήσουμε την ψηφοφορία να κάνουμε έναν έλεγχο του ηλεκτρονικού συστήματος ψηφοφορίας. Ψηφίστε παρακαλώ. And του ελέγχου της ψηφοφορίας. Ψηφίσατε υπέρ. Κάτω πλειοψηφία στον έλεγχο. Ωραία. Εντάξει, λειτουργεί το σύστημα. Να ελέγξουμε λίγο την εκπροσώπηση των ομάδων. Είναι σωστός ο αριθμός των βουλευτών. Επομένως μπορούμε να ξεκινήσουμε. Συμβαστική 1 υπέρ Κατά. αποχέ, Εγκρίνεται. Ε, τροπολογία 14 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 15 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 2 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 23 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβεβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 28 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβιβαστική 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 34 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 5 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 38 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 39 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 40 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 41 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Σαράντα δύο υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Σαράντα τρία υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Σαράντα τέσσερα υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Σαράντα πέντε υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 46 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβιβαστική 6 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 7 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 56 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 57 υπέρ, κατά,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 αποχές εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία, ε, ηλεκτρονική ψηφοφορία της, ε, του ψηφίσματος όπως τροποποιήθηκε. Ψηφίστε παρακαλώ. The vote is closed. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται. Δίνουμε λοιπόν εντολή για την προσώπησή μας στο Υπουργικό Συμβούλιο. Σημείο 9 της ημερήσιας διάταξης, μία ψηφοφορία ηλεκτρονική για το προφορικό ερώτημα για τον IMC. Ε, ψηφίστε παρακαλώ. And the ψηφοφορία. Ομόφωνα εγκρίνεται. και ολοκληρώσαμε τις ψηφοφορίες. Σας ευχαριστώ πολύ και θα περάσω στο σημείο 10 της της διάταξης. Εξελίξεις στις διαπραγματεύσεις στον τριμερή διάλογο. Ε, μόνο ένα είναι ο τρίμερη διάλογο που έχουμε ανοιχτό αυτή τη στιγμή. Είναι ότι ε, ο ξεχρονισμό του TDI έγινε μια συνάντηση την προηγούμενη εβδομάδα, 7 Νοεμβρίου παραμένουν σημαντικά ζητήματα ανοιχτά. Πρώτα απ' όλα το lesser duty rule, ο κανόνας για τον ελάχιστο δασμό. Η συμπερίληψη προτύπων περιβαλλοντικών και ε, εργασιακών στις και άλλα θέματα. Άρα χρειάζεται ακόμα αρκετή διαπραγμάτευση. Έχει υπάρξει συμφωνία σε ορισμένα ζητήματα τεχνικού χαρακτήρα και θα οργανώσουμε σύντομα τις επόμενες ε, συναντήσεις τεχνικού χαρακτήρα για να μπορέσουμε στις 27 Νοεμβρίου να κάνουμε την επόμενη συνάντηση του τριμερή διάλογο. Πάμε στο σημείο 11. Εδώ έχουμε την παρουσίαση μιας μελέτης. Τρέχουσες και ε, νέες τάσεις στις τεχνολογίες που δημιουργούν μεγάλες αλλαγές, disruptive technologies, και τι επιπτώσεις θα έχει αυτό για την σημερινή και μελλοντική πολιτική εμπορίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα δώσω το λόγο στον δόκτωρο ε, ε, Μπούρη από το Πανεπιστήμιο της Λουκέρνης. Είναι διευθύντη του Κέντρου Διεθνούς Δικαίου και συντάκτρια της ε, έκθεσης. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ και που μου δίνετε την ευκαιρία να παρουσιάσω την έκθεση αυτή για τις εξελίξεις στην τεχνολογία που επιφέρει ανατροπές και τις επιπτώσεις που θα έχουν αυτές οι ανατροπές στην πολιτική εμπορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης μελέτη χωρίζεται σε τρία, τρεις ενότητες. Πρώτα απ' όλα ποιες είναι αυτές οι ανατρεπτικές τεχνολογίες και τι ακριβώς αντίκτυπο έχουν. Πρόκειται για ψηφιακές τεχνολογίες, κατά κύριο λόγο. Δεύτερος σκοπός της έκθεσης είναι να ε, εξετάσουμε το διεθνές εμπορικό δίκαιο και την εξυγχρονισμό του, τις αλλαγές που έχουν υπάρξει μετά τις διάφορες διεθνείς συμφωνίες και τις αλλαγές που αυτές επέφεραν, γιατί πολλές από αυτές τις αλλαγές ε, επήλθαν ακριβώς εξαιτία των της εξελίξεων στην ψηφιακή τεχνολογία και το τρίτο μέρος της έκθεσης εστιάζει στο πώς μπορεί να μεταβληθεί και να προσαρμοστεί η πολιτική εμπορίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης έτσι ώστε να ενισχύσει η Ένωση τη θέση της στο, στην παγκόσμια οικονομία και αξιοποιώντας τη δυνατότητά της να ε, καινοτομεί. Θα προσπαθήσω να παρουσιάσω και τα τρία θέματα αυτά με αυτή τη σειρά. Το πρώτο ερώτημα λοιπόν, τι είναι αυτές οι ανατρεπτικές τεχνολογίες. Πολλοί θα έλεγαν ότι είναι απλώς μια νέα μόδα να χρησιμοποιούμε αυτή την έκφραση ε, και να καλύπτουμε με αυτή την έκφραση πολλά φαινόμενα. Αυτό ισχύει. Ε, Ακούμε ορισμένους να αναφέρονται στην, στον ψηφιακό μεταχειρισματισμό, στην τέταρτη βιομηχανική επανάσταξη. Ε, πολλές φορές στο πλαίσιο αυτών των συζητήσεων γίνονται αναφορές στην τεχνική, τεχνητή νοημοσύνη. Γενικά μιλούμε πάντως για τεχνολογίες οι οποίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε πολύ μεγάλες κοινωνικές αλλαγές, να ανατρέψουν τα δεδομένα. Και Υπό αυτή την έννοια είναι σημαντικό να αντιληφθούμε ότι ως ε, ρυθμιστές του, του, του, του, τρόπου με τον οποίο διεξάγονται οι εμπορικέ συναλλαγέ, οι τεχνολογίες αυτές μπορούν να φέρουν, μεγάλες να φέρουν μεγάλες αλλαγέ. Στι τεχνολογίε αυτέ θα συμπεριλάμβανα την τρισδιάστατη εκτύπωση της εξέλιξη στο ίντερνετ, στην κινητή τηλεφωνία, τη μεταφορά μεγάλων όγκων δεδομένων, την ανάλυση τους. Οικονομολόγοι σήμερα λένε ότι τα δεδομένα έχουν γίνει το πιο σημαντικό οικονομικός πόρος, γιατί είναι πλέον στο ίδιο επίπεδο με τις πρώτες ύλες και το ανθρώπινο δυναμικό σε μια παραγωγή. Και δεν αναφέρομαι μόνο στις ε, εταιρείε πληροφορική, αυτά που σκέφτεται κανεί αμέσω σκεπτόμενο τι εταιρείε μηχανών αναζήτηση ή τα κοινωνικά μέσα δικτύωση, αλλά την χρήση δεδομένων ακόμα και σε πιο συμβατικέ μορφέ παραγωγή ή επιχειρήσει. Διαπιστώνουμε ε, επιπτώσεις αυτών των αλλαγών στην πολιτική εμπορίου. Πρώτα απ' όλα είναι η ανάπτυξη που επέρχεται εξαιτία τη ψηφιοποίηση. Το δεύτερον είναι ότι το περίπου 50% των υπηρεσιών που ε, εμπορεύονται στον κόσμο, που ε, αποτελούν αντικείμενο εμπορικών συναλλαγών, είναι ήδη ψηφιακές οι ροέ δεδομένων σε παγκόσμιο επίπεδο είναι και ένα μέσο πολέμηση του αποκλεισμού υπό την έννοια ότι μικρότερε χώρε οι μικρότερε επιχειρήσει μπορούν να βρουν και αυτέ τη θέση του στο παγκόσμιο εμπόριο. Ταυτόχρονα όμω, ε, σε αυτές τις νέες ε, ψηφιακές αγορές ε, βλέπουμε όλο και μεγαλύτερη συγκέντρωση, δημιουργία συγκεντρωτικών δικτύων και καταστάσεις στις οποίες τελικά μία επιχείρηση επικρατεί. Στο γράφημα αυτό βλέπετε την σχέση των υπηρεσιών αυτών ως προς τον πληθυσμό της κάθε χώρας. Σίγουρα έχετε ακούσει ορισμένες από αυτές τις φράσεις, παγκόσμια εφοδιαστική λυσίδα, η μεταβολή, το πέρασμα προς την παροχή υπηρεσιών, οι διασυνοριακές ροές δεδομένων, δεν θα σταθώ σε κάθε, πω, σε κάθε μια από αυτές τις έννοιες, όμως αυτό που θέλω να πω είναι ότι αυτές οι εξελίξεις έχουν σημασία για, την, για το παγκόσμιο εμπόριο. Το γεγονό ότι όλο και περισσότερο χρησιμοποιούμε ε, υπηρεσίες, ε, εφαρμογές, ε, σημαίνει ότι τα δεδομένα πρέπει να μετακινούνται διασυνοριακά όρο και περισσότερο. Και αυτό δημιουργεί πολλά σημαντικά και δύσκολα ερωτήματα για εμάς. Μπορεί κανείς να, να αξιοποιήσει αυτές τις προές για σημαντικά οικονομικά ωφέλη. Ε, βλέπετε εδώ πώς το έχουν αξιοποιήσει αυτό οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως, τίθενται επίσης και ζητήματα ε, σημαντικά για το ρυθμιστικό πλαίσιο που θα έχουμε για να προστατεύεται η ιδιωτικότητα, να προστατεύεται η εθνική ασφάλεια, και δεν θα λέγαμε ότι όλες οι οικονομίες, όλα τα κράτη σε ολόκληρο τον κόσμο έχουν ανοίξει τα σύνορά τους σε αυτές τις διασυνοριακές ροές συγγνώμη, δεδομένων. Αντιθέτως, ε, βλέπουμε τα τελευταία χρόνια να υψώνονται όλο και περισσότερα εμπόδια. Ε, πρώτα απ' όλα, ε, ένα προφανές μέτρο είναι τα μέτρα που λαμβάνονται για την παροχή ψηφιακών υπηρεσιών μόνο τοπικά, με κάποιους τοπικούς περιορισμούς ανάλογα με το που βρίσκεται ο πάροχος της υπηρεσίας. Ε, ε, κάποιες χώρες ζητούν να βρίσκεται σε μια συγκεκριμένη χώρα στη δικιά τους επικράτεια για να μπορούν να τον ελέγξουν νομικά. Επίσης, θα έρθω τώρα στο σχέδιο της παρουσίασης που αφορά στο πώς έχει ε, εξελιχθεί η πολιτική εμπορίου για να ανταποκριθεί σε αυτές τις ψηφιακές αλλαγές. Βεβαίω το διεθνέ εμπορικό δίκαιο έχει σημασία, έχει, επηρεάζει τις μεταφορές ε, δεδομένων γιατί ε, ρυθμίζει όλα τα επίπεδα του ίντερνετ από τις υποδομές ε, μέχρι την παροχή των υπηρεσιών αυτών. Πάντοτε οι εξελίξεις στο διεθνές εμπορικό δίκαιο ξεκινούν με πολυμερείς συμφωνίες και χωρίς να πω σε λεπτομέρειες πιστεύω ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου είναι, έχει, πολύ μεγάλο, έχει ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα. Είναι ένας οργανισμός ο οποίος βασίζεται σε κανόνες, ο οποίος έχει αποδείξει τη σταθερότητά του, στην οποία ε, εκπροσωπούνται πάρα πολλές χώρες και ο οποίος καταφέρνει να έχει αποτελέσματα εφόσον υπάρχει πολιτική βούληση βέβαια. Ωστόσο, πρέπει να ε, δεχτούμε, πρέπει να δούμε ότι ο ΠΟΕ δεν έχει καταφέρει να ανταποκριθεί επαρκώς στην ψηφιακή αλλαγή. Ούτε να σταματήσει πρακτικές ε, forum shopping, επιλογής του πιο ευνοϊκού ρυθμιστικού πλαισίου. Ούτε ε, οι μεγάλες διεθνείς εμπορικές συμφωνίες έχουν καταφέρει να το αντιμετωπίσουν. Οι αλλαγές έχουν προέρθει σε μεγάλο βαθμό από τις Ηνωμένε Πολιτείε, οι οποίες στο πλαίσιο της ψηφιακή ε, ατζέντα που, που υιοθέτησαν το 2002 έχουν επιβάλει το μοντέλο τους όσον αφορά τη ρύθμιση του ψηφιακού εμπορίου. Μπορεί να το διαπιστώσει κανείς αυτό εξετάζοντας ε, τις, ε, τα, τα κεφάλαια που αφορούν στα πνευματικά δικαιώματα, στις υπηρεσίες ε, ή το, ή το ηλεκτρονικό εμπόριο των διαφορών συμφωνιών. Όλες και, όλο και περισσότερες από αυτές τις συμφωνίες έχουν πλέον ένα ξεχωριστό κεφάλαιο για το ηλεκτρονικό εμπόριο. Και στο πλαίσιο των συμφωνιών που συνάπτονται εντός του ΠΟΕ ε, καλύπτονται όλο και περισσότερα αυτά τα ζητήματα και δημιουργούν νέες ε, διατάξεις στο, στο, στο δίκαιο. Βλέπουμε επίσης όλο και μεγαλύτερη ρύθμιση των ροών δεδομένων στις ε, διεθνείς εμπορικές συμφωνίες. Εδώ η το, το σημαντικότερη ρύθμιση που έχουμε στα χέρια μας είναι αυτή που προβλέπεται στην TPP, όπου προβλέπεται ξεκάθαρα η απαγόρευση του να ε, τίθενται εμπόδια στις, ροές, ε, εμπόδια στις ροές δεδομένων. Και απορρίπτονται ρητά μέτρα που επιβάλλουν την τοποθέτηση του σερβερ σε μια συγκεκριμένη χώρα. Περάσαμε από το, τη ε, ελαφρότερη προσέγγιση soft law των Ηνωμένων Πολιτειών που σας προανέφερα σε ρητές διατάξεις. Ο στόχος αυτών των ρυθμιστικών πρωτοβουλειών δεν οδηγεί πάντα σε αύξηση ε, της αυστηρότητας των προτύπων. Αντιθέτως, όσον αφορά την προστασία προσωπικών δεδομένων, υπάρχει υποχώρηση. Θα λέγαμε ότι ε, δίνουμε μεγαλύτερη έμφαση στο, στο να λειτουργεί το εμπόριο παρά στην προστασία των προσωπικών δεδομένων και άλλωστε είναι και θέμα το οποίο ε, απασχόλησε τις ε, το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, λοιπόν, σε αυτό το περιβάλλον να σας πω τι βλέπουμε όσον αφορά και την εξέλιξη των συμφωνιών ε, ελεύθερου εμπορίου. Από τη μία πλευρά, όσον αφορά τους κανόνες, ας πούμε, βλέπουμε ότι το ψηφιακό εμπόριο έχει ένα νέο καθεστώς ε, το οποίο το διέπει και δεν αφορά μονάχα την πρόσβαση αγοράς, αφορά περισσότερο ε, την, ε, τη διασύνδεση των εσωτερικών ε, ε, ημεδαπών καθεστώτων έτσι ώστε να προκύψει βεβαιότης για τις επιχειρήσεις αυτές οι οποίες δρούν στην αγορά. Σημαντικό είναι να αναφερθεί εδώ ο τρόπος με τον οποίο το μοντέλο των ΗΠΑ έχει διαχυθεί. Το template των ΗΠΑ είναι το πλέον δεσπόζων στις Ηνωμένες Πολιτείες φυσικά, αλλά, ε, στη συμφωνία δηλαδή με τις Ηνωμένες αλλά έχει μεταφερθεί ε, και σε άλλες συμφωνίες όπως ας πούμε με την συμφωνία. Στην ουσία έχουν κάνει copy-paste, αντιγραφή και επικόλληση. Ε, στις άλλες συμφωνίες. Ποια είναι η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης λοιπόν σε αυτό το νέο περιβάλλον. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε ιδιαίτερα καινοτόμα ε, ε, προσέγγιση όσον αφορά ε, την ψηφιοποίηση λοιπά, Δεν βρέθηκε στην εξωτερική πολιτική, στην πολιτική εξωτερικού εμπορίου, δεν βρέθηκε ακριβώς αυτή η αντιστοίχηση. Έχουμε δει βεβαίως εξέλιξη από τις πρώιμες ε, συμφωνίες μέχρι τη ΣΥΤΑ και την ε, ΤΑΛΑ. Παρ' ε, παρόλα αυτά εξακολουθεί να υπάρχει μια γενική τάση που είναι παρόμοια και βάσει της μελέτης προκύπτει ότι ενδεχομένως υπάρχει ανάγκη προσαρμογής, καλύτερης στοχοθέτησης της ψηφιακής οικονομίας και τις θέσεις που ε, μπορεί να έχει στις συμφωνίες ε, αυτές. Ε, σύμφωνα με την μελέτη μπορούν να γίνουν και κάποιες συστάσεις, ορισμένες μερικέ, περισσότερο γενικού χαρακτήρα, διαθεσμική συμφωνία, διοργανική συμμετοχή κτλ. Αλλά υπάρχουν και κάποιες συστάσεις οι οποίες είναι πολύ συγκεκριμένες. Εγώ θα ήθελα να αναφερθώ κυρίως στην σύσταση υπαριθμών 3 η οποία πραγματικά μπορεί να δώσει κίνητρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση να πάρει μια προενεργητική θέση έτσι ώστε να δημιουργηθούν αυτές οι προϋποθέσεις ε, οι οποίες ε, θα εφαρμόσουν λοιπόν όλα τα στοιχεία της ψηφιακή πολιτικής και στις συμφωνίες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό μπορεί να γίνει μέσα από πολυτομιακή στρατηγική να προωθηθούν δηλαδή τα, οι στόχοι αυτοί και στα πλαίσια του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου αλλά όχι μόνο ε, μέσω όλων των συμφωνιών ελεύθερου εμπορίου μέσα από μια σωστή και καλή αλληλουχία της στρατηγικής ε, γιατί μέσα από αυτή τη σωστή αλληλουχία τελικά ε, φτάνουμε σε ένα καλό αποτέλεσμα όσον αφορά τις τηλεπικοινωνίες και όσον αφορά τον τομέα των διανοητικών δικαιωμάτων, διανοητικής ιδιοκτησίας κτλ. Και εκεί βλέπουμε ότι συγκλίνουν και τα templates και υπάρχει και σαν δεύτερο βήμα κάτι το οποίο μπορεί να ληφθεί υπόψη ε, το ε, ε, μορατόριο όσον αφορά την ηλεκτρονική μετάδοση, την γλώσσα όσον αφορά την ουδετερότητα του δικτύου και όσον αφορά την λογοκρισία. Και τέλος, όσον αφορά την ενδιάμεση υποχρέωση ε, όσον αφορά τα διανοητικά δικαιώματα. Όλα αυτά βεβαίως μπορεί να είναι αποτελεσματικά μονάχα εάν ε, συνοδεύονται από τα βασικά χαρακτηριστικά τα οποία θα διασφαλίζουν, τα οποία υπάρχουν ήδη στην ενωσιακή νομοθεσία και τα οποία διασφαλίζουν ακριβώς την ασφάλεια, αποτελούν εχέγγυο για την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας ευχαριστώ πολύ. Εμείς σας ευχαριστούμε, λέει ο Πρόεδρος. Πάρα πολύ ενδιαφέροντα αυτά που μας είπατε. Uh, και ευχαριστούμε ιδιαίτερως και για τις συστάσεις που κάνετε. Αλλά πολλή δουλειά, πολλή δουλειά προϋποθέτουν όλα αυτά που μας λέτε. Υπάρχουν συγκεκριμένες ερωτήσεις. Χάιντι παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω αγαπητή κυρία για την ε, μελέτη η οποία ξεκαθαρίζει λίγο το τοπίο και τις ε, προοπτικές για την καλύτερη δυνατή προώθηση αυτών των ε, συμφωνιών. Έχω συγκεκριμένες ερωτήσεις. Πιστεύετε ότι ήρθε η ώρα να προχωρήσουν οι διαπραγματεύσεις ε, για το ε, ηλεκτρονικό εμπόριο με, με τη Διεθνή Οργάνωση Εμπορίου. Τώρα ολοκληρώνεται και η εντολή. Δεύτερη ερώτηση. Τι θα γίνει με την διανοητική ιδιοκτησία που περιλαμβάνει και την ε, ενωσιακή νομοθεσία για το copyright. Πιστεύετε ότι μπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο. Δηλαδή μήπως το copyright παρισφρήσει ε, στο ψηφιακό εμπόριο δημιουργώντας υπερβολική νομοθεσία όσον αφορά το εμπορικό ε, κομμάτι ε, δηλαδή δεν ξέρω ακριβώς πώς να σας το πω αλλά ε, πώς θα πρέπει να λάβουν υπόψη το copyright οι συνομοθέτες. Τρίτον, προστασία προσωπικών δεδομένων και ιδιωτικής ζωής η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα μπορούσε εδώ να θέσει ε, τα διεθνή πρότυπα, τα global standards μια και έχει ένα υψηλό ε, επίπεδο ε, προστασίας δεδομένων και ιδιωτική ζωή σε βάση του σχετικού κανονισμού που έχουμε εγκρίνει. Αυτή είναι η εντύπωση τουλάχιστον που έχω. Η κυρία Ζαμέ. Κοιτάξτε, εγώ δεν έχω τον ίδιο ενθουσιασμό όταν ακούω τέτοια πράγματα γιατί θεωρώ ότι ε, ε, ε, πίσω από μια μεγάλη προστασία ας πούμε της προώθησης του ψηφιακού εμπορίου τελικά βλέπω να κρύβονται επιθετικές πολιτικές όσον αφορά ειδικέ δεσμεύσεις ή ειδικέ αρμοδιότητες των κρατών μελών ας πούμε για μέτρα διακριτικά, για την προώθηση της τοπικής πολιτικής κτλ. Επίσης υπάρχουν και κάποιες έννοιες οι οποίες είναι ασαφείς και στις οποίες μπορεί να δοθούν αμφιλεγόμενες ε, ε, ερμηνείες. Λέμε ότι ε, οι εμπορικές συμφωνίες άρουν ε, έχουν μάλλον την τάση να ε, κάνουν πιο υψηλό το επίπεδο προστασίας ενώ ταυτοχρόνως παρακάτω λέμε ότι θα πρέπει να αρθούν οι προστατευτικές πολιτικές. Ε, ωραία είναι όλα αυτά, αλλά νομίζω ότι δεν μπορώ να συμφωνήσω με κάποιες ε, κρίσεις ουσία, ε, ουσίας αξίας τις οποίες αναφέρετε και οι οποίες μάλλον προκύπτουν από την προσωπική σφαίρα. Τώρα, ναι, να συζητήσουμε με, το Διεθνό Οργανισμό Εμπορίου, ναι, αλλά δεν είναι μόνο εκεί το πρόβλημα πιστεύω ότι τα κράτη, τα κράτη έχουν δικαιώματα, έχουν δικαίωμα και καθήκον μάλιστα να προστατεύσουν τις επιχειρήσεις τους απέναντι σε ε, παγκόσμιους ε, γίγαντες. Υπάρχει ο οικονομικός ε, πόλεμος στον οποίο πολύ συχνά πηγαίνουμε χωρίς όπλα και πιστεύω ότι και οι πολίτες ενδιαφέρονται πάρα πολύ να συζητήσουν το θέμα αυτό τη στιγμή που έχουμε μια τεράστια έκρηξη του κυβερνοεγκλήματος ε, και τις κυβερνοεγκληματικότητας τη στιγμή που έχουμε ένα τεράστιο κύκλωμα παραχάραξης, ε, πλαστογράφησης ε, φαρμάκων κλπ. Επίσης, έλεγχος κυκλοφορίας των δεδομένων και γεω εντοπισμός. Αυτά όλα είναι ένα συνοθήλευμα το οποίο δημιουργούν μία λίγο ασαφή κατάσταση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Κοιτάξτε εδώ, μιλάμε για δικαιώματα, για ελευθερίες των ε, πολιτών των κρατών μελών. μιλάμε ε, για κρυπτογραφημένες ε, πληροφορίες. Εγώ πιστεύω ότι κάθε κράτος θα οφείλει να έχει κυριαρχία όσον αφορά και έλεγχο όσον αφορά την κυκλοφορία των στοιχείων αυτών. Πρόεδρος, τις συστάσεις σας ίσως πρέπει να αναφέρεται και το θέμα της προστασίας των καταναλωτών. Έχω την αίσθηση ότι λείπει αυτή η αναφορά, δεν ξέρω. Όταν μιλάμε για ελεύθερη διασυνοριακή κυκλοφορία αγαθών, υπηρεσιών, η προστασία των καταναλωτών είναι κάτι πάρα πολύ σημαντική. Τουλάχιστον ε, θα πρέπει να είναι η ίδια προστασία όπως κάναμε και για την ε, αντίστοιχη προστασία στην ε, εσωτερική ψηφιακή αγορά. Αυτό ήταν η πρώτη μου παρατήρηση. Δεύτερον, ε, ε, Ίσως αυτό το θέμα της ουδετερότητας. Ε, εδώ ίσως θα πρέπει να δούμε και την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για τις ε, πλατφόρμες και τους παρόχους Uh, Σας ευχαριστώ πολύ για τις πολύ ενδιαφέρουσες ε, ερωτήσεις. Όλες ε, πολύ εύστοχες. Θα προσπαθήσω να απαντήσω. Πρώτον, σε ό,τι αφορά το ΟΠΟΕ, νομίζω ότι από νομικής πλευράς ο ΠΟΕ ε, παρέχει δυνατότητες για την αντιμετώπιση των ζητημάτων που άπτονται του ψηφιακού εμπορίου. Απλά μέχρι στιγμής δεν υπήρχε πολιτική βούληση για να συμφωνήσουμε παρκώς πώς θα προχωρήσουμε σε αυτά τα ζητήματα. Πολλά από το πρόγραμμα ηλεκτρονικό εμπόριο του ΠΟΕ δυστυχώς έχουν ε, σταματήσει τα κράτη-μέλη του ΠΟΕ από το να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες. Γίνεται λόγος παραδείγματος ακόμη για την ταξινόμηση των υπηρεσιών, τι θα πει η υπηρεσία, τι θα πει αγαθό, και όλα αυτά τα θέματα είναι σημαντικά μεν. Μπορούμε όμως με τον νέο νομικό σχεδιασμό να προχωρήσουμε δε και να δούμε τα πιο επίγοντα σύγχρονα ζητήματα και να προχωρήσουμε. Και υπάρχουν πολλοί τρόποι να γίνει αυτό. Έχει κάνει μια ενδιαφέρουσα πρόταση η Κομισιόν για τη συμβάση με ηλεκτρονική υπογραφή προστασία καταναλωτών αλλά το κατόφλι είναι χαμηλό σχετικά και δεν υπάρχει δέσμευση για τα σημαντικά ζητήματα. Η Ένωση νομίζω ότι μπορεί να προχωρήσει προς τα εμπρός. Ίσως ε, στηριζόμενοι αρχές ε, του ηλεκτρονικού εμπορίου του 2011 ε, και να προσπαθήσει να αποσπάσει κάποιες δεσμεύσεις από τα κράτη-μέλη του ΠΟΕ. με οριζόντια δεσμεύσεις, παραδείγματο χάρη, σε ό,τι αφορά το ΚΑΤ και συγκεκριμένες δεσμεύσεις. Μπορούν να υπάρχουν όσο πλέον, επιπλέον δεσμεύσεις, ε, κάποια reference papers. Και στο άρθρο 18 του ΓΚΑΤ λέγεται θα μπορούσε να υπάρχει μία πολυμερή συμφωνία που θα είναι δεσμευτική για τους ε, υπογράφοντες στη συμφωνία, αλλά μπορεί να είναι και ανοιχτή συμφωνία και να έχει έτσι μια κρίσιμη μάζα μελών του ΠΟΕ για να αντιμετωπίσει ε, σημαντικά ζητήματα από το ψηφιακό εμπορίο. Αυτά σε ό,τι αφορά τον ΠΟΕ. Σε ό,τι αφορά το copyright. Δεν είμαι ξεκάθαρη. Γιατί ο στόχος μου δεν είναι τόσο το να πάρω μέρος, να προτιμήσω κάποιο στρατόπεδο. Οι αναπτύ εξελίξεις ε, μας κάνουν να θέλουμε να επιβάλλουμε υψηλά πρότυπα και για το ψηφιακό copyright, αλλά ίσως να πηγαίνουμε πολύ μακριά. Σε ό,τι αφορά τα πνευματικά δικαιώματα, σε ό,τι αφορά τη κυβέρνηση του εμπορίου και τα templates τα οποία θα ε, διαμοιραστούν στις διάφορες συμφωνίες. Εκεί η μορφή είναι λιγότερη. Οι ΙΠΑ κάνουν λίγο πολύ τα ίδια με τις ε, χώρες της Ένωσης. Το ψηφιακό copyright ε, εντάσσεται. Έχουμε και τα θέματα ευθύνη των παρόχων διεκτικού περιεχομένου που θα είναι ένα σημαντικό ζήτημα. Και η Κομισιόν, μάλλον η Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει να φροντίζει οι συμφωνίε συμφώνονται και στρατηγική ψηφιακή αγορά. Ένα σημείο απόκλησης, για παράδειγμα, έχει να κάνει τα δικαιώματα των εκδοτών. Σε αυτά τα Αυτό δεν αντιμετωπίζεται μέχρι στιγμής σε κάποια, εμπορία, ε, σε συμφωνία ελεύθερου εμπορίου. Προστασία δεδομένων και προστασία ιδιωτικότητας. Εγώ νομίζω ότι έχουμε θετικές εξελίξεις. Υπάρχουν κάποιες μελέτες της ΕΠΑ που δείχνουν ότι ναι μεν το νομικό πλαίσιο δεν αλλάζει, αλλά πολλές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις ψηφιακές αγορές και θέλουν να έχουν και ευρωπαϊκή παρουσία, ήδη προβαίνουν σε αλλαγές ενδοτερικά για την προστασία των δεδομένων. Νομικά βέβαια αυτό θα έπρεπε να κατοχυρωθεί ε, το υψηλό επίπεδο νομικής προστασίας το δεδομένο Να υπάρχει μεγαλύτερη μάλλον η Κομισιόν να εγκρίνει κάποιες αποφάσεις ε, καταλληλότητας επάρκειας. Υπάρχει επίσης μια πρόταση για τη σύμβαση, για μια σύμβαση ό,τι αφορά το καθεστώς δεδομένων και άλλα εξωτικά. Ε, μπορούμε να τα δούμε. Θα ξαναβάλω το καπέλο του πανεπιστημιακού και εντάξει μπορεί να έχω επιθετική προσέγγιση σε κάποια ή να θεωρηθούν ε, οι προσεγγιση μου επιθετικές σε κάποια ζητήματα. Δεν ήταν στόχος αυτός όταν συνέγραψα το πόνημά μου. Νομίζω ότι υπάρχουν πολύ καλοί λόγοι για να προστατεύσουμε την, ε, τα δεδομένα και για να τα εντοπίσουμε κάπου σε κάποιο συγκεκριμένο σημείο. Άλλο προστασία και άλλο προστατευτισμό δεδομένων. Μπορούμε να βάλουμε τη διαχωριστική γραμμή. Σε ό,τι αφορά τον νομικό σχεδιασμό, νομίζω ότι αυτό μπορεί να γίνει με εξαιρέσεις. Είτε για συγκεκριμένους σκοπούς, είτε γενικές εξαιρέσεις όπως στο άρθρο 14 του Ίσως είναι λίγο περιοριστικό βέβαια αυτό το άρθρο, αλλά στην TPP για πρώτη φορά το ενδιαφέρον είναι ότι έχουμε ένα πείραμα, δηλαδή για τις εξαιρέσεις. Θα μπορούσαν τα μέτρα εντοπισμού να απαγορεύονται ή ελεύθερη ροή δεδομένων για θεμητούς σκοπούς. Βέβαια δεν καταγράφονται κάπου αυτοί οι στόχοι, αυτή η σκοπή, είναι λίγο ανοιχτό το πεδίο. Αλλά βλέπουμε να αλλάζει λίγο και η γλώσσα σε ό,τι αφορά το νομικό σχεδιασμό των συμφωνιών αυτών. Και εδώ νομίζω η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να κάνει και ένα βήμα παραπάνω. Για τα αντισταθμίσματα αυτά, ναι, είναι σημαντικά και πρέπει να εξευρεθεί ισορροπία μεταξύ της προστασίας ιδιωτικών των πολιτών, της εθνικής ασφάλειας και άλλων ζητημάτων αλλά όχι προστατευτισμός. Δεν είναι η σωστή λύση. Και αν δει κανείς και οικονομικά την πρόσβαση αγορές, ε, την ε, θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης αγορές ως μια ανταγωνιστική δύναμη, καινοτόμος δύναμη. Είναι αποφάσεις ε, που πρέπει να ληφθούν. Συμφωνώ για την προστασία των καταναλωτών ότι λείπει. Θα το προσθέσω. Η εμπιστοσύνη των καταναλωτών είναι κομβική σημασία για την εύρυθμη λειτουργία αυτών των αγορών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ μπορεί να συντεριάσει αυτά που κάνει σε ε, εσωτερικό επίπεδο και στην εξωτερική πολιτική, την εμπορική. Ουδετερότητα δικτύου το ανέφερα αλλά με μια λέξη, ότι TPP έχουμε τα πρότυπα για την τέλο του δικτύου, αλλά είναι ασαφώς διατυπωμένα. Καλό θα ήταν οι κανόνες να ενδυναμωθούν και να βάλουμε, να, μπούμε εμείς, να γίνουμε εμείς το παράδειγμα ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόεδρο, σας ευχαριστώ. Πολύ επικοδομητική και μελέτη σας και η συζήτηση. Να περάσουμε τώρα στο επόμενο σημείο της μερικής διάταξης. Αντίδραση, ανταπόκριση σε αυτή την πρόκληση. Για τη στρατηγική για το ψηφιακό εμπόριο. Η Μαρίτσα Σάτια έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν ξέρω αν είναι η αντίδραση που έχουμε αμέσως στο θέμα αυτό, αλλά είναι ε, μια πρώτα, πρώτη προσέγγιση ε, έχει ενδιαφέρον γιατί τώρα θα μιλήσω για θέματα τα οποία σχεδόν τα κάλυψε όλα η προλαλήσα ομιλήτρια με αυτή τη ε, μελέτη και θα ήθελα να σας ρωτήσω πώς σκοπεύουμε να οργανώσουμε τη συζήτηση. Εν πάση περιπτώσει, ε, για να δούμε διαδικαστικά πώς θα μπορούσε να γίνει αυτό. Πάντως ήθελα να εκδηλώσω το ενδιαφέρον μου. Ο στόχος της παρουσίασης μου είναι να σας ενημερώσω για τις εξελίξεις που είχαμε στην προσπάθεια να καταρτιστεί μια ευρωπαϊκή στρατηγική για το ψηφιακό εμπόριο. Να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα όλους όσοι συμμετείχαν και υπέβαλαν τροπολογίες. Έχουμε επίσης ε, ε, γνωμοδοτήσεις από άλλες επιτροπές του Κοινοβουλίου, Ήτρε, Λίμπε. Και το προσχέδιο μου βασίζεται σε τρεις πυλώνες. Πρώτα απ' όλα η πρόσβαση στην αγορά, σε σε τρίτες χώρες και πώς θα εξαλείψουμε τους φραγμούς. Το δεύτερο είναι πώς οι κανόνες θα έχουν ε, αποτελέσματα απτά για τους κατανοητές και τρίτον η προώθηση των ψηφιακών δικαιωμάτων μέσω των συμφωνιών ελευθέρων εμπορίου. Ένα ζήτημα που το ανέδειξαν και άλλες συνάδελφοι. Από τις διάφορες τροπολογίες προκύπτουν τα εξής. Ε, κάποια συμπεράσματα μάλλον τα, τα οποία προσπάθησαν να αποκρισταλώσουν στις συμβιβαστικές τροπολογίες τις οποίες θα συζητήσω με τους σκιώδεις. Πολλές τροπολογίες αναφέρονται στον ισότιμο ανταγωνισμό, στον δίκαιο ανταγωνισμό και πώς θα αντιμετωπίσουμε τις νέες μορφές προστατευτισμού στην ψηφιακή ε, οικονομία, πώς θα προστατεύσουμε τα δικαιώματα του καταναλωτή και θα αποφύγουμε τη δημιουργία μονοπωλιακών καταστάσεων. Δεύτερον, πώς θα αποφύγουμε επαχθείς διαδικασίες ε, που δημιουργούν προβλήματα και για στις επιχειρήσεις και στους καταναλωτές, ιδιαίτερα όταν μιλάμε για ψηφιακό εμπόριο. Μετά, ε, υπήρχαν πολλές τροπολογίες που ανέρικτεν τη σημασία της ψηφιοποίησης για την ανάπτυξη και το πώς τελικά θα ε, γεφυρώσουμε το ψηφιακό χάσμα αντί να το βαθύνουμε κι άλλο. Μετά ε, αναφέρθηκε η μεγάλη σημασία που έχει η ειδωτερότητα του δικτύου για να αναπτυχθεί το ψηφιακό εμπόριο και οι υπηρεσίες γενικά. Δηλαδή το γεγονό ότι η, ανάπτυξη, το, η όποια ανάπτυξη στις υποδομές δικτύου θα πρέπει ταυτόχρονα να, γνωρίζει την ε, ουδετερότητά του, δηλαδή το δικαίωμα κάθε χρήστη του δικτύου να έχει πρόσβαση ισότιμη σε κάθε μέρος του δικτύου. Ένα άλλο ζήτημα που αναδεικνύεται από του συναδέλφου είναι η σημασία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που θέλουμε να συνεχίσουν να είναι ατμομηχανικέ τη ψηφιακή οικονομία όπω υπήρξαν οι ατμομηχανοί τη παραδοσιακή οικονομία. Ένα άλλο σημαντικό θέμα είναι η καταπολέμηση της ανεργίας, η δημιουργία θέσεων εργασίας. Ε, αν θα μπορούσατε, Χάιντι, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι, έχει πολύ καλή δυστυχώς ακουστική αίθουσα και με ενοχλείται όταν ψιθυρίζετε. Το συγγνώμη, αλλά... Λοιπόν, ένα άλλο σημαντικό ε, θέμα μετά και από τα ειδήσει που ακούσαμε αυτή την εβδομάδα. Δηλαδή τώρα που μαθαίνουμε σιγά σιγά πώς χρησιμοποιούν τους φορολογικούς παραδείσους μέσω του Paradise Papers σε διάφορες εταιρείε ε, τεχνολογίας, υψηλής τεχνολογίας για να αποφεύγουν να πληρώσουν φόρους έχει μεγάλη σημασία να δούμε πώς θα καταπολεμήσουμε αυτές τις πρακτικές. Δεν συμφωνούν όλοι σε όλα και παραμένουν κάποια ανοιχτά ζητήματα. Για παράδειγμα, για τα πνευματικά δικαιώματα, σε ποιο βαθμό θέλουμε να τα προασπίσουμε και σε ποιο βαθμό θέλουμε σε αυτή την πρόσπιση να συμμετέχουν οι, οι μας. Είναι μια συζήτηση που την είχαμε και στο παρελθόν, αλλά ξανά έρχεται. Την είχαμε τη συζήτηση για την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων για τα αγαθά, τα, τα αντικείμενα. Ε, είχαμε σχετικές συζητήσεις όταν συζητούσαμε για τα φάρμακα θα πρέπει να δούμε ποιο είναι το κατάλληλο επίπεδο προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων αναλόγως με το εάν μιλάμε για ένα φυσικό προϊόν ή αν μιλάμε για μια υπηρεσία για να αποφύγουμε δυσμενείς επιπτώσεις από την υπερρύθμιση. Ένα άλλο θέμα είναι η, η προώθηση μάλλον της προστασίας ε, του καταναλωτή έναντι της αστικής ευθύνης που έχει ο ενδιάμεσος. Είναι ένα ζήτημα το οποίο αποσχολεί πολλούς πολίτες αλλά και μεγάλες επιχειρήσεις όπως για παράδειγμα το Google και η Facebook που αναρτιούνται ποιε είναι οι ευθύνε του για την προστασία των ε, πνευματικών δικαιωμάτων. Οποιοδεσδήποτε ρυθμίσεις όμως σε αυτόν τον τομέα θα έχουν σημαντικές επιπτώσεις και στην ελευθερία της έκφρασης online. Επομένω πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και ελπίζω ότι θα συνεργαστούμε καλά με τους χιώδεις στο θέμα αυτό. Και τέλος κάτι που είναι πολύ σημαντικό για τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο ψηφιακό ε, ε, εμπόριο είναι το θέμα της διασυνοριακή μεταφορά δεδομένων. Είχαμε πολλέ τροπολογίες από αυτού. Νομίζω ότι υπάρχει η συνένεση ως, το, ως, ως προς το ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αποκτήσει μια δικιά της θέση, μια δικιά της στρατηγική για το θέμα αυτό. Και να χρησιμοποιούμε τις εμπορικές συμφωνίες ε, ως ένα εργαλείο για να προστατεύουμε την εφαρμογή της ε, ενωσιακής νομοθεσίας που αφορά στην προστασία προσωπικών δεδομένων και την προστασία της ιδιωτικότητα. Και τα δύο είναι σημαντικά και η διασυνοριακή ροή δεδομένων και τα δικαιώματα των πολιτών και η ιδιωτικότητά τους και δεν θα πρέπει να υπερισχύει το ένα έναντι του άλλου. Ελπίζω να ε, συνεχίσουμε την καλή συνεργασία με τους κοιόδες και τους συναδέλφους έτσι ώστε ε, να γίνει ψηφοφορία τον Νοέμβριο, να εγκριθεί και από την Ολομέλεια πριν το τέλος της χρονιάς η έκθεση αυτή και να στείλουμε ένα σημαντικό μήνυμα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το πώς αντιμετωπίζουμε εμεί αυτά τα σημαντικά ζητήματα. Πράγματι, λέει ο πρόεδρος, το timing είναι εξαιρετικό. Θα δώσουμε το λόγο στου ασκιώδες ξεκινώντας από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Να ευχαριστήσω την εισηγήτρια και να σας ενημερώσω ότι αντικαθιστώ την κυρία Vivian Ρέντινγκ ε, και αναφέρομαι στις ιδέες πολλών συναδέλφων Πρέπει να, μην, να καλύψουμε το χαμένο έδαφο, πρέπει να τρέξουμε γιατί ο κόσμος κινείται όλο και περισσότερο προς τις ψηφιακέ τεχνολογίες. Κυρία Ρέντινγκ, θα ήθελα να αφιστεί στην προσοχή τη συζητήτριας και τη επιτροπή μα στα εξή. Έχουμε υποβάλει τροπολογίες για ζητήματα προτεραιότητε για το ΕΛΚ. Πρώτον, η προστασία των δικαιωμάτων του καταναλωτή. Θα πρέπει να γίνει πιο ξεκάθαρη, σαφής στο, ε, στις περιπτώσεις του, του μπλοκαρίσματος λόγω γεωγραφικής προέλευσης, geoblocking, το roaming και ε, δεύτερον θα πρέπει να αξιοποιήσουμε τις δονομικά εργαλεία του, του ΠΟΕ και ε, τη, τη ΣΥΤΑ και τη, τη, τη ε, TPP δεν θα πρέπει να καλύπτεται στις, στις εμπορικές συμφωνίες στην έκθεση αυτή το ζήτημα των πλατφορμών ε, που απλώς μοιράζουν δεδομένα, passive platforms, ε, γιατί δεν αμπίπτει στις αλπικές μας αμμοδιότητες. Και τέλο, όλε οι εμπορικέ συμφωνίε θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν κανόνε για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και θα έπρεπε να φτάσουμε μέχρι το σημείο να απορρίπτουμε τέτοιε συμφωνίε, αν δεν το έχουν αυτό. Ε, η θέση μα του ΕΛΚ και την έχουν εκφράσει και άλλες πολιτικές ομάδες όπως οι σοσιαλιστές, όπως το ΣΥΑΡ, ότι θα πρέπει να έχουμε ξεκάθαρες διατάξεις για την προστασία των προσωπικών δεδομένων πέρα από αυτές που έχουμε στην ΚΑΤΣ. Συμφωνούμε πάντως ότι η ψηφιακή οικονομία και η παγκοσμιοποίηση είναι ταυτόχρονα μοχλή ανάπτυξης αλλά και πηγή ανησυχίας θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα εμπόδια αφενό που αντιμετωπίζουν ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, αλλά επίσης και τις εύλογε ανησυχίε που έχουν οι Ευρωπαίοι πολίτες. Σα ευχαριστούμε. Για τους σοσιαλιστές, Καρλίν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε για την συμβαστική που μας στείλατε. Νομίζω ότι πηγαίνει προς τη κατεύθυνση. Έχουμε κάποια ε, τροπολογία όμως την οποία ε, θα θέλαμε να περάσει. Λέμε ότι ε, πέρα από τις ευκαιρίες το ψηφιακό εμπόριο ενέχει και κινδύνους που θα μπορούσαν να, από τους οποίους, μόνο θα μπορούσαν να προκύψουν αρνητικές επιπτώσεις τις οποίες θα πρέπει να προλάβουμε. Επίσης υπάρχουν κάποια κενά όσον αφορά τον πάροχο που πρέπει να καλυφθούν. Όσον αφορά το digital divide. Νομίζω ότι, ε, ότι υπάρχει μια διάσταση ανάμεσα στις αναπτυγμένες και λιγότερο αναπτυγμένες ε, ε, χώρες αυτό το ψηφιακό χάσμα υπάρχει αλλά και εντός των χωρών. Το, θα πρέπει να συνεχίσουμε την εργασία πιστεύω, κατά την άποψή μου δηλαδή, πιστεύω ότι θα πρέπει να ε, ε, συμπεριλάβουμε και μικρό μικροεπιχειρήσεις και start-up ε, που ε, πρέπει να έχουν πρόσβαση προς την αγορά. Ε, και γι' αυτό ακριβώς ε, θα πρέπει να προκύψουν κανόνες οι οποίοι θα γίνουν σεβαστοί και θα γίνουν σεβαστές και οι δεσμεύσεις που έχουμε αναλάβει. Η κυρία Σάκε επίσης είπε κάτι σημαντικό και εμείς έχουμε ένα αίτημα. Θα πρέπει ο φόρος να παρακρατείται εκεί εκεί όπου ε, ε, προκύπτει το κέρδος. Ε, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και νομίζω ότι και λόγω των Paradise Papers είναι πιο σημαντικό να ασχοληθούμε με το θέμα αυτό με μεγαλύτερη ένταση και πιστεύουμε ότι το θέμα της φορολογίας δεν θα πρέπει να αναφέρεται μονάχα σε αιτιολογική σκέψη αλλά και στο ίδιο το σώμα του κειμένου. Ε, θα πρέπει ε, στην ε, φορολογική διάσταση να συμπεριλάβουμε και την ευθύνη των ενδιαμέσων χρειαζόμαστε ένα ισοδίκιο σύστημα και επομένως θα πρέπει να βρούμε ισορροσημείο ισορροπίας ανάμεσα στην κυκλοφορία των δεδομένων από τη μία και την προστασία των δεδομένων από την άλλη. Υπάρχουν όμως και άλλα ερωτήματα τα οποία προκύπτουν και τα οποία δυστυχώς ε, δεν περιλαμβάνονται στον ε, συμβιβασμό και που είναι σημαντικά. Θα πρέπει να ενδυναμώσουμε το ρόλο των γυναικών ε, στην ψηφιακή οικονομία. Διαβούλευση για τα θέματα αυτά μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών. Σήμερα έγινε λόγος και για την προστασία των καταναλωτών, θέμα που όμως δυστυχώς δεν αναφέρεται επαρκώς εις το κείμενο για το ψηφιακό εμπόριο. Και κάτι άλλο. Ε, ορισμένα στοιχεία όσον αφορά ε, την προστασία των δεδομένων ε, δεν αναφέρονται αρκετά εκτεταμένα εδώ. Ευελπιστούμε ότι θα μας υποστηρίξουν οι συνάδελφοι την επόμενη εβδομάδα έτσι ώστε να προκύψει μια ισορροπημένη έκθεση. Σας ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ λέει ο Πρόεδρος. Ο συνάδελφος Χέλμουντ Σόλτ δεν είναι εδώ. Έχουμε όμως λαμπρό συνάδελφο από το ECR. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχω και εγώ δύο λόγια να πω ε, εξ ονόματο Σέμα Μακλάρκιν της κιόδους από την ομάδα μας. Είναι ευτυχής ε, και συγχαίρει του συναδέλφους ε, για την εργασία η οποία κατεβλήθηκε και η οποία έχει σαν αποτέλεσμα μια ευρεία συνένεση δημιουργία θέσεων εργασία, δημιουργία ανάπτυξη, μελλοντική καινοτομία, όλα αυτά προκύπτουν από την ψηφιακή οικονομία. Εμεί έχουμε θετική, ομα, ε, θετική στάση όσον αφορά ε, την ε, αναλογική άρση των κανονιστικών και μη κανονιστικών εμποδίων στην ελεύθερη ροή σε αφορά την προστασία, πιστεύουμε ότι ναι, υπάρχει, χώρος ε, για εμπορική πολιτική, γιατί θα πρέπει να ενθαρρύνουμε ε, τους Ευρωπαίους ε, προθέσεις της καινοτομίας να ασχοληθούν και με την προστασία της πνευματικής διανοητικής ιδιοκτησίας Ξέρουμε επίση ότι το ζήτημα αυτό είναι πολύ σημαντικό για τι μικρομεσαίε επιχειρήσει και μπορούμε να συμφωνήσουμε με κάποιου συναδέλφου που υπέβαλαν τροπολογίε ε, μέσω των οποίων καλύπτουν ιδιαίτερε ανάγκε, εξειδικευμένε ανάγκε αυτών των ε, μορφών επιχείρηση. Θα πρέπει ε, όλα αυτά να γίνουν προ το συμφέρον και των επιχειρήσεων και των πολιτικών. Όσον αφορά διορθώνω και των εταιριών και των καταναλωτών. Όσον αφορά τους ενδιαμέσους, Ε, θα πρέπει να προληφθούν ε, κάποιες ε, διαφορές οι οποίες θα μπορούσαν να ανακόψουν την πορεία των πλατφορμών και θα πρέπει να ε, ε, ε, επιλέξουμε μια πιο παγκοσμιοποιημένη τοποθέτηση βάσει και των νομοθετικών κειμένων που έχουμε ήδη εγκρίνει σε σχέση με το ψηφιακό εμπόριο. Σε γενικέ γραμμέ πιστεύουμε ότι εδώ πρέπει να ληφθούν κάποιοι βασικοί και να αναφερθούν κάποιοι βασικοί κανόνε οι οποίοι θα αποτελέσουν θεμέλιο για να προχωρήσουμε για το μέλλον και ε, πάντως σε γενικές γραμμές πιστεύουμε ότι εδώ επιτεύχθη ε, κάτι πολύ θετικό και ε, η ισχυώδης μας ευχαριστεί την εισηγήτρια. Ευχαριστούμε πολύ. Η Χάιντι Χαουτάλα για τους πράσινους. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για, τους, για τις συμβαστικές της και θα ήθελα συντόμως να θίξω κάποια θέματα. Όσον αφορά την γενική συνένεση η οποία αναφέρθηκε όσον αφορά την προστασία των δεδομένων. Ε, θα ήθελα, παρακαλώ, να ξανασκεφτείτε το συμβιβασμό υπαριθμό 13 και να δείτε λίγο την διατύπωση η οποία υπάρχει στην κοινή τροπολογία της ε, κυρίας Ρέντινγκ, του κυρίου Λαν και, και άλλων για να αντικατασταθεί το τμήμα που λέει providing that this provision κλπ. Ε, δηλαδή να μην ε, υπάρξει ε, κρυμμένη διακριτική μεταχείριση κλπ. Γιατί αν δούμε την κοινή τροπολογία λέει η μόνη, ο μόνος όρος που θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί έτσι ώστε να περιοριστεί η ροή των δεδομένων εκτός της προστασίας προσωπικών δεδομένων και συνεχίζει. Αυτό το πνεύμα θέλω να κρατήσουμε εγώ και επίσης Υπάρχουν και κάποια άλλα ζητήματα τα οποία είναι πολύ σημαντικά και νομίζω ότι καλά αντιπροσωπεύονται εις ε, την, ε, το συμβιβασμό 11. Ίσως θα μπορούσαμε να διαγράψουμε το τελευταίο τμήμα του συμβιβασμού 10 που υπενθυμίζει ότι ε, οι αποφάσεις συμμόρφωσης δεν αποκλείουν τις, δεν, τον αποκλεισμό μεταφοράς προσωπικών δεδομένων. Um, that on data protection and then και επίσης θα ήθελα λίγο να χτενίσουμε το κείμενο για να δούμε να το ευθυγραμμίσουμε λίγο ε, με τις ε, διαπραγματεύσεις οι οποίες λαμβάνουν χώρα αυτή τη στιγμή, δηλαδή να μην προδικάσουμε τίποτα σε αυτήν την έκθεση, γιατί νομίζω ότι στην Οδηγία Προστασίας Δεδομένων ίσως βρεθούν λύσεις πιο καλές. Τέλος, συμφωνώ με την διατύπωση όσον αφορά το profit shifting, την μεταβίβαση, μετατόπιση μάλλον ε, του κέρδους και τη φορολόγηση στο, ε, εκεί που ε, γίνεται το κέρδος. Πιστεύω ότι αυτό θα πρέπει να αναφερθεί σε μια παράγραφο του κειμένου και όχι σε αιτιολογική σκέψη. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Από την Κομισιόν ο κύριος Κίνα. Πού είστε κύριε Κίνα κύριο Σκίνα από την Κομισιόν. Ευχαριστώ πολύ. Αν μου επιτρέπετε θα ήθελα να πω δύο λόγια όσον αφορά την έκθεση που συζητούμε και μετά θα επανέλθω σε κάποια θέματα τα οποία παρέμειναν από την προηγούμενη συζήτηση. First, the uh, Για την έκθεση της κυρίας Μπούρη. Η δέσμευση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά το ψηφιακό εμπόριο είναι πάρα πολύ σημαντικό, κυρίω δεν λαμβάνοντα υπόψη και την ε, ε, έκθεση για την, ε, με τίτλο Προ μια νέα ψηφιακή στρατηγική. Εμεί ήδη έχουμε συζητήσει δύο φορέ για το θέμα αυτό, δώσαμε τα κάποια πρώτα σχόλια και οπωσδήποτε επιζητούμε την συζήτηση της τελικής εκδοχής της έκθεσης ε, όταν θα έχουν εγκριθεί και οι τροπολογίες σε τις οποίες αναφέρει και η κυρία Χάκερ. Όσον αφορά την προηγούμενη συζήτηση, αν μου επιτρέπετε, πολύ σύντομα υπάρχουν κάποια θέματα τα οποία θα ήθελα να θίξω. Ε, ε, εξ αρχής να πω ότι ενδεχομένως θα πρέπει να πούμε το εξής. Οποτεδήποτε έχετε τέτοιες μελέτες, θα ήθελα να ζητήσω από τις αρχές του Κοινοβουλίου να λένε κάθε φορά στους ερευνητές, μελετητές ότι μπορούν να έρθουν σε επαφή με την Κομισιόν για να έρθουν οποιαδήποτε στοιχεία. Και βεβαίως ε, η πρόσκληση αυτή ισχύει και για την κυρία Βιωρή. Κάτι άλλο το οποίο θα ήθελα να πω ε, ε, είναι το εξής. Ε, δίνεται η εντύπωση ότι η TTIP και η προσέγγιση των ΗΠΑ αποτελεί benchmark, αποτελεί σημείο αναφοράς. Ε, αυτό αποτέλεσε απλώς ένα στοιχείο στο τραπέζι. Και αν δει κανείς ε, την συμφωνία των ΗΠΑ με την Ιαπωνία, και την πρόταση που έχουμε κάνει εμείς για ψηφιακό κεφάλαιο με την Ινδονησία ή το Μεξικό, εάν τα βλέπατε αυτά λοιπόν θα καταλάβαινατε ότι οι αποχρώσεις ε, είναι πολύ πιο έντονες όσον αφορά την περιγραφή της κατάστασης αυτής. Επίσης ε, για θέματα αποκάλυψης εμείς ε, ε και απορρίτου εμείς προχωράμε πολύ περισσότερο από ότι στην TTIP έχουμε, ε, έχουμε προστασία καταναλωτών, έχουμε ηλεκτρονική υπογραφή, έχουμε προστασία προστασία ηλεκτρονικών ε, εγγράφων και της εμπιστοσύνης ταυτοποίησης των ε, ιδίων. Όσον αφορά τώρα ε, και την, και την ροή των δεδομένων, ναι, η Κομισιόν το λαμβάνει υπόψη και το μελετά. Ο συγγραφέας της μελέτης ε, θεωρώ ότι έχει δίκιο όταν λέει ότι θα πρέπει να ε, ε, δούμε την διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στην προστασία των δεδομένων και τον προστατευτισμό όσον αφορά τα δεδομένα. Πολύ σωστά το θέτει η, η μελέτη Κάτι άλλο το οποίο ξεχάστηκε στην έκθεση ε, και το οποίο κατά την άποψή μας είναι πολύ σημαντικό είναι ε, κάτι το οποίο αναφέρθηκε στην ε, στρατηγική της Κομισιόν με τίτλο «Οι νέες προκλήσεις των ψηφιακών δεδομένων σε μια παγκοσμιοποιημένη κοινωνία». Ε, αυτό μπορεί να αντιμετωπιστεί με κατάλληλες αποφάσεις με τους κεντρικούς εταίρους και μάλιστα στην έκθεση αυτή αναφέρεται ότι μπορεί να ακολουθηθεί ένας διαφορετικός διάβλος ε, που θα μπορούσε να συμπληρώσει κατά κάποιο τρόπο ε, τον αντίκτυπο, τον θετικό αντίκτυπο που μπορεί να έχει ε, αυτή η πολυτομιακή προσέγγιση. Δηλαδή να μην πηγαίνουμε απαραίτητα και μόνο στον ΠΟΕ που είναι βεβαίως μια καλή λύση. Θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε και διμερείς ε, διάβλους, όχι κάτι ε, ε, κατά αποκλειστικό. Αλλά και παραπέρα για όλες τις αποφάσεις επάρκειας και συμμόρφωσης με την επάρκεια. Πολύ ωραία. Αναφερθήκατε στην ε, συμφωνία ε, το, με το Μεξικό και την ε, Ιαπωνία. Δεν θα μπορούσατε μήπως να μας δώσετε αυτές τις προτάσεις σας, ας πούμε, γραπτά, να ξέρουμε, γιατί διαφορετικά δεν ξέρουμε τι έχετε προτείνει. Κύριε Κίνα, παρακαλώ η ένδειξη της κυρίας Μάλστρομ και ε, βάσει και της στρατηγικής ε, της ε, Κομισιόν πάντα δημοσιεύουμε επιγραμμικά online τις αποφάσεις μας πρόεδρος. Άρα όλοι θα έχουν την ευτυχία και την ικανότητα να δουν όλα αυτά τα στοιχεία. Η Μαρίτη Σκάκ. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Οι παρεμβάσεις των σκιωδών μου έδειξαν ποιες είναι οι προτεραιότητές τους. Θα συνεχίσουμε τη συζήτηση αναλυτικά στην πρώτη ευκαιρία, έτσι ώστε να καταλήξουμε στις συμβαστικές τροπολογίες. Κάποια τελικά συμπεράσματα, για να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση, πρέπει να δούμε τελικά τι εμπίπτει και τι δεν εμπίπτει στο πλαίσιο ε, της έκθεσης αυτής. Γιατί υπάρχουν κάποιες τροπολογίες που έχουν προταθεί από σκιώδεις που δεν θα ενέπιπταν κανονικά στο πεδίο της. Βεβαίως ε, υπάρχει σχέση, έχουν σχέση όλα τα ζητήματα αυτά με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, για την ουδετερότητα του δικτύου ή την προστασία του καταναλωτή και θα θέλαμε αυτές τις αρχές να τις περάσουμε και στο εξωτερικό. Και εξ, ε, ε, ε, τις ε, εμπορικέ συμφωνίε. Όμω, πρέπει να είναι ξεκάθαρο ότι δεν είναι οι εμπορικέ συμφωνίε ένα εργαλείο για να αλλάξει η ευρωπαϊκή νομοθεσία. Αντιθέτω, πρέπει να είναι πολύ ξεκάθαρο ω προ του συνομιλητέ μα, προ του συνομιλητέ μα, ποια είναι τα πρότυπα που έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό να το εκφράζουμε σε οποιαδήποτε διαπραγμάτευση, πολυμερή, διμερή πλειονομερή. Ε, θα, θα, πρέπει να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση ως επίγουσα γιατί υπάρχουν εξελίξεις σε ολόκληρο τον κόσμο. Διάβαζα χτες ένα πολύ αναλυτικό άρθρο στους New York Times για τις φιλοδοξίες που έχει η Κίνα να παίξει το ρόλο του συγγέτιδας δύναμης στην ψηφιακή οικονομία. Ας μην είμαστε αφελείς λοιπόν. Αν ε, φτάσουμε στο σημείο να δεχόμαστε τους κανόνες των άλλων ε, αντί να επιβάλλουμε τους δικούς μας επειδή θεωρούμε ότι οι δικοί μας εσωτερικοί κανόνες είναι οι καλύτεροι, στην πραγματικότητα θα έχουμε αυτό... Ε, αυτοκροτηριαστεί. Ε, είναι απαραίτητο λοιπόν να βρούμε μια ισορροπία. Ιδίω βλέποντα προ τα που πηγαίνουν οι ανταγωνιστές μας όσον αφορά το τρόπο διακυβέρνηση, λήψη αποφάσεων, θα ήθελα να προτείνω στους σκιώδες συζητητές να το δούμε και από, αυτό το, ε, από αυτή τη σκοπιά το θέμα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Η ψηφοφορία στην Επιτροπή θα γίνει στις 23 Νοεμβρίου. Και μπορούμε να ολοκληρώσουμε το συζήτηση του σημείου 12 και να πάμε στο 13. Η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων προετοιμάζει δύο εκθέσεις για τις σχέσεις μας με δύο σημαντικούς οικονομικούς εταίρους, με την Κίνα και με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Συμφωνήθηκε με την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου να συνεισφέρει στα θέματα που άπτονται του Διεθνούς Εμπορίου με βάση το άρθρο 54 του κανονισμού. Με βάση αυτό το άρθρο, η συνεισφορά της ε, ΙΝΤΑ στην έκθεση αυτή δεν θα μπορεί να τροποποιηθεί από την ΑΦΕΤ. Η πρώτη από τις δύο έκθεσεις, λοιπόν, εξετάζει τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης Κίνας και πιο συγκεκριμένα για εμάς α συζητήσουμε το ζήτημα των εμπορικών σχέσεων με την Κίνα και δίνω το λόγο στον κύριο Βίκλερ. Σας ευχαριστώ Προέδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, έχει τεράστια σημασία η Κίνα για τις εμπορικές συναλλαγές ε, με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ο δεύτερος εμπορικός μας εταίρος μετά τις Ηνωμένε Πολιτείε και είμαστε, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο σημαντικότερος εταίρος της Κίνας. Είναι η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία προς την οποία εξάγουμε. Έχουμε δισεκατομμύρια ε, που είναι αντικείμενο των οικονομικών συναλλαγών με, αυτές, με αυτή τη χώρα. Κάτι που συνεισφέρει στην ευημερία της Υπήρου μας και της Κίνας. Έχουμε εκτιμήσει ότι δημιουργούνται ε, εκατομμύρια θέσεις, εξαρτώνται μάλλον εκατομμύρια θέσεις εργασίας ε, από το εμπόριο με την Κίνα. Δεν αρκεί όμως να βλέπει κανείς το εμπορικό ισοζύγιο για να εξετάσει τη σχέση μας με την Κίνα. Συνεχίζουμε να έχουμε ένα σημαντικό έλλειμμα εμπορικών συναλλαγών με τη χώρα αυτήν, γιατί οι εξαγωγές μας, ιδιαίτερα αγαθών, δεν έχουν αυξηθεί, έχουν μάλλον υποχωρήσει τα τελευταία χρόνια, ενώ οι εισαγωγές από την Κίνα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν αυξηθεί ραγδαία. Ίσως και λύζεται το έλλειμμα στα αγαθά από τις εξαγωγές υπηρεσιών που κάνουμε προς τη χώρα αυτή. Αυτές οι συναλλαγές συνεισφέρουν στην ευημερία των πολιτών και στην Ευρώπη και στην Κίνα, όμως υπάρχουν και κάποια ανησυχητικά σημάδια. Πολλές από τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη χώρα αυτή μας έχουν κρούσει τον κόδωνα του κινδύνου για θέματα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Για παράδειγμα, δεν επιτρέπεται ε, να έχουν ισότιμη μεταχείριση. Το 55% των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων θεωρούν ότι υφίστανται διακρίσεις σε σχέση με τις αντίστοιχες κινέζικες εταιρείες το, οι άμεσες διεθνείς επενδύσεις ευρωπαϊκές στην Κίνα έχουν μειωθεί, ενώ οι άμεσες ε, επενδύσεις κινέζικων επιχειρήσεων στην Ευρώπη έχουν αυξηθεί ραγδαία. Ε, έχουν ξεκινήσει οι διαπραγματεύσεις IT από το 2013 και δεν είχαμε επαρκή πρόοδο το ζήτημα της πρόσβασης στην αγορά αυτή πρέπει να παραμείνει στη, στην ημερήσια διάταξη. Γιατί αν κάνουμε τη σύγκριση, είναι δύσκολο για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να ε, επενδύουν ή να επιχειρούν στην Κίνα, ενώ από την άλλη πλευρά οι κινέζικες επιχειρήσεις που αξιοποιούν το γεγονό ότι στην Ευρώπη έχουμε μια ελεύθερη αγορά. Βεβαίως, η επενδύσεις εάν βασίζονται σε ένα ισότιμο πλαίσιο ανταγωνισμού μπορεί να έχουν πλέον εκτίματα για όλους όμως σε πολλούς τομεί, η κινέζικη οικονομία έχει υπερβολικά μεγάλες δυνατότητες. Έχουν επίσης την πρωτοβουλία Made in China 2025 η οποία δημιουργεί κάποιες ανησυχίες. Αυτά τα στοιχεία λοιπόν ε, δημιουργούν ανησυχία και στις επιχειρήσεις μας που δραστηριοποιούνται στην χώρα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να εξετάσει την πιθανότητα να υιοθετήσει κάποια μέτρα για την προστασία ευαίσθητων τομείς, ε, τομέων για να προστατεύσει την βιομηχανία της που είναι πολύ σημαντική για την καταπολέμηση της αναργίας και για την κοινωνία στην Ευρώπη. πρωτοβουλία Balkan Law, αν ακούσαμε σωστά τον ομιλητή, είναι επίση ε, κάτι που δεν είναι ξεκάθαρο ε, το πώ θα λειτουργήσει και δεν έχουμε επίσης σαφήνεια, δεν είναι επίση σαφέ το πώ λαμβάνονται οι αποφάσεις. Ένα άλλο σημείο ανησυχία είναι οι κανόνες για τις διεθνείς ε, προμήθειες και η προστασία των περιβαλλοντικών προτύπων. Η προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων θα έπρεπε να πηγαίνει χέρι-χέρι με την πρόσβαση στην αγορά. Τα εμπορικά μας επιμελητήρια έχουν επισημάνει ποια είναι τα μέτρα που θα έπρεπε να λάβουν οι κινέζικες αρχές έτσι ώστε να σέβονται τα πνευματικά δικαιώματα το ρυθμιστικό πλαίσιο της Κίνας δεν έχει βελτιωθεί σε αυτόν τον τομέα αυτόν. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Και τις αποτρέπει από το να συνεισφέρουν στην ανάπτυξη της κινέζικης οικονομίας. Οι κινέζικες αρχές έχουν αναλάβει σημαντικές πρωτοβουλίες που θα έχουν ε, ε, επιπτώσεις στον πώς ε, λειτουργεί η βιομηχανία τους, όπως για παράδειγμα την αξιοποίηση μεγάλων όγκων δεδομένων για να δουν πώς λειτουργούν οι βιομηχανίες τους. Ε, όμως αυτές οι πρωτοβουλίες δημιουργούν και ανησυχίες όσον αφορά την προστασία των προσωπικών ε, δικαιωμάτων, των προσωπικών δεδομένων και των πολιτών μας και των επιχειρήσεών μας. Ε, η υποχώρηση των περιβαλλοντικών προτύπων επίση δημιουργεί προβλήματα και στις ε, κινέζικες και στις ξένες επιχειρήσεις. Χρειάζεται ε, συνεργασία τη χώρα αυτή για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής για να προσπίσουμε το, το ελεύθερο διεθνές εμπόριο όταν άλλοι διεθνοί παίχτες φαίνεται να πηγαίνουν προς περισσότερο προστατευτισμό Πρέπει να δούμε πώς η Κίνα θα εμπλακεί καλύτερα στη διεθνή λήψη αποφάσεων, στη λήψη αποφάσεων σε διεθνές επίπεδο, γιατί αναγνωρίζουμε τη σημαντική θέση που έχει αυτή η χώρα ε, στην παγκόσμια οικονομία, όμως πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι θα σέβεται και τις αρχές μας. Είναι μια εποχή λοιπόν προκλήσεων στο διεθνέ επίπεδο, γι' αυτό πιστεύω ότι πρέπει να ε, μιλήσει πιο ξεκάθαρα η Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά τις θέσεις της. Θεωρούμε ότι η Κίνα είναι ένας σημαντικός εταίρος στη διεθνή οικονομία και έτσι πρέπει να τον αντιμετωπίσουμε. Έτσι πρέπει να αντιμετωπίσουμε τη συνεργασία μαζί τους έτσι ώστε να οδηγηθούμε σε μια κατάσταση ε, προστασίας του ισότιμου ανταγωνισμού και του δικαίου. Αν συμβεί αυτό, θα είναι θετικό και για την Κίνα και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα δημιουργήσει ευκαιρίες. δεν θα πρέπει να επαναχωρήσουμε σε ζητήματα αρχών και σε σεβασμού των κανόνων, αλλά ταυτόχρονα να προσπαθήσουμε να έχουμε μια θετική προσέγγιση στους Κινέζους. Σας ευχαριστώ. Δεν βλέπω κάποιον άλλο σκιώδηση γιατί εδώ. Άρα θα ακούσουμε άλλα μέλη της... Ε, α, συγγνώμη, συγγνώμη, ξέχασα. Ζάντι από το νομάδα ECR. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. κάποιες παρατηρήσεις. Σήμερα άκουσα ότι ο κύριος Τραμπ και ο Κινέζος Πρόεδρος έχουν υπογράψει συμβάσεις αξίας 250 δις αμερικανικών δολαρίων. Και νομίζω ότι και αυτό είναι ακόμα ένα δείγμα της ε, κινέζικης ε, προσέγγισης ε, στην παγκόσμια οικονομία και αγορά. Το Μάιο η Κίνα είχε και φιλοξενήσει ένα φόρουμ ε, με πάνω από 130 χώρους, πέντε πρωθυπουργοί και ένας πρόεδρος από ευρωπαϊκή χώρα ήταν παρόντες. Σίγουρα αυξάνεται η παγκόσμια σημασία της Κίνας. Νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κάθε λόγο να θέλει να διαδραματίσει ένα σημαντικό ρόλο. Πρέπει να υπάρξει λοιπόν μια ισχυρή και προβλέψη μετερική σχέση μεταξύ Κίνας και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εξακολουθούμε να ζούμε σε μια κατάσταση που ε, ε, χαρακτηρίζεται από απουσία κάποια σημαντική εμπορική συμφωνία με την Κίνα. Ωστόσο, οι ροέ υπηρεσιών, αγαθών και οι επενδύσει ε, είναι υψηλότατε. Επομένω, αυτό το οποίο χρειάζεται είναι να ορίσουμε ξεκάθαρα το πεδίο των διαπραγματεύσεων στην επενδυτική συμφωνία με την Κίνα. Όπως είπε και ο κ. Βίνκλερ, Οι Ευρωπαίοι επενδυτέ έχουν να αντιμετωπίσουν ήδη πολλά, ακόμη μάλλον πολλά εμπόδια στην προσπάθειά του να έχουν πρόσβαση στι κινέζικε αγορέ. Και με τι άμεσε ξένε επενδύσει να ε, ε, επιβραδύνονται στην Κίνα και οι Κινέζοι επενδυτέ να έχουν εύκολη πρόσβαση στην αγορά, όλα αυτά στην Ευρωπαϊκή Ένωση σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε ένα πιο σωροπημένο επενδυτικό περιβάλλον. Το ίδιο ισχύει για τις επιχειρήσεις μας που προσπαθούν να δραστηριοποιηθούν στην κινέζικη αγορά. ενώ υπάρχουν κρατικές επιχειρήσεις ε, και κρατικές ενισχύσεις. Είναι ένα θέμα που πρέπει να μας απασχολήσει. Πανέρχομαι στη δυνητική αυτή συμφωνία. Θα χρειαστεί να εστιάσουμε σε τρία πράγματα. Πρώτον, βελτιωμένες συνθήκες πρόσβασης στις κινέζικες αγορές από τους, ε, για τους επενδυτές από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγγυήσεις για την αντιμετώπιση των επενδυτών από την Ένωση, προστασία τους από αθέμητη ο ανταγωνισμό διακρίσης και μεταφορά κεφαλαίων πληρωμών που σχετίζονται με επενδύσεις. Δεύτερον, ισότιμο πεδίο ανταγωνισμού. Με βάση την αρχή τη μη διακριτική μεταχείρισης. Τρίτον, αντιμετώπιση βασικών προκλήσεων. Για τη δημιουργία κοινού ρυθμιστικού πλαισίου. Για να υπάρχει συμβατότητα των δύο μερών. Και συμβατότητα και με τους διεθνεί κανόνες. Πολύ πρόσφατα βρεθήκαμε σε μια σχιζοφρενική κατάσταση. Καταμένη. Γιατί από τη μία θέλουμε να προωθήσουμε τις εμπορικές και επενδυτικές σχέσεις με την Κίνα και από την άλλη θεσπίζουμε νέους κανόνες για την προστασία ορισμένων κλάδων της ευρωπαϊκής οικονομίας από αδικαιολόγητο θέμη το dumping θα ψηφίσουμε δε την επόμενη εβδομάδα στην Ολομέλεια το σχετικό νομοθέτημα. Υπάρχει μία ερώτηση προς την Κομισιόν και θέλω μια σαφή απάντηση. Σε ό,τι αφορά το πάνελ του ΠΟΕ, πού βρισκόμαστε ακριβώς. Μπορούμε να περιμένουμε άμεσα μια ετοιμιγορία και αν η ετοιμιγορία δεν είναι θετική για την Ευρωπαϊκή Ένωση, είμαστε προετοιμασμένοι για ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Η Κίνα ξέρουμε ότι επιτίθεται και έχει και κάθε δικαίωμα να το κάνει. Το παλιό σύστημα ε, θέλει ε, να το Ε, καταργήσει και το γιος δεν συμφωνήσαμε το Δεκέμβριο να τις χορηγηθεί καθεστώς ε, χώρες οικονομίας της αγοράς ε, είναι κάτι που θα κάνει την Κίνα να θελήσει να επιτεθεί κατά του συστήματος. Άρα ποιες είναι οι δυνατότητες, οι πιθανότητες, οι προβλέψεις και τέλος έγινε μια πολύ προκαταρκτική συζήτηση για ένα λεγόμενο investment screening scheme και επίκειται, το ανακοίνωσε ο πρόεδρος Γιουκέρ. Και νομίζω ότι θα πρέπει και εδώ να έχουμε κάποιες εγγυήσεις. Ελπίζω να μην επηρεάσει αυτό τις εθνικές δικαιοδοσίες και να μην είναι πολύ επεμβατικό ως προσέγγιση. Ο κύριος ε, Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Αλέσια Μόσκα παρακολουθεί το θέμα. Μου ζήτησε να διαβάσω την παρέμβασή τη και θα το κάνω με μεγάλη χαρά. Παρά τα θετικά τη στοιχεία, η έκθεση για τον τελευταίο γύρο των διαπραγματεύσεων για μια επενδυτική συμφωνία με την Κίνα δεν θα πρέπει να μας δημιουργεί αυταπάτες. Καμία πρόοδος δεν, έχουμε, ε, δεν έχει σημειωθεί σε, θέματα που έχουν να κάνουν με παλαιοτεώσεις. Ε, η προστασία των επενδυτών. Οι Κινέζοι επενδυτές υποφελούνται από το άνοιγμα της ε, ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς. Έχουν ισότιμη μεταχείριση, ενώ αντιθέτως το Ευρωπαϊκό Εμπορικό Επιμελητήριο στην Κίνα μας περιγράφει όλο και χειρότερες συνθήκες χρόνο με το χρόνο για τους Ευρωπαίους επενδυτές. Γιατί λοιπόν ενδιαφέρεται η Κίνα να συνάδει άψε μια συμφωνία που θα βάλει Κινέζους και Ευρωπαίους ε, σε, ε, στο ίδιο επίπεδο. Επίσης, η πολιτική της Ένωσης με βάση τα θετικά κίνητρα δεν έχει λειτουργήσει με τους Κινέζους εταίρους, γιατί αυτοί στηρίζονται πιο πολύ σε ε, μια συναλλακτική προσέγγιση. Για να υπάρχει αμοιβαιότητα θα πρέπει να διδαχθούμε τα δάγματα του διεξόδου αυτού και να αξιοποιήσουμε ως μοχλούς τα εργαλεία που έχουμε στη δεσή μας. Η κυρία Μόσκα λοιπόν λέει για μια φορά πλέον ας χρησιμοποιήσουμε το ε, μαστίγιο αντί του καρότου για τρία σημεία. Πρώτον, ε, για το φυτάρισμα των επενδύσεων. Χρειάζεται επενδύσεις ε, στην ευρωπαϊκή οικονομία, όχι με κάθε τίμημα. Έχουμε εχθρικούς, εχθρικές ελέγχους, εχθρικούς ελέγχους από τις ξένες χώρες. Αυτό διασπά την ενότητα. Προσπαθεί να αλλοιώσει την εσωτερική ισορροπία στην Ένωση, η Κίνα και τη σχέση με τις τρεις. Δεύτερον, πάντα με την κυρία Μόσκα, σύστημα αμοιβαιότητας ε, για τις δημόσιες προμήθειες με βάση τη δυναμική που υπάρχει. Έχουμε τις νέες ε, τροπολογίες ε, για τον και το φιλτράρισμα κτλ. Το θέμα είναι να βρούμε ένα συμβιβασμό για την αμοιβαιότητα στι δημόσιε προμήθειε. Αυτό που ζητούμε και εδώ είναι να γίνει σεβαστή αρχή τη αμοιβαιότητα. Εργαζόμενοι και βιομηχανίε δεν θα μπορούν πλέον να υφίστανται αυτό τον ε, ολοκληρωτικό ανταγωνισμό χωρί να μπορούν να ε, δραστηριοποιηθούν σε τρίτε αγορέ. Τρίτο θέμα. Μέτρα εμπορική άμυνα. Πολύ καλή συμφωνία για τη νέα μεθοδολογία κατά του ντάμπινγκ. Αυτό που πρέπει να κάνουμε τώρα είναι να χρησιμοποιήσουμε τις προσπάθειες, ε, τα λέω καλά κύριε Μάρτιν, να έχουμε ένα, ένα ενισχυμένο σύστημα και να μην έχουμε μόνο τη μεθοδολογία αλλά και τα απαραίτητα εργαλεία για να είμαστε αποτελεσματικοί. Το τελευταίο που θέλει να πει η κυρία Μόσκα και δεν έχει συζητηθεί μέχρι στιγμή στη ε, συζήτηση και επαφή με στη δική σας σοφία. Ιβάν. Θέλω να την αναφέρω. Με την ε, πολιτική της ενία Κίνας πρέπει να μπορούμε να έχουμε συζητήσει και με την Ταϊβάν. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με διάφορα ψηφίσματα πάντοτε έδειξε ότι είναι υπέρ τη έναρξη άμεσων διαπραγματεύσεων με την Ταϊβάν. Στην ανακοίνωση του εμπόρου για όλου η Κομισιόν καταλήγει στο ίδιο συμπέρασμα, ωστόσο οι πόρου, Δηλαδή τη σύναψη παρόμοια συμφωνία με την πρωτική ε, Κίνα. Επειδή λοιπόν το Πεκίνο δεν δείχνει επαρκέ επίπεδο φιλοδοξία, θα έπρεπε ίσω να ζητήσουμε την Κομισιόν να ξεκινήσει από τώρα διαπραγματεύσει με την Ταϊβάν. Εγώ δεν είμαι ειδικό για την Ταϊβάν, τα λέει η κυρία Μόσκα. Για τα υπόλοιπα όμω συμφωνώ απόλυτα με τι απόψει και τα συμπεράσματά τη. Δηλαδή, ναι, ότι ε, υπάρχουν ακόμη στρεβλώσει στην Κίνα και ναι, δεύτερον, το είπαν και οι συνάδελφοι, η Κίνα εξακολουθεί να ασκεί επιθετική εμπορική πολιτική με βάση τη στρατηγική του διέρη και βασίλευε, δηλαδή διέρη την Ευρώπη για να βασιλεύει. Και κλείνει τις δικές της αγορές ενώ ε, έχει πρόσβαση στις άλλες αγορές. Και τέλος, κάτι που μας βρίσκει όλους σύμφωνοι στην ομάδα, Περισσότερο από ποτέ χρειάζονται αυτά τα μέτρα αμοιβαιότητα για την καταπολέμηση του ντάμπινγκ, για την πράσπισή μας από τις εχθρικές επενδύσεις και για να υπάρχει και ευνοϊκή πρόσβαση των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στις ξένες ε, αγορές, στους ξένους διαγωνισμούς. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστούμε πολύ και εσά και την κυρία Μόσκα που τα έγραψε τόσο ωραία. Θα δώσω τώρα το λόγο στην Κομισιόνα. σε μια κυρία από την Κομισιόν, της οποίας το όνομα δεν μπορώ να πω, λέει ο Πρόεδρος. Σας ευχαριστώ πολύ. Δεν έχω και πολλά να πω και να προσθέσω, γιατί νομίζω ότι οι εισηγητέ και οι σκιώδες εισηγητές έκαναν εξαιρετική προσπάθεια σύνοψη όλων, όλων των στοιχείων που χαρακτηρίζουν τη σχέση μας με την Κίνα. Κατανοώ ε, τα μελήματα, τους προβληματισμούς της κυρίας Μόσκα στη στρατηγική μας ε, για την ε, Κίνα βάσει του κοινού ανακοινωθέντος ε, είναι σαφής, δηλαδή έχουμε υψώσει πολύ τον τόνο και παραμένει χώρος βέβαια για διαδικασίες όσον αφορά τις εμπορικές ε, συναλλαγές. Ε, δεν φαίνεται να είναι τόσο εύκολη η αλλαγή όπως όλοι ελπίζαμε. Ε, δεν μας εκπλήσει όμως αυτό γιατί ζητούσαμε και πολλά πράγματα. Ε, σχετικά με, τις, ε, με τους ε, μικροφόρους, σχετικά με το ρυθμιστικό πλαίσιο, σχετικά με την αμοιβαιότητα και την ίδια πρόσβαση. Κοιτάξτε, δεν προχωρούν τα πράγματα όσο γρήγορα θα επιθυμούσαμε, αλλά πάντως έχουμε κάποια ενθαρρυντικά μηνύματα, σημάδια δέσμευσης από την άλλη πλευρά. Και εμείς βέβαια προσπαθούμε τα μάλλα έτσι ώστε να προοδεύσουμε όσον αφορά τις διαδικασίες αυτές. Υπάρχουν πολλά στις διμερείς μας σχέσεις ε, που δεν είναι εύκολο ή ε, η υπερβολική παραγωγή είναι ε, ένα από αυτά τα προβλήματα. Δουλεύουμε σε πολλά επίπεδα έτσι ώστε να προσπαθήσουμε να αντιμετωπίσουμε όλα τα προβλήματα. Συλλέγουμε πληροφορίες, προσπαθούμε και σε πολιτικό επίπεδο να δεσμεύσουμε την Κίνα να δούμε μέχρι πού μπορούν ε, να μας δώσουν οι υφιστάμενοι κανόνες ε, την δυνατότητα να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα. Ένα μήνυμα από τη δική μας πλευρά. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο να ε, βρούμε το σωστό βαθμό και σημείο πίεσης με την Κίνα παραδοσιακά, αλλά είναι σημαντικό να διατηρήσουμε τους μοχλούς πίεσης που έχουμε και ο κυριότερος μοχλός είναι να παραμείνουμε ενωμένοι οι εσωτερικοί διαχωρισμοί είναι αυτοί που μας κάνουν πιο ευάλωτους. Γι' αυτό λοιπόν ζητώ από το Κοινοβούλιο να παραμείνει στο ενωτικό μέτωπο απέναντι στην Κίνα. Ευχαριστώ. Εν τη ενώση ισχύς, λέει και ο Πρόεδρος. Έχετε δίκιο, κύριε Βίνκλαρ. Πρώτα απ' όλα, κύριε Πρόεδρε, δεν άκουσα καμία απάντηση σχετικά ε, με την επίλυση διαφορών Καταλαβαίνω ότι δεν υπάρχουν πληροφορίες για το θέμα. Απάντηση. Ε, οι διαδικασίες δεν έχουν ολοκληρωθεί. Βρίσκονται ακόμα ε, σε διαπραγμάτευση. Δεν έχουμε κάτι προς ώρας. Είμαστε πάντως απολύτως πεπισμένοι ότι η πρότασή μας και η υφιστάμενη νομοθεσία πλήρως συμμορφούνται με τους ε, κανόνες ε, του ΠΟΕ και θεωρούμε ότι είναι ικανό νομικό, ικανή νομική βάση, αλλά ακόμα δεν έχουμε ε, τελική απάντηση. Σας ευχαριστώ πολύ, λέει ο κύριος Βίγκλερ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ συνάδελφοι. Πολλά σωστά υπόθηκαν, τρία συμπεράσματα από τη δική μου πλευρά. Βεβαίως, θα συνεχίσουμε την εργασία επί του θέματος και βεβαίως είμαι διατεθειμένος να βρω κάποιες ε, κοινέ ε, ε, θέσεις και οι παρατηρήσεις μου τώρα σχετικά με τον κανονισμό anti-dumping και τη μεθοδολογία anti-dumping είμαι απολύτως πεπισμένος ότι η υποστήριξη της ευρωπαϊκής βιομηχανίας δεν σημαίνει ταυτόχρονα και προστατευτισμό. Έχουμε εργαλεία για να προστατέψουμε, για να προωθήσουμε την, τα συμφέροντα τη βιομηχανία. Δεύτερον, ε, ναι βεβαίω το διέρη και βασίλευε ε, δεν είναι κάτι καινούριο, το γνωρίζουμε, ίσχυε στο παρελθόν, ισχύει τώρα, θα ισχύσει και στο μέλλον. Μα είπε και η Κομισιόν ότι πρέπει να παραμείνουμε ενωμένοι. Ναι, αλλά επί, σε ποιο μέτωπο θα πρέπει να παραμείνουμε ενωμένοι, ειδού το ερώτημα. Ε, πρέπει να βρούμε ένα ε, σταθερό ε, υπέδαφος, ε, υπόβαθρο για, την, ε, για, τη, για το κοινό μέτωπο και εκεί θα πρέπει οπωσδήποτε να περιλαμβάνεται και η προστασία των, της ευρωπαϊκής βιομηχανίας. Χαιρόμαστε που το ΕΛΚ και άλλες ομάδες υποστηρίζουν το άνοιγμα των διαπραγματεύσεων με την Ταϊβάν. Θα πρέπει να δούμε από κοινού τι θα πρέπει ακριβώς για το θέμα αυτό να περιληφθεί στη νέα γνωμοδότηση. Αυτά ήθελα να πω, Πρόεδρε, και σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, κύριε Βίγκλερ. Προς όλες δεν έχουμε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Όταν η και η Άφετ θα, θα έχουν συμφωνήσει επί του χρονοδιαγράμματος, θα σας το κοινοποιήσω. Ωραία λοιπόν, ολοκληρώθηκε και το σημείο 13 και πάμε κατευθείαν στο 14. Είναι παρόμοια διαδικασία. Θέλουμε να προσπαθήσουμε να ε, θέλουμε να προσπαθούμε πάντα να έχουμε καλές συμφωνίες με τους κύριους εμπορικούς εταίρους, εν προκειμένου με τις ΗΠΑ. Και τώρα θα αλλάξω το καπέλο μου γιατί, και θα φορέσω το καπέλο του εισηγητή, γιατί είμαι εγώ εισηγητής. Και θα αλλάξω και γλώσσα. Θα σας κάνω μια εισαγωγή. Η σχέση με την Στι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ε, κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Έχουμε πολύ καλές εμπορικέ σχέσεις με τις ΗΠΑ. Αλλά δεν υπάρχει και μεγάλη ισορροπία. Έχουμε πλεόνασμα εμπορικού ισοζυγίου, το οποίο δεν αρέσει στη ΣΥΠΑ και ασκούν κριτική και θα πρέπει να δούμε εσωτερικά τι μπορούμε να κάνουμε εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αν δούμε τις ροές, διαπιστώνουμε ότι σε ό,τι αφορά τα κατεργασμένα προϊόντα, η προϊόντα αξίας, ε, τα εξάγουμε πιο πολύ στη ΣΥΠΑ, ενώ εισάγουμε πιο πολύ πρώτες ύλες για τον γεωργικό κυρίως τομέα. Και εκεί δηλαδή δεν υπάρχει εντελώς απόλυτη ισορροπία. Θεωρώ λοιπόν ότι πραγματικά έχει σημασία να βελτιώσουμε τις εμπορικές μας σχέσεις μέσω διαπραγματεύσεων. Με το TTIP τα ξέρουμε και τα θυμόμαστε πάρα πολύ καλά και είδαμε πόσο δύσκολο ήταν να έχουμε μια εύλογη σχέση, μια λογική σχέση, για να μπορέσουμε να αναπτύξουμε ακόμη περισσότερο τις σχέσεις μας. Ιδίως σε ό,τι αφορά τη βελτίωση των ε, όρων πρόσβασης στους διάφορους τομείς. Δασμοί, αλλά όχι μόνο. Θέσπιση κοινών κανόνων σε πολλούς τομείς. Ανταλλαγή, ε, πληροφοριών, διευκόλυνση στον τομέα αυτό επί Ομπάμα δεν μπορούσαμε να επιτύχουμε συμφωνία και επί Τραμπ είναι, θα έλεγα κάτι μπορούμε να το θεωρούσουμε απίθανο. Άρα αυτή τη στιγμή είμαστε στις εμπορικές μας σχέσεις σε ένα στάδιο που χαρακτηρίζεται από βεβαιότητα. Σε πολλούς τομείς δεν υπάρχουν σαφείς προοπτικές σε σχέση με το πώς βλέπουν οι, οι τις εμπορικές τους σχέσεις ε, με εμάς και προς εμάς. Πώς θέλουν να τις διαμορφώσουν στο μέλλον. Και μάλιστα ενίοτε ε, γίνονται και κάποια περίεργα, περίεργα γεγονότα. Το βλέπουμε ε, και μεταξύ του Οίκου και του Υπουργείου Εμπορίου και των ε, ειδικών για το εμπόριο να λέει άλλο ένας και άλλο άλλος. Άρα ξεκάθαρα δεν γνωρίζουμε ποια είναι η στρατηγική εμπορική της Αμερικής απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και υπήρξαν και κάποια στοιχεία τα οποία τα αντιμετωπίζουμε με επιφύλαξη και σκεπτικισμό στην Ευρώπη για την αύξηση παραδείγματο χάρη των δασμών ορισμών προϊόντων 22% συγκεκριμένα αύξηση θεωρώ ότι αυτό ε, δεν δικαιολογήθηκε επαρκώς και με ατράνταχτα επιχειρήματα χρησιμοποιήθηκε ένας ε, νόμος από το, την εποχή του για τη χαλιβουργία. Το άρθρο 232 για το κατά πόσον ο Χάλιβας εμπίπτει στα αστικά συμφέροντα ή όχι. Τίθεται λοιπόν ε, και το θέμα της εθνικής ε, δεν το έχουμε ακόμα ξεκαθαρίσει. Ίσως και τον Ιούλιο θα το συζητήσουμε και θα δούμε τις διάφορες επιλογές που έχουμε, αλλά προς το παρόν επικρατεί μεγάλη αβεβαιότητα. Είχαμε επίσης μια νέα συζήτηση για ε, κάποιο δυνητικό dumping για τις ελιές και την εισαγωγή ελιάσα στις ΙΠΑ. Και επίσης, σε ό,τι αφορά την απαγόρευση εισαγωγών, για κάποιες ε, κατηγορίες βοηού Έχουμε και αυτό το θέμα με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και υπάρχει μια τάση να το κυνηγήσουν το θέμα ενεργά. Αυτό το οποίο με ανησυχεί ιδιαίτερα είναι το γεγονός ότι δεν έχουμε από κοινού μία στρατηγική εμπορική σε παγκόσμιο επίπεδο. Στο Πανοσάρι, σε διάσκεψη, 24 Οκτωβρίου. Εκεί ακούσαμε από τον Αμερικανό μια θέση ριζοσπαστική σε ό,τι τα θέματα που έχουμε επιτάπητος. Ότι δεν θα πρέπει τα θέματα που άπτονται αυτή τη διάσκεψη και, αυτού, και του ΠΟΕ να τα συζητούμε πια γιατί είναι πάρα πολύ αμφιλεγόμενα και δεν μπορούν να ξεκαθαριστούν. Άρα δεν χρειάζεται να ασχοληθούμε πλέον και πρότεινε να διαπραγματευτούμε στο πλαίσιο της του ΠΟΕ μία μεταρρύθμιση. Μάλλον δεν το λέω ακριβώς έτσι. Είπε not a negotiation, just an exchange. Δηλαδή ανταλλαγή μόνο για μεταρρυθμίσεις ενδεχομένως. Τελείως διαφορετική προσέγγιση με αυτή που σήμερα εμείς αποφασίσαμε με το ψήφισμά μας για τον ΠΟΕ. Μεγάλη λοιπόν η διαφορά σε ό,τι αφορά την εμπορική στρατηγική των δύο πλευρών. Σε ό,τι αφορά τις εμπορικές σχέσεις, το μόνο που μου φαίνεται να έχουμε κοινό προσέγγιση είναι η σχέση σε, με άλλους μεγάλους εμπορικούς εταίρους. Μιλήσαμε για την Κίνα πριν από την Ασία και έχουμε το θέμα του dumping. Πράγματι την κερδοσκοπία, την νομισματική επίσης. Εδώ νομίζω ότι βλέπουμε τα πράγματα το ίδιο μήκος Το θέμα είναι βιώσιμα, αν θα προχωρήσει έτσι το πράγμα. Και κατά συνέπεια όλων αυτών, η δετικοποίηση και ενίσχυση των εμπορικών σχέσεων βασίζεται σε συγκεκριμένες συμφωνίες. Αυτό δεν το βλέπουμε προς το παρόν. Το μόνο που μπορούμε να δούμε είναι ότι χρειάζεται να συνεχιστεί ο διάλογος. Αυτά είχα να πω για ε, το θέμα αυτό είναι εισαγωγής και τώρα θα δώσω το λόγο στους σκιώδεις συγκητές. Ο Χέλμου του Σόλτς είναι ο πρώτος. Ε, ε, Ευχαριστώ πολύ, Μπέρντ περιέγραψες ε, πολύ καλά την κατάσταση για τις μελλοντικές, θα για τις παρούσες και μελλοντικές εμπορικές μας σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και συμφωνώ σε πολύ μεγάλο βαθμό με αυτά που είπες. Θα πρέπει ε, όμως να δούμε να ε, μην περιοριστούμε στις εμπορικές πτυχές αλλά γενικά πώς δρά στο πλαίσιο εξωτερικής πολιτικής ε, η Αμερική. Έχουμε ε, ένα χρόνο από την ανάληψη καθηκόντων του Τραμπ, το ταξίδι του στην Ασία, είδαμε τις, ε, το που έδωσε έμφαση, τα σημεία που τόνισε, America First. Και στο μέλλον πιστεύω και οι εμπορικές σχέσεις και οι εμπορικές συνομιλίες θα ε, έχουν ως γνώμονα αυτή την αρχή. Θα δούμε τι θα γίνει ε, με την, ε, στο πρώτο τρίμηνο της επόμενης χρονιάς και αν υπογραφεί η συμφωνία. Θα δούμε αν θα έχουμε πρόταση από τις Ηνωμένε Πολιτείες για να επαναληφθούν οι συνομιλίες και ε, αν συμφωνούμε, ελπίζω να δούμε ε, αν θα μπορούσαμε να κάνουμε ένα βήμα για το μέλλον των εμπορικών μας ε, σχέσεων με τη ΣΥΠΑ. Αλλά για να το κάνουμε αυτό πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι. Θα πρέπει να, να δούμε τι θα κάνουμε μετά το Δεκέμβριο του 2016 με βάση την πολιτική και οικονομική ε, εξέλιξη και κατάσταση που έχουμε και με βάση αυτά να δούμε πώς θα εξελιχθούν οι εμπορικές μας σχέσεις με τις ε, ΗΠΑ. Πολύ προσεκτικά τον κύριο Σαλαφράκα που είπε για το Μεξικό. Δεν θα πρέπει να ε, μας περιορίζουν οι εξελίξεις σε διαπρα... συμφωνίες που διαπραγματεύονται τρίτη εταίρη. Αντίστοιχα πιστεύω ότι έτσι θα πρέπει να σκεφτούμε και εδώ. σε σχέση με πολιτικές συμφωνίες και πιθανή συζητήσεις και πιθανή συμφωνία. Και στην ε, ε, δική μας γνωμοδότηση ε, στην έκθεση ΑΦΕΤ νομίζω ότι θα πρέπει να το πούμε ξεκάθαρα. θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας κυρίως ε, τα ευρωπαϊκά εμπορικά, βιομηχανικά και κοινωνικά συμφέροντα της Ένωσης. Ευχαριστώ. Κύριε Σαραντιο, εκ μέρους της κυρίας Έμα Σας ευχαριστώ. Θα είμαι σύντομος. Γνωρίζετε όλοι ότι η πολιτική μας ομάδα υποστηρίζει μια ισχυρή διατλαντική συνεργασία εμπορική, όχι μόνο για οικονομικούς λόγους, αλλά επίσης και για γεωστρατηγικούς. Πάντοτε θεωρούσαμε αυτή τη σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες κρίσιμες σημασίας και ζωτικής σημασίας. Ακόμη και χωρίς την TTIP. Είναι τεράστιες εμπορικές συναλλαγές και τεράστιες επενδύσεις κατέρωθεν. Άρα η TTIP μόνο το ερώτημα που τίθετο είναι αν θα πρόσθετε κάτι και πόσο. Όμως δεν είναι καταστροφή το δεν έχουμε ακόμα τη TTIP. Θα θέλαμε όμως να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις και να αξιοποιήσουμε οποιαδήποτε ευκαιρία θα μπορούσαμε να έχουμε για να τις αναζωογονήσουμε, για να ξαναξεκινήσουν με όποιον τρόπο. Και αν μπορούμε το Σεπτέμβριο η Έμα και εγώ επισκεφτήκαμε την Ουάσιγκτον, συζητήσαμε με προσώπους του Υπουργείου Εμπορίου. Η αίσθηση τους είναι ότι δεν έχει ακόμα πάψει η διαπραγμάτευση, δεν είναι, πια, δεν είναι ακόμα ε, νεκρή η TTIP και ότι θα μπορούσε να αναθερμανθούν οι διαπραγματεύσεις όπως σωστά επεσήμανε ο Πρόεδρος βέβαια υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στη λειτουργία του και την οτροπία του Υπουργείου Εμπορίου και του Λευκού Οίκου Πάντως, θα πρέπει από τη δικιά μας πλευρά να είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε σε, μια πρόσκληση για επανάληψη των διαπραγματεύσεων και να θωρακιστούμε έτσι ώστε αν ξαναξεκινήσουν τέτοιες διαπραγματεύσεις να μην επαναλάβουμε τα λάθη του παρελθόντος. Δηλαδή, χρειάζεται διαφάνεια στις διαπραγματεύσεις για εμπορικέ συμφωνίες στο μέλλον. Θα πρέπει επίσης να είναι απολύτως ξεκάθαρες οι επιδιώξεις μας και εξίσου ξεκάθαρα να παραδεχόμαστε και να αναδεικνύουμε τις διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των δύο πλευρών. Να έχουμε επίσης μια πολιτική, μια στρατηγική για τη δημοσιότητα, για την επικοινωνία, για να αποφύγουμε παρεξηγήσεις. Αυτή τη στιγμή η αύξηση του διεθνούς εμπορίου υπολείπεται της διεθνούς οικονομικής μεγέθυνσης για πρώτη φορά μετά τα μέσα του προηγούμενου αιώνα. Το οποίο σημαίνει ότι χρειάζεται ε, να ξαναξεκινήσουμε την προώθηση της, του ελεύθερου εμπορίου διεθνώς και το πιο λογικό και εύλογο να κάνει κανείς είναι να το επιδιώξει αυτό με τη μεγαλύτερη ε, οικονομία παγκοσμίω. Ευχαριστώ, Πρόεδρε το κίνημα των πέντε αστέρων ήταν πάντα κατά του TTIP. Όχι γιατί δεν αγαπάμε το εμπόριο, τις ελεύθερες συνταλλαγές ή μια μεγαλύτερη επαφή με τις ε, Ηνωμένες Πολιτείες. Ε, είμαστε κατά ε, του περιεχομένου της συμφωνίας TTIP λόγω της έλλειψης των εγγύησεων όσον αφορά τις ενδείξεις γεωγραφικής προέλευσης, όσον αφορά τον μη σεβασμό και τη μη τήρηση των υγειονομικών κανόνων, την προστασία των ε, μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να σταματήσουμε τη σχέση με τις Ηνωμένε Πολιτείε, ε, αλλά ε, σίγουρα θεωρούμε ότι ό,τι έχει βγει από την πόρτα δεν μπορεί να ξαναμπεί κρυφά από το παράθυρο η Κομισιόν τώρα θέλει ε, να συνάψει συγκεκριμένες και για συγκεκριμένους τομείς ε, συμφωνίες ας πούμε στον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας ή στον κλάδο της φαρμακοβιομηχανίας. Πρόκειται οπωσδήποτε για ε, τομείς στους οποίους πραγματικά είναι ευκταίο να μπορέσουμε να βρούμε κοινέ αρχές ας πούμε για την αυτοκινητοβιομηχανία. Είναι καλό λοιπόν να βρεθούν κάποιες κοινέ λύσει ε, για προβλήματα τα οποία είναι στην ουσία τα προβλήματα και τα προσκόμματα μονάχα τεχνικά και ενδεχομένως πιο ε, εύκολα να λυθούν. Εκεί όμως που ε, πραγματικά θα είμαστε ακαπτοί είναι οπουδήποτε πρέπει και να εφαρμοστεί η ρήτρα πρόληψης. Δηλαδή οτιδήποτε σχετίζεται με την προστασία των καταναλωτών, προστασία της υγείας των πολιτών κτλ. Ε, οποιασδήποτε αρχές ε, ε, αμβλύνουν τα όρια προστασίας μας δεν μπορούν να μας βρουν σύμφωνος. Επομένως εμείς μπορούμε να συμφωνήσουμε με τεχνική συνεργασία η οποία θα πρέπει αναπερίπτωση να ελέγχεται αλλά δεν είμαστε σύμφωνοι με οποιαδήποτε στοιχεία της συμφωνίας TTIP με τις Ηνωμένες που απειλούσαν την υγεία των πολιτών. Ευχαριστώ πολύ ο David Μάρτιν. Um, σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Βεβαίω χρειάζεται μια συζήτηση του πώ θα βελτιώσουμε τι εμπορικέ μα σχέσει με τι Ηνωμένε Πολιτείε και με την παρουσία σα φτάσατε να φτάνω να διαπιστώνω ότι συμφωνούμε ότι αυτή τη στιγμή είναι πολύ καλές οι εμπορικές μας σχέσεις με τις Ηνωμένε Πολιτείες και αυτό που θα έπρεπε να φροντίσουμε είναι να αποφύγουμε τη ζημία σε βραχυπρόθεσμο επίπεδο και να δούμε πώς πιο μακροπρόθεσμα θα μπορούσαμε να φροντίσουμε να επανέλθουν γνώμη για την έκφραση, να επανέλθουν στο διεθνές σύστημα ρύθμισης του παγκοσμίου εμπορίου και πιο συγκεκριμένα του ΠΟΕ γιατί με την σημερινή κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών δεν μπορώ να περιμένω κάτι καλύτερο. Η περίπτωση της Μπομπάρντια είναι μια εξαιρετικό παράδειγμα για το τι εννοώ όταν λέω να αποφύγουμε τις περισσότερες ζημιές. Όταν ουσιαστικά είχαμε την Boeing να προσπαθεί να εισέλθει σε μια ε, εγχώρια αγορά. Να προστατεύσει μάλλον με, ε, την εγχώρια αγορά με ουσιαστικά προστατευτικά μέτρα. Και η Αμερικανική κυβέρνηση ουσιαστικά απείλησε ότι θα προκαλέσει ζημίες στην Μπομπάρντια για να ε, μην ε, ανταγωνιστεί η Μπομπάρντια την Boeing. Όμως υπάρχουν παραγγελίες για 4.000 αεροπλάνα ε, της Μπομπάρντια προς τη Δέλτα και το οποίο θα παραδοθούν μετά το 2020. Υπό αυτή την έννοια δεν φαίνεται ότι είχε μια άμεση ζημία η εταιρεία η ευρωπαϊκή αυτή. Αυτό που θα ήθελα να ακούσω όμως πιο κάθαρα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι τι σκοπεύει να κάνει για έναντι της Boeing η οποία προσπαθεί να αξιοποιήσει, να προστατεύσει τη θέση της στην αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών και να αποτρέψει τη Bombardier από το να εισέλθει σε αυτήν. Τι θα συμβεί αν αρχίσουν να επιβάλλονται ε, τέλη, δασμοί. Δεδομένων και των παλαιότερων ε, παραδειγμάτων που έχουμε προστατευτικών μέτρων όπως τον τομέα του Χάλιβα πρέπει να ίσως να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε το ενδεχόμενο ε, αντιπίνων ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν έχει νόημα να περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει τελικά ε, ο πρόεδρος Τραμπ, από ό,τι φαίνεται μόνο το, τη δύναμη του ισχυρού αντιλαμβάνεται. Βεβαίως και γνωρίζω ότι δεν είμαστε υπέρ του προστατευτισμού και τέτοιου τύπου μέτρων εδώ. Όμως, εάν οι ε, Ηνωμένε Πολιτείε ξεκινήσουν να προσπαθήσουν σαν οδοστρωτήρε να περάσουν πάνω από πολλέ άλλε χώρε, θα πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε εμεί και τι σκοπεύει να κάνει η Ευρωπαϊκή ε, η Επιτροπή για να το σταματήσει αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Θα συγχαρώ τον Ντέιβιντ, αλλά πρώτα πρέπει να σας πω ότι υπάρχει αντιπροσωπεία της Μπομπάρντια από τη Βόρεια Ιρλανδία στο Κοινοβούλιο και είναι κρίμα ε, που η ίδια μου η ε, κυβέρνηση ε, δεν έκανε τα, αυτά που έπρεπε αντί δηλαδή να, να βγουν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι η ίδια η εταιρεία για να προστατεύσει τον εαυτό της και όχι το αρμόδιο Υπουργείο ε, και ε, το αρμόδιο αρμόδιος υπουργός από, από το Ηνωμένο Βασίλειο. Εν πάση περιπτώσει, ε, ρωτήθηκε τι έχει κάνει το Ηνωμένο Βασίλειο. Το ρωτήσαμε εμείς τι έχει κάνει το Ηνωμένο Βασίλειο μέσω επιστολής ε, για την Μπορμπάρντια, αλλά δεν ε, λάβαμε απάντηση. Ποιες είναι οι διασυνδέσεις ε, που ενδεχομένως υπήρξαν μεταξύ της κυβερνήσεως του Ηνωμένου Βασιλείου και των υπηρεσιών της Κομισιόν όσον αφορά την περίπτωση τη Μπομπάρντια. Έχουμε τις ελιές της Ισπανίας, έχουμε το ελαιόλαδο, έχουμε τον χάλιβα. Πολλές περιπτώσεις ε, όπου πραγματικά αντιμετωπίστηκαν πάρα πολλά ε, προβλήματα ε, και ε, ε, του χρόνου θα έχουμε και τις αποφάσεις ε, για την Airbus και την Boeing. Στην ουσία αυτό που μας δείχνει η υπόθεση της Bombardier είναι ότι εταιρείε οι οποίες έχουν και εκτιμένα συμφέροντα στην αγορά της, των Ηνωμένων Πολιτειών υπό την διακυβέρνηση Τραμπ πιέζονται πάρα πολύ. Νομίζω ότι ο Τραμπ ως επιχειρηματίας καταλαβαίνει πότε ε, υπάρχει ένα κοινό μέτωπο ή πότε αντιθέτως δεν υπάρχει ε, συνένεση και νομίζω ότι ε, όταν οποτεδήποτε εμείς έχουμε κινηθεί όπως το 2003 ή το 2002 όταν είχαμε ενωτικό μέτωπο όσον αφορά ας πούμε μεταποιημένα προϊόντα λοιπά ήταν τότε η διακυβέρνηση Bush τότε ε, ε, ε, μπορέσαμε να κερδίσουμε. Βεβαίω τότε στο Ηνωμένο Βασίλειο υπήρχε και μια κυβέρνηση η οποία έχει ιδιαίτερε σχέσει με, το, με τι Ηνωμένε Πολιτείε και εν πάση περιπτώσει μονάχα όταν απειλήθηκαν συγκεκριμένα μέτρα όσον αφορά δασμού για γεωργικά προϊόντα, πορτοκάλια κλπ. καταφέραμε να ξεπεράσουμε το πρόβλημα ότι εδώ δεν χρειάζεται να ξεκινήσουμε έναν ε, τρομερό εμπορικό πόλεμο, αλλά θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Ε, πρέπει να ξέρουμε λοιπόν και ποια είναι τα σχέδια της ε, Κομισιόν. Έχουμε μερικές φορές την αίσθηση ότι ε, τελικά ε, ε, προσπαθούμε να φερθούμε στη διακυβέρνηση Τραμπ όπως κάνουμε με τον θείο που έχει μεθύσει στη γιορτή των Χριστουγέννων, τον βάζουμε σε μια ακρούλα εκεί πέρα και λέμε δεν βαριέσαι ο καημένος, θα του περάσει το μεθύσι. Δεν είναι έτσι όμως, γιατί εδώ διακυβεύονται πολλές χιλιάδες ε, ε, θέσεις εργασίας και στον Belfast έχω να σας πω ότι αυτό μας καίει πάρα πολύ. Ναι, αυτό είναι μια πολύ ωραία εικόνα, λέει ο Πρόεδρο για το που ίσως θα έπρεπε πραγματικά να βρει θέση ο Τραμπ, αλλά εν πάση περιπτώσει. Ο κύριο Χούμπερτ, από την Κομισιόν. Σας ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι που ξανά είμαι σήμερα εδώ. Σε γενικέ γραμμέ, κύριε Πρόεδρε, και σε μεγάλο ποσοστό νομίζω ότι μπορώ να ενστερνιστώ τα σχόλια που κάνατε στι αγωγέ σα παρατηρήσει και ίσω να σα πω και δύο λόγια σχετικά με την δική μα αξιολόγηση τη εργασία τη καθημερινή και επαφή που έχουμε με του ε, ε, Αμερικανού ε, εταίρου. Δύο χρόνια περίπου έχουν περάσει από την εκλογή Τραμπ και ένα χρόνο, συγγνώμη, έχει περάσει <laughs> από την ε, ε, εκλογή του κυρίου Τραμπ και έχουμε ε, κάνει πολλές συζητήσεις για πολλά θέματα ε, και υπάρχουν και τέτοιες αποφάσεις οι οποίες δεν έχουν ακόμα ε, θέσεις μάλλον ε, σχετικά με το εμπόριο υπουργών, υφυπουργών κλπ. που δεν έχουν ακόμα περάσει και επικυρωθεί από την Γερουσία. Επομένως θα πρέπει να δούμε ποιες είναι οι προτεραιότητες των Ηνωμένων Πολιτειών. Σε τούτη την συγκεκριμένη περίπτωση νομίζω ότι θα πρέπει να ξεκινήσουμε να μελετούμε τα θέματα από, των Ηνωμένων, από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών γιατί οπωσδήποτε ε, η έκβαση των ε, εκλογών ε, είχε επίπτωση στην εμπορική πολιτική. για να μην αναφέρω και τα όσα σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή και τις διεθνείς σχέσεις. Πέρα από αυτό όμως, ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί η ε, διαμόρφωση πολιτικής γιατί ε, ξέρετε ότι πάντα υπάρχουν διαφορές ανάμεσα ε, στους ρεπουμπλεκανούς στην κυβέρνηση. Ξέρετε ότι ότι η διαδικασία διατησίας είναι αυτή η οποία δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί γιατί ε, το Κογκρέσο έχει ισχυρές ε, ενστάσεις και ε, έχει μάλλον δύναμη όσον αφορά τη διαμόρφωση της εμπορικής πολιτικής. Όσον αφορά τώρα τομιακέ διαφωνίες Ξέρετε ότι υπάρχει μία έρευνα για ε, για το αλουμίνιο και για τον χάλιβα από πλευράς ε, της Υπηρεσίας Εθνικής Ασφάλειας ε, και που σχετίζεται και με την πολιτική των προμηθειών στις Ηνωμένε Πολιτείες. Επίσης, στην ίδια την ουσία των διαπραγματεύσεων ναύτα έχει προωθηθεί και το θέμα ε, των ελιών και του ελαιολάδου γιατί ε, και εδώ έχουμε είχαμε ένα γύρο πριν από τρεις-τέσσερις εβδομάδες ε, και όλες οι προτάσεις πλέον έχουν υποβληθεί. Δεν έχουμε όμως πρόσβαση στις προτάσεις αυτές, αλλά ξέρουμε πάνω κάτω ποια είναι η εστίασή τους. και υπάρχουν και 5-6 ε, κύριες, ε, ε, κύρια πεδία εντός της ναύτα και εκεί μπορεί κανείς να δει ποια είναι η πραγματική και τι σημαίνει πραγματικά για, το, για την εμπορική πολιτική η πολιτική ε, Τραμπ και όσον αφορά της προμήθειας και όσον αφορά ε, την, ε, το, το λεγόμενο κεφάλαιο 19 και όσον αφορά την γενική επίλυση διαφορών για το κεφάλαιο 19 είναι για τις εμπορικές ε, επίσης όσον αφορά την ρήτρα sunset για το εμπόριο. Αυτές όλες είναι προτάσεις ε, τις οποίες έχει ε, υποβάλει στον Καναδά και στο Μεξικό ε, η διακυβέρνηση Τραμπ. εξ όσων γνωρίζουμε και από τους Μεξικανούς και Καναδούς φίλους. Όλες αυτές οι διαπραγματεύσεις είναι ευρέως γνωστό ότι είναι δύσκολες. Ε, και οι αποφάσεις έχουν μετατεθεί για το πρώτο τετράμινο, τρίμηνο μάλλον, του επόμενου έτους, το 2018. Και η άλλη προτεραιότητα των ΗΠΑ, από ό,τι φαίνεται, ε, αφορά τις σχέσεις με την Κινία, την Κίνα. Ε, Φαίνεται ότι ο Υπουργό Εμπορίου είναι ο μόνο ο οποίο ε, συνοδεύει τον ε, κύριο Τραμπ σε αυτήν την ε, περιοδία που κάνει στην Ασία. Είναι αυτό ο οποίο είναι και σύμβουλο υπεύθυνο για τα θέματα τη Κίνα. Μα ενδιαφέρει επίση και η συνέχεια που θα δοθεί στην πρώτη έρευνα για την Huawei που ξεκίνησε τον Αύγουστο στι Ηνωμένε Πολιτείε η πρώτη ε, αναφορά ε, βρίσκεται σε, ακόμα σε φάση ε, σύνταξης. Πιστεύω ότι αυτές οι δύο σχέσεις είναι οι πιο σημαντικές για τον Τραμπ. Απ' τη μία η ναύτα και οι σχέσεις εντός της ναύτα για θέματα τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά και διαπραγματεύσεις οι οποίες είναι ιδιαίτερα κρίσιμες Ε, και αυτό μας ε, ε, οδηγεί στο ερώτημα πού θα φτάσουν οι διαδικασίες αυτές βάση και του αμερικανικού πολιτικού συστήματος, του βάρους που έχει το Κογκρέσο κλπ και εσείς βεβαίως ως Κοινοβούλιο φαντάζομαι ότι ενδιαφέρεστε ε, στην κατανόηση ε, της δυσκολίας διαιτησίας που ε, από αυτή τη διαδικασία μπορεί να προκύπτουν. Το δεύτερο σκέλος είναι οι σχέσεις ΗΠΑ με την Κίνα υπό το φως των ερευνών που έχουν ξεκινήσει. instruments that you don't use very often. It's been sort of polished again and brushed up. And potentially it can lead to good outcomes if they are market opening outcomes. It can lead to... Εν πάση περιπτώσει θα πρέπει οπωσδήποτε να τα δούμε όλα αυτά συνολικά και εντός του Διεθνούς Οργανισμού Εμπορίου πράγμα όχι εύκολο. και ε, εν πάση περιπτώσει ε, δεν μπορούμε να λησμονήσουμε ότι οι σχέσεις με την Κίνα είναι πάρα πολύ σημαντικές για τις ΗΠΑ. Ε, υπάρχουν προβλήματα, υπάρχουν σύννεφα στην σχέση αυτή, το ανέφερα και προηγουμένως και αυτό θα έχει ιδιαίτερο βάρος στις εμπορικές αποφάσεις της Κίνας και τη συζήτηση επί των εμπορικών αυτών αποφάσεων. Εμείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση ε, ενδιαφερόμαστε για τα δικά μας συμφέροντα. Έχουμε ε, τα ζητήματα που σχετίζονται με το Διεθνή Οργανισμό Εμπορίου, έχουμε τα ζητήματα που σχετίζονται με το Apple Buy, έχουμε και αν μου επιτρέπετε μάλλον να απαντήσω σύντομα στις ερωτήσεις ε, που, υπέλαβε, ε, ε, ε, υπέβαλαν οι δύο συνάδελφοί σας για το Bombardier. Εμείς βεβαίως συνεργαζόμαστε με τις αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου για αυτές τις έρευνες, καθώς επίσης και με τις καναδικές αρχές, αλλά δεν έχουν ακόμα ληφθεί μέτρα. Θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι τα μέτρα τα οποία θα ανακοινωθούν αλλά μην ξεχνάτε ότι εμείς πρέπει να είμαστε, οφείλουμε να είμαστε οι θεματοφύλακες ε, της διαδικασίας. Ποια είναι τα μέτρα τα οποία θα χρησιμοποιηθούν ε, και εν πάση περιπτώσει οτιδήποτε αποφασιστεί να είναι απολύτως ε, συμμορφωμένο με τις διαδικασίες και συμφωνίες αντι-dumping καθώς επίσης και με τις διαδικασίες και συμφωνίες επί των επιδοτήσεων. Πολλές εξελίξεις ε, θα υπάρξουν και σε επίπεδο ε, επιχείρησης γιατί οπωσδήποτε δεν πρέπει να δούμε αυτά τα εμπορικά μέτρα ε, από μόνα τους και σε κενό αέρος. Τώρα, ποια θα είναι τα ενδεχόμενα μέτρα που σε των ΗΠΑ δεν μπορώ να το πω αλλά ε, αυτό που μπορώ να πω είναι ότι μας ενδιαφέρει ιδιαιτέρως ε, και πραγματικά με μεγάλη προσοχή παρακολουθούμε και το ενδιαφέρον της Βόρειας Ιρλανδίας για το θέμα αυτό και ευχαριστούμε πολύ που το θίξατε. Ευχαριστούμε πολύ. Δεν θα πω πολλά λόγια γιατί σίγουρα πολλά ακόμη θα τα συζητήσουμε εντατικά, όμως το θέμα το οποίο ε, ετέθη κατά πόσον εμείς θα πρέπει να αντιδράσουμε πιο έντονα σε ό,τι αφορά αυτήν την αναμονή μας για τους ε, δασμούς που είναι τόσα χρόνια ε, σε ίσχυ για συγκεκριμένους τόπους ή το θέμα με το κράσι και τις ορμόνες ε, ή το άρθρο 232 εγώ πιστεύω ότι πράγματι πρέπει να σκεφτούμε πάρα πολύ σοβαρά πώς θα αντιδράσουμε. Πώς, ε, αν θέλετε, να οξύνουμε ε, τα όπλα μας. Λοιπόν, ας ε, ολοκληρώσουμε εδώ με αυτό το σημείο και πλέον βάζω το καπέλο όχι του συντακτονόματος αλλά του Προέδρου. Να σας πω το χρονοδιάγραμμα μετά το συνεισμό με την ΑΦΕΤ. Θα σας δώσουμε τα σχετικά, δεν έχουμε ακόμη ε, συγκεκριμένα χρονοδιάγραμμα. Any other business, το αγαπημένο μου σημείο. Δεν υπάρχουν διάφορα, ελπίζω. Και το επόμενο σημείο είναι η επόμενη συνεδρίαση. 22 και 23 Νοεμβρίου θα ξανασυνεδριάσουμε. Αυτά και μένω. Καλό Σαββατοκύριακο.